Meine Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, zur Tagesordnung. Έχετε παρατηρήσει για τη μέση διάταξη, όχι από ό,τι βλέπω. Ούτε και ο πρόεδρο δεν έχει καμία ανακοίνωση να σα κάνει. Μερικές παρατηρήσει μόνο. Για το ταξίδι της μιας αντιπροσωπείας της Επιτροπής μας στην Ιορδανία, στην αρχή και μετά στο Λίβανο την περασμένη εβδομάδα. Βλέπω ότι παρεμβρίσκεται η κυρία Άννα Γκόμες. Και η κυρία Μανέσκου, κύριος Γιούρεκ, η πλειονότητα των μελών της ε, αντιπροσωπείας αυτής παρεμβρίσκεται. Λοιπόν, σύντομα, θα μπορέσουν να με υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν ε, ότι έχω ξεχάσει. Άλλοι συμμετέχοντες ήταν ο κύριος Καν, Χαν από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ε, είχαμε πολύ καλά προγράμματα. Ε, Δήμερη ήταν η επίσκεψη, μια μέρα στο Αμάν και μια μέρα στο Λίβανο και στις δύο χώρες. Μιλήσαμε με των Ηνωμένων και του Γραφείου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια έχω για την κατάσταση των προσφύγων και στις δύο χώρες είναι πολύ μεγάλη η επιβάρυνση, αποσταθεροποιητική θα έλεγα, για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά. Στο Λίβανο σήμερα, αν μετρήσουμε και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, σε μια χώρα που έχει 4 εκατομμύρια κατοίκου και είναι κατακαιρματισμένη πολιτικά, 1,3 εκατομμύρια με 1,5 εκατομμύριο είναι πρόσφυγε. Καταλαβαίνετε, από 4 εκατομμύρια κατοίκου συνολικά, 1,5 εκατομμύριο σχεδόν είναι οι πρόσφυγε. Και ε, είναι απλή αριθμητική αυτή. Και υπολογίζω ε, ε, και πόσους θα έπρεπε να έχουμε στη Γερμανία αν είχαμε αντίστοιχο ποσοστό στο Λίβανο δεν είναι σε καταβλισμούς αυτοί οι πρόσφυγε. Λέει ο Λίβανο, βέβαια ότι πριν από 60-70 χρόνια το είχαμε ξαναζήσει αυτό με του Παλαιστίνιου και παραμένουν οι καταβλισμοί είναι εκεί. Και από αυτή την εμπειρία λοιπόν διδάχθηκαν και τώρα ε, είναι μοιρασμένοι σε όλη τη χώρα, μένουν ε, ε, σε σπίτια κανονικά ιδιωτών που αυτό ενέχει και πιέσεις και κόστος. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση ούτε για τον πληθυσμό ούτε για τους πρόσφυγες τους ίδιους στον ίδιο το Λίβαν, μάλλον το πόλιο στην Ιορδανία, είναι κλασική καταβλισμή προσφύγων. Συχνά πολύ κοντά στα Συριακά σύνορα και έχουμε κλασικές καταστάσεις σε καταβλισμούς γύρω στο 1 εκατομμύριο επισήμως είναι 700.000 ή 1,3 Τώρα πώς να τους μετρήσεις κιόλας δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αλλά έτσι κι αλλιώς 60% του πληθυσμού της Ιορδανίας είναι Παλαιστίνοι ουσιαστικά. Και αν το προσθέσουμε αυτό, ε, έχει κάποια προβλήματα για τη σταθερότητα του οίκου των ε, χασεμιτών ε, που βασιλεύουν στη χώρα αυτή. Λοιπόν, έχουμε την ιστορία με το Ιράκ και τη Συρία και δεν μπορούν αυτές οι δύο χώρες να αποσταθεροποιηθούν, ο Λίβανος και η Συρία δηλαδή έτσι Επόμενο θέμα. Η Ορδανία, από ό,τι φαίνεται, είναι αποφασισμένη ε, μετά και ε, την ε, το θάνατο το τραγικό του κυβερνή, του χειριστή του αεροσκάφους που τον έκαψαν ζωντανό είναι αποφασισμένη να πατάξει αυτή την κατάσταση και είχα πάει και στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ, στο Ιράκ και αν δεν καταφέρει η Βαγδάτη να βρει μια άκρη ανάμεσα σε μετριοπαθείς Άραβες, Σουνίτες και Σιήτες και υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι δεν πρόκειται να το καταφέρουν γιατί επί Μαλίκη χάθηκε πάρα πολύ εμπιστοσύνη και είναι πάρα πολύ καχύποπτη. Λοιπόν, αν δεν συμβεί αυτό, μπορεί οι Ορδανοί να μεσολαβήσουν με τις επαφές τους στο Ιράκ και τη Συρία ε, προς φυλές σουνητικές μετριοπαθείς για να γίνουν κάποιες συνεννοήσεις και ε, σε στρατικό επίπεδο, για να το πω έτσι κάπως μαλακά. Αυτά είναι τα στρατηγικά ε, συμπεράσματα, τα υπόλοιπα δεν είναι τίποτα τραγικά νέα πολύ διαφορετικά. Θέλω να τονίσω ότι και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και στο Ιράκ και στο Ιρακινό Κουρδιστάν και στη Συρία, το θέμα των μειονοτήτων έχει τεράστια σημασία. Μειονότητες, χριστιανικές, γιζιδοί και άλλες εθνικές μειονότητες, αλεβίτες, Κούρδοι και στη Συρία ας πούμε και λοιπά. Είναι ένα συνοθήλευμα εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε στο Λίβανο, ότι είναι διαφορετικές οι απόψεις. Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που λέγουν ότι θα πρέπει να ε, συνεργαστούμε με τον Ασάτ για την καταπολέμηση του ISIS, του Ισλαμικού κράτους, ενώ κάποιοι άλλοι λέγουν ότι, ε, ενώ αντιμετωπίζουμε το ISIS θα πρέπει να είμαστε και κατά του Ασάντ. Αυτή πάνω κάτω είναι και η τουρκική θέση για τους γνωστούς λόγους. Η Τουρκία είναι σημαντικός παράγον στην περιοχή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις εμείς λέγαμε ότι η λύση δεν θα πρέπει να είναι κάτι που θα αναμένεται από την Ευρώπη κατά πρώτο λόγο. Έχει σημασία τα Ισλαμικά κράτη της περιοχής και τα Αραβικά δηλαδή αραβικά συν Τουρκία συν Ιράν, να καθίσουν, να συνεργαστούν για να βρουν μια λύση για τη δική τους περιοχή και ο καθένα να αναλάβει τις ευθύνες τους. Αυτοί μεταξύ τους σακώνονται, κάνουν πολέμους για αντιπροσώπων από το Ιράκ μέχρι το Λίβανο. Είναι proxy wars, είναι πόλεμοι δια αντιπροσώπου που ε, προέρχονται από τη σύγκριση Ιράν-Σαουδικής Αραβίας και ε, οι Σουνίτες, οι διάφοροι χριστιανοί στο Λίβανο και οι Σιήτες, ο καθένας έχει στην ε, Ριάντη ή στην Τεχεράνη άλλο ως σημείο αναφοράς. Και αυτός από τη Τεχεράνη μετά πάει στη Δαμασκό. Καταλαβαίνετε ότι για να σπάσουν αυτοί οι πόλεμα διατή προσώπων θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρξει μια λειτουργική ενότητα επιχειρησιακή. Καλό είναι που έχουμε αυτή τη συμμαχία των 60 χωρών. Αλλά για να είσαι επιχειρησιακό θα πρέπει και λειτουργικό να έχουν όλοι οι γείτονε την ίδια στρατηγική. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο κανονικά θα ήταν ε, ευρωπαϊκή πολιτική. Να επικεντρωθούμε σε αυτό. Μεταξύ των 60 κάπου να ε, υπάρξει μια πιο μικρή ομάδα λειτουργική επιχειρησιακή και αυτό έχει σημασία πολύ περισσότερο από ότι να συνεχίσουμε τις παραδόσεις όπλων ή να στείλουμε εκεί χερσαίες δυνάμεις. Και είναι και πίεση για να τα βρούνε κάπου ο Ισλαμικός κόσμος να ενωθεί προς τη σωστή κατεύθυνση και για καλό σκοπό. Μεγάλες τώρα ανησυχίε, το λέω και δημόσια στη συνεδρίαση, μας προκάλεσε μάλλον μας εξέφρασαν παντού ε, άτυπα ως προς την πολιτική της Τουρκίας. Ανησυχούν πάρα πολύ για την πολιτική της Τουρκίας διότι δεν γνωρίζουν τελικά πού το πάει η Τουρκία. Επίσης εδώ έρχεται να προσθεθεί και το θέμα της Λιβύης. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Διότι η υποστήριξη των ε, ακεροφρόνων, των φουνταμενταλιστών στη Λιβύη, από την Τουρκία είναι ένα ζήτημα και πολύ αποσταθεροποιητικό. Και η Αίγυπτος που ανέκαθεν ήταν σταθεροποιητικός παράγων έχει βρεθεί τώρα μεταξύ δύο πυρών. Και έχουν κάνει και δράσεις. Είχαν μια αεροπορική επιχείρηση η Αίγυπτη ε, μετά από την εκτέλεση των 21 σκοπτών χριστιανών στη Λιβύη. Όλα αυτά είναι ενισχυτικά και Ξέρουμε ότι ο καθένα στην περιοχή έχει τη βλέψη, τις βλέψεις του και τις φιλοδοξίες του μπορεί να έχει προσωπικά ο κάθε ηγέτης, αλλά το θέμα είναι να αντιμετωπίσουμε ε, αυτό το θέμα του Ισλαμικού κράτους με όλα τα πλοκάμια και τις διακλαδώσεις από την Ιγυρία μέχρι το Πακιστάν. Δηλαδή είναι μια τεράστια υπόθεση αυτή και έχει και ε, διασυνοριακές ε, επιπτώσεις και προεκτάσεις πέρα από τη Ιρία και το Ιράκ. Φυσικά ε, περισσότερη βοήθεια για τους πρόσφυγες και τα λοιπά. Μας τα είπανε, δεν χρειάζεται να το τονίσω κι εγώ εδώ. Αν έχετε πάει σε καταβλισμό τέτοιο προσφύγων ή έχετε δει πώς καταχωρίζονται εκεί οι οικογένειες με πάρα πολλά μικρά παιδιά. Δεν χρειάζεται και δικαιολόγηση περισσότερη αυτό το θέμα. Πέρα από τα πολιτικά και τα οικονομικά λοιπόν κυριαρχεί αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα παντού. Α, και ένα τελευταίο. Στο Ερμπίλ κοντά, σε ένα καταβλισμό, μου είπε μία Γερμανίδα νεαρή που δουλεύει στον Ερυθρό Σταυρό ότι ε, η Ευρώπη δίνει τόσα λεφτά, οι Γιατί δεν προβάλλεται αυτό που πουθενά, γιατί δεν υπάρχει καμία ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πολλούς τομείς δίνουμε και 50 και 60 και 70% των πόρων, αλλά οι άνθρωποι επιτόπου δεν το βλέπουν ότι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί μπαίνουν όλα ε, υπό τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών, που δεν με πειράζει αυτό, αλλά κάπου να φαίνεται και η Ευρώπη εκτός από τα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί και αυτό είναι ένα μήνυμα. Ο κόσμος εκπλήσεται όταν ακούει ε, ποια ποσά δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πολλοί πολιτικοί θύνονται εκεί πέρα δεν τα γνωρίζουν αυτά. Και αυτό θα πρέπει να είναι ένα τμήμα της πολιτικής, να τα λέμε και να τα επισημαίνουμε και να φτάνουμε μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Θέλει κανεί το λόγο, κύριε Μανέσκου. Mulțumesc, domnule președinte. Ați uh, rezumat foarte bine uh, discuțiile pe care... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνοψίσατε τις συζητήσει που έλαβαν χώρα κατά την επίσκεψή μας στην Ιορδανία και στο Λίβανο. Απλώς θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Ναι, η Ορδανία και ο Λιβανός δείχνουν προθυμία να πολεμήσουν την τρομοκρατία, δείχνουν αφενός ότι είναι αποφασισμένες οι χώρες αυτές, αλλά από την ΑΕΛΗ χρειάζονται και στήριξη και στρατιωτική αλλά και οικονομική. τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δηλώσει ότι θα δοθεί η στήριξη αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω ότι και οι δύο κυβερνήσεις είπαν ότι ανησυχούν πάρα πολύ για την επιρροή του Ιράν στην περιοχή και την ε, απειλή που θέτουν οι Ιρανικές πολιτικές στην περιοχή. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Θα πρέπει αυτά να μην τα ξεχνάμε όταν ε, θα εξετάζουμε το θέμα των διαπραγματεύσεων ε, με το Ιράν. Και σε ό,τι αφορά την κατάσταση των προσφύγων στο Λίβανο, υπάρχουν ε, δύο οπτικές στο Λίβανο και αυτό είναι επίσης κάτι άλλο που πρέπει να έχουμε κατά νου. Θα πρέπει να παράσχουμε στήριξη για το μελλοντικό κίνημα και τους συμμάχους του στο Λίβανο που θέλουν να ακολουθήσουν ένα παρόμοιο μοντέλο με το παράδειγμα της Ιορδανίας ό,τι αφορά ε, τους καταβλισμούς των προσφύγων ε, γιατί είναι εύκολο να διαχειριστούν αυτούς τους καταβλισμούς. Από την αρχή ήταν κατά της δημιουργίας αυτών των καταβλισμών αν και είδαμε επιτόπου στην Ιορδανία και γνωρίζουμε ότι αυτοί οι καταβλισμοί καθιστούν πιο διαχειρίσιμο το ζήτημα των προσφύγων επιτόπου. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Στο Λιβανό Υπάρχει ένα μέρος ε, των πολιτικών που υποστηρίζει τη δημιουργία αυτών των καταβλισμών. Έτσι λοιπόν και εμείς θα πρέπει να προσφέρουμε την υποστήριξή μας προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πείσουμε τη Χεσμολά και τους ε, συμμαχούς της ότι είναι χρήσιμο να δημιουργούνται στρατόπεδα συγκέντρωσης, ένα σύστημα της συγκέντρωσης και ότι αυτό θα πρέπει να γίνει γιατί διαφορετικά ναι μπορούμε να δώσουμε οικονομική βοήθεια όμως, ε, αν είναι διασκορπισμένοι οι πρόσφυγες, όλη την επικράτη είναι πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση. Και επίσης είναι και πάρα πολύ δύσκολο για όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να το διαχειριστούν αυτό. Η γενική εντύπωση ήταν ότι ναι, υπάρχουν κάποιοι κύριοι παίκτες στην περιοχή, φυσικά το Ιράν, μια χώρα που δημιουργεί αστάθεια και θα μπορούσε να θέσει ενδυνάμει ένα κίνδυνο λόγω των πολιτικών ακολουθεί, αλλά έχουμε και την Τουρκία και την Αίγυπτο. Αυτοί θα έπρεπε να εμπλακούν περισσότερο και θα πρέπει να τους παράχουμε υποστήριξη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συμφωνώ με την περίληψη που κάνατε. Απλώς θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ κάποια θέματα. Όπως είπατε, πολλοί από τους συνομιλητές μας ε, τόνισαν το 100η ζήτημα, θεώρησαν ότι είναι κεντρικό θέμα στη σύραξη και μάλιστα μας είπαν ότι τη σύραξη αυτή δεν ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με στρατιωτικά μέσα χρειάζεται ένας ε, μακροπρόθεσμος ε, ιδεολογικός ε, αγώνας γιατί πρέπει να δούμε και ότι πάρα πολλοί άνθρωποι από όλη την περιοχή αλλά και από την Ευρώπη ελκύονται από αυτή την ιδεολογία και επιλέγουν τις διαστράσεις. Εγώ Θεώρησα ότι είναι ενισχυτικό το εξή, ότι παρά τι τεράστιε προσπάθειε ε, που γίνονται από την υποτερμαστία του ΙΕ ε, για του πρόσφυγε και από εμά, που είπατε, υποστηρίζουμε και πληρώνουμε ε, για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των διεθνών προσπαθειών, εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλοί λόγοι ανησυχία και παρά το ότι ο Λίβανος και η Ορδανία καταβαλούν τεράστιες προσπάθειες ε, για να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες. Ε, όπως είπατε, το 1 τέταρτο του πληθυσμού αυτή τη στιγμή στο είναι πρόσφυγες. Εγώ θεώρησα ότι είναι πολύ σχετικό το ότι μας είπαν ότι, για παράδειγμα, στο Λίβανο από 385 παιδιά που... Ε, παιδιά που είναι σε ηλικία σχολείου 300.000 ε, δεν φοιτούν στο σχολείο. Ε, δεν φοιτούν λοιπόν στο σχολείο, δεν θα μπορούν να νοικοδομήσουν τη Συρία μια μέρα. Και σε κάποια χρόνια θα είναι βορρά ε, για στρατολόγηση από τους ε, τρομοκράτες. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό λοιπόν και φυσικά δεν διευκολύνει το γεγονός ότι στο Λιβάνο δεν υπάρχουν καταβλισμοί, το ότι υπάρχουν καταβλισμοί στην Ιορδανία είναι πιο εύκολο για να δοθεί βοήθεια. Όμως ε, για την ε, Ιορδανία είδαμε ότι και είναι δυσάρεστο ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν ε, και να είμαστε ξεκάθαροι, δεν θα επαντρέψουν οι άνθρωποι στη Συρία όσοι είναι εκεί ο Ασάντ, δεν θα το κάνουν αυτό και φυσικά τώρα υπάρχει και μία αίσθηση στο Λίβανο ότι υπάρχουν και μία προσπάθεια να τους ξαναστείλουν πίσω στη Συρία, οπότε αυτό ότι θα είναι εισφαλής και οι άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε και αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια. Όμως εγώ δεν νομίζω ότι ο ΣΑΝΤ αποτελεί τμήμα της λύσης, αλλά είναι μέρος του προβλήματος, ακριβώς γιατί δεν θα επιστρέψουν ποτέ οι πρόσφυγες. Κάποιοι από εμά στην Ευρώπη πιστεύουν ότι μπορούμε να βασιστούμε τώρα στον ΣΑΝΤ για να είναι σύμμαχος για να καταπολεμηθούν οι τρομοκράτες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεχάσουμε τέτοιες ιδέες. Θέλω να τονίσω, όπως είπατε, ότι τώρα πράγματι βλέπουμε πολέμους δια προσώπων και ε, ήταν ε, η σύνταξη της Συρίας στη συνέχεια έγινε πόλεμος δια και μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Κατάρ. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος και φυσικά από την άλλη πλευρά έχουμε το Ιράν, έχουμε τον Ασάτ και φυσικά τη Ρωσία. Κάτι άλλο ιδιαίτερα ενοχλητικό για μένα ήταν ότι πολλοί από τους συνομιλητές μας και μέλη του Κοινοβουλίου και από την Ιορδανία και το Λίβανο μας είπαν ότι πίστευαν ότι η Δύση κατά κάποιο τρόπο ήταν πίσω από το Ισλαμικό κράτος. Πάρα πολύ ενοχλητικό αυτό, αλλά αυτό μας είπαν. Και γιατί. γιατί ε, ε, ε, είδαμε ότι είχαμε υποστηρίξει στους Σουνίτες με τις πολιτικές του Μαλική και αλλά και από το ρόλο που παίζει το Ισραήλ. Είναι κάπως περίεργος ο ρόλος του Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η αντίληψη πραγματικά ήταν ενισχυτική. Έκρουσε τον κοδύλο του κινδύνου για μένα, γιατί σίγουρα χρειαζόμαστε τέρου για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Αλλά αν δεν είναι απόλυτο πεπισμένοι, τι θα κάνουμε. Και είχαμε και άλλη μια συνάντηση. Υποτίθεται ότι έπρεπε να συναντήσουμε κάποιον από τη Σισβολάχ στο Κοινοβούλιο. Δεν μπορούσαμε να συναντηθούμε με αυτόν τον άνθρωπο γιατί δεν εμφανίστηκε αλλά έχω τη δυνατότητα να συναντήσω κάποιον από τη Χεσμολά και συνάντησα εκπροσώπους από την πολιτική πτέρυγα και νομίζω ότι και αυτά που έλεγαν ήταν ενδιαφέροντα, γιατί είχα την εντύπωση ότι η Χεσμολά από τη μια προσπαθεί να καταστήσει τον εαυτό της απαραίτητο ραχοκοκαλιά του Λιβανέζικου στρατού, και φυσικά αυτό έχει συνεπείς ε, και ότι τώρα έχουν κλείσει τώρα την μία πτέρυγα με τους χριστιανούς, αυτό λέει πάρα πολλά. Αλλά επίσης είχα την εντύπωση ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανησυχία για την ενότητα του Λιβάνου. Σε αντίθεση με άλλες δυνάμεις που λένε «Α, εν τέλει μπορεί να τσεκωνόμαστε, αλλά αν διακινδυνευτεί η ενότητα του Λιβάνου, θα υπερασπιστούμε την ενότητα του Λιβάνου. Δεν θα επιτρέψουμε στο Σολομόντα να κόψει το μόρο στα δύο. Και τέλος, για την δυνατότητα για την ε, συμφωνία με το Ιράν, θα ήταν σε κάπως δύσκολη θέση ένιωθαν ότι δεν επρόκειτο για τον Ασάντα, αλλά για τη στρατηγική σημασία της Συρίας. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται με τον πόλεμο διατυπροσώπων που ανέφερα νωρίτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γιουρέκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η επίσκεψη αυτή ήταν εξαιρετικά σημαντική και ευχαριστούμε πραγματικά τους ε, οικοδεσπότες μας και όσους ε, προετοίμασαν αυτή την επίσκεψη, την αποστολή. Είδαμε και εμείς ε, την κλίμακα της θεραπευτικής κρίσης, το μέγεθός της που έχει προκληθεί από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία. Μα έδωσε τροφή για σκέψη, καταφέραμε να συνεργάγουμε κάποια αποτελέσματα σχετικά με τι διάφορε αντιθέσει και συγκρούσεις στην ευρύτερη περιφέρεια και πώς μπορούν αυτές να έχουν ε, ανθρωπιστικές ε, επιπτώσεις και έτσι να επηρεάσουν τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων ε, ανθρώπων. Υπάρχει και ένα πιο πρακτικό ζήτημα το οποίο θα ήθελα να επισημάνω. Στο Λίβανο έχουμε τόσες διαφορετικές μειονότητες και θρησκευτικέ, μουσουλμάνους, χριστιανούς, σουνίτες και σιήτες αυτή η χώρα δεν λαμβάνει ιδιαίτερη αρρωγή όπως άλλες χώρες για να επιλύσει το ζήτημα των προσφύγων. Η Ορδανία είναι εξαιρετικά σημαντική χώρα για μας και θα πρέπει να το στηρίξουμε την επίλυση της ε, κρίσης με τους πρόσφυγες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να φανταστούμε καν στην Ευρώπη, το μέγεθος αυτής της κρίσης. Και ταυτόχρονα στο Λίβανο έχουμε 30% αυτή τη στιγμή το 1 τέταρτο δηλαδή του πληθυσμού, πρόσφυγες. Είναι πρόσφυγες το 1 τέταρτο του πληθυσμού. Χρειάζονται λοιπόν μεγαλύτερη βοήθεια. Τώρα, για την εσωτερική κρίση. Και κατά, πόσο αυτό αποτελεί λόγο να μην δώσουμε την απαραίτητη βοήθεια, αυτό για μένα δεν ευσταθεί ως επιχείρημα. Προφανώς, η διαδικασία του εκδημοκρατισμού είναι ε, πιο δύσκολη σε σχέση με άλλες μοναρχίες. Αν πούμε ότι είναι μια ε, χώρα ε, όπου υπάρχει που διέρχεται ένα μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά την εξουσία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει επιχείρημα κατά της περαιτέρω παροχής βοήθειας. Είναι κοινό μας συμφέρον. Όλοι αυτοί οι πρόσφυγες γιατί όλοι αυτοί οι πρόσφυγε, ακόμα και αν λήξει ο πόλεμο, δεν θα επιστρέψουν στη Συρία και στο Ιράκ κατά πάσα πιθανότητα, αλλά θέλουμε όσο δυνατόν περισσότεροι να επιστρέψουν στις χώρες τους, ούτως ώστε να μην ε, συμβάλλουν στην αποσταθεροποίηση, όπως είδαμε στη Λιβύη τη δεκαετία του 70. Και δεν θέλουμε περαιτέρω εισρωή προσφύγων, μεταναστών μάλλον, στην Ευρώπη. Γι' αυτό η στήριξη πρέπει να είναι πολύ σημαντική και αισθητή για να μπορούν να την αξιοποιήσουν οι χώρες όπως ε, ο Λίβανος. Ευχαριστώ. thank you, A uh, Πολλοί συνάδελφοι κάλυψαν ε, πολλά ζητήματα. Εγώ θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, το θέμα των προσφύγων. Τεράστια πίεση ασκούν οι πρόσφυγες στις γειτονικές τους χώρες ε, και στην Ιορδανία και στο Λίβανο και σίγουρα χρειάζονται επιπρόσθετη βοήθεια. Υπάρχει και το θέμα της εκπαίδευσης και το ανέφεραν διάφοροι συνάδελφοι. Νομίζω ότι έχουμε χάσει ήδη μία γενιά και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις περαιτέρω απώλειες. Και κάτι άλλο που με εκπλήττει είναι το εξής και οι δύο έχει να κάνει με τη δυνατότητα των προσφύγων να δουλέψουν. Οι δύο χώρες ουσιαστικά υιοθετούν τιμωρητικά μέτρα και δυσκολεύουν τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τα προσόντα τους. Τώρα, για το θέμα της Συρίας γενικότερα. Αυτό το οποίο διαφαίνεται σαφέστατα κατά τη γνώμη μου είναι ότι ο Ασάντ είναι πρόβλημα, είναι θέμα και έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Πολλοί το υποστηρίζουν. Ε, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα την παρουσία του Ασάντα. Πρέπει να δούμε και το ρόλο της Χεσμολάχ, η οποία τον βοηθάει. Θέτει σε κίνδυνο τη λεπτή ισορροπία που υπάρχει στο Λίβανο και γι' αυτό υπάρχει ο κίνδυνος να εξαπλωθεί η σύγκρουση και στο Λίβανο. Ε, και τίθεται και το θέμα του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας και του πολέμου αντιπροσώπων. Πρέπει να δούμε ποιος είναι ο ρόλος που μπορούμε εμείς να διαδραματίσουμε για να καταλαγιάσουμε τις υποψίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες όχι μόνο για το θέμα της Συρίας αλλά και για πολλές άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Υπάρχει αυτός ο πόλεμος δια το οποίο το μόνο που κάνει είναι να καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο ασταθή. Τώρα, ως προς το θέμα της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Κατάρ, τίθεται το εξής ερώτημα. Το κατά πόσο το Ιράν πρέπει να είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά. Ξέρετε, ε, έχει μακρά ιστορία στην περιφέρεια αυτή, στην περιοχή αυτή. Θα ήταν επικίνδυνο για εμάς να τους πρόξουμε προς την πλευρά του Ιράν με τρόπο κατά τον οποίο θα ενισχύσει το μήνυμα ότι δηλαδή ο πόλεμος πράγματι είναι εναντίον των μουσουλμάνων και του Ισλάμ. Ενώ εμείς θέλουμε ξεκάθαρα να στείλουμε το μήνυμα ότι ο πόλεμος δεν είναι εναντίον των μουσουλμάνων και του Ισλάμ. Τώρα το πώς θα διευκρινίσουμε αυτό το ζήτημα, το Χουάν, είναι πολύ σημαντικό. Και ε, τίθεται και το θέμα της, ε, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει στο Κοινοβούλιο, ωστόσο είναι κάτι που ε, αυξάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερο για να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Και όσα περισσότερα κάνουμε, τόσο πιο κοντά θα έρθουμε σε λύση και θα νικήσουμε το ΝΤΑΣ και την Αλκάιντα στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια παλιά γερμανική ε, παροιμία ε, που λέει ότι όποιος ταξιδεύει έχει πολλά να πει γιατί βλέπουν πολλά τα μάτια του ε, η οποία επιβεβαιώνεται σήμερα και το ακούσατε και από τους συναδέλφους ε, ο κύριος Βάγκελ ζητώ συγγνώμη που μακρηγορήσαμε αλλά είχαμε τους πολλά να πούμε ευχαριστώ λέει ο κύριος Βάγκελ θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω ότι είναι σημαντικό για εμάς να δείξουμε στήριξη σε δύο δημοκρατικές χώρες οι οποίες υποφέρουν από το πρόβλημα των προσφύγων και έχουν μακρά παράδοση αμφότερες αποδοχής, ανεκτικότητας, ανοίγματος αν θέλετε, είναι ανοιχτές τα προβλήματα των ανθρώπων από όπου και αν προέρχονται. Αυτή είναι η παράδοσή τους. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα μάθαμε και ακούσαμε πόσο προβληματική είναι η κατάσταση από την πλευρά της Ούνρα, η οποία ε, στην αρχή ασχολόταν μόνο με τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες και τώρα πρέπει να βοηθήσει για τη λύση ενός πολύ ευρύτερου προβλήματος. Ωστόσο, σε όλα τα λεχθέντα από τους άλλους συναδέλφους θα ήθελα και εγώ να προσθέσω το εξή και να το υπογραμμίσω. Σίγουρα ένας από τους πυρήνες του προβλήματος έχει να κάνει με τη σχέση μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραήλ, έχει να κάνει με την ευθύνη και των δύο μερών να βρουν λύση ε, στο ε, πρόβλημά τους. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξής κύριε Μπρόκ. Ποια φαίνεται η θέση της Ιορδανίας αυτή τη στιγμή έναντι του διαλόγου Ισραήλ-Παλαιστινίων, διότι ο μόνος παράγων στην περιοχή που κάποιες φορές ήταν δυνατόν να επικοινωνήσει και να γίνει αποδεκτός και από τα δύο μέρη, αυτός ήταν η Ιορδανία. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι η Ορδανία παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Με δεδομένο το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τον πόλεμο στη Συρία. Παρ' όλα αυτά με ενδιαφέρει η άποψή σας, τι ακούσατε, τι μάθατε από τους πολιτικούς της Ιορδανίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό να πω σύντομα μόνο ότι και στις δύο χώρες το θέμα του Ισραηλο-Παλαιστινιακού είναι κάτι που κυριαρχεί σε ημερήσια διάταξη και στην Ιορδανία παραμένει ζωντανή η πρόθεση και η διάθεση να μεσολαβήσουν για ειρηνική λύση. Αλλά και οι δύο χώρες γνωρίζουν και ξέρουν και το λέγουν ότι αυτή η σύγκρουση είναι άλοθη πάντα για ομάδες όπως είναι το Ισλαμικό κράτος. Ακόμα και αν υπάρξει ειρηνική λύση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, λύση δύο κρατών, αυτό όμως θα βοηθούσε ε, να ε, αφαιρέσουμε πολλά επιχειρήματα από τους ακραίους αυτούς που στρατολογούν ε, νέους την ακούσαμε αυτή τη θέση, δεν μπορώ παρά να την επαναλάβω και στη Ραμάλα και στη Βηρητό, επανειλημμένα. Τώρα, ο κύριος Μποστινάρου, παρακαλώ. Thank you very much, Mr. ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα στοιχεία που μας δώσατε και για το γεγονός ότι παρόλο που η Ευρώπη ξοδεύει πάρα πολλά χρήματα για να βοηθήσει τη χώρα και τους πρόσφυγες, θεωρείται η βοήθειά της μη αποτελεσματική ή είναι αόρατη. Και θα ήθελα να αναφέρω τη διάσταση της Λιβύης, γιατί το είπατε κι εσείς κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σημάνω το συναγερμό. Είναι επίγουσα η κατάσταση στη Λιβύη. Την περασμένη εβδομάδα 21 χριστιανοί αποκεφαλίστηκαν. Πέρα από το έγκλημα αυτό αυτό το οποίο είναι άνευ προηγουμένου, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι δραματικές εξελίξεις στη Λιβύη, οι οποίες ε, πολύ γρήγορα μια τοπική σύγκρουση θα τη μετατρέψουν σε περιφερειακή, η οποία πλέον μπορεί στη συνέχεια να ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Καλό λοιπόν όλους εσάς να συνεργαστείτε με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ο χρόνος τελειώνει. Τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρώπη, ως διεθνής κοινότητα για να ε, σταθεροποιήσουμε την κατάσταση και να υπάρξει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Γιατί ξέρετε η Λιβύη μπορεί να γίνει διάδρομος που να διασχίσει όλη την περιοχή και να συνδεθεί με την Μπόκο Χαράμ. Και ε, θα αποσταθεροποιηθεί ακόμα περισσότερο όλη η περιοχή, όλη αυτή η περιφέρεια και η κρίση θα λάβει πραγματικά εκρηκτικές διαστάσεις. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεργαστούμε με την Αίγυπτο και με άλλες τέτοιες χώρες για να υπάρχει μια ανάσχεση της κατάστασης και ε, να ε, παρεμποδίσουμε το Ισλαμικό κράτος έτσι ώστε να μην γίνει ε, πιο δραστήριο στην περιοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το πρόβλημα των προσφύγων είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως ε, είναι οι συνέπειες του προβλήματος. Ε, πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε να συνεχίζει να αυξάνεται το πρόβλημα και να έχουμε όλο ένα και περισσότερους πρόσφυγες, πράγμα που συμβαίνει γιατί δεν αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές και κοινωνικές ε, συνθήκες που δημιουργούν τους πολέμους αλλά και τους πρόσφυγες. Εγώ διαφωνώ όταν μιλάμε για προξηγούς, για πολέμους διαδιπροσώπων. Κανείς ε, δεν πεθαίνει επειδή του δίνουν εντολή κάποιοι ξένοι παράγοντες που καθορίζουν ότι κάποιος θα πρέπει να πολεμήσει το γείτονά του, ε, τον, ε, το διπλανό του στον Ιράκ, οι Σουνίτες και οι Κούρδοι και οι δεν πολέμησαν μεταξύ τους επειδή υπήρχαν διαβολικά συμφέροντα που τους έσπρωξαν, αλλά υπάρχουν ίδιες αντιφάσεις και αντιθέσεις στις χώρες αυτές. Ε, τώρα το να σκεφτόμαστε ότι ε, το Ιράν ή η συνωμοσία της Δύσης έχει προκαλέσει τον πόλεμο στη Συρία είναι ακραίο. Αυτό πρέπει να έχουμε όμως κατά νου, να έχουμε ένα πολιτικό κριτήριο και όχι ε, απλώς ένα υπερδιαστατικό κριτήριο και να σκεφτόμαστε ότι οι πόλεμοι αποτελούν συνέπεια εξωτερικών αποφάσεων ο κύριος Μπλοκ καλοφέρθηκε σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, την ε, Ισραηλοπανεστινιακή σύραξη. Δεν θα λυθεί η σύραξη αυτή αν ε, επιτρέψουμε να συνεχίζονται ε, οι συγκρούσεις εκεί παραβιάζοντας τις αποφάσεις του διεθνούς δικαίου. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν σειράξει στην περιοχή. Αυτό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε είναι να συνεχίζεται να παραβιάσει τη δυνατότητα των κρατών μέσω πρακτικών προσάρτησης και εκδίωξη των Παλαιστινίων γιατί ε, τελικά αυτό θα αποτελεί το τέλος και του ίδιου του κράτους του Ισραήλ. Εμείς ε, δεν μπορούμε να δεκτούμε τα τετελεσμένα. Και συμπερασματικά, ε, κάτι είπε ο συνάδελφος και είναι αλήθεια, η Ευρώπη θεωρείται ότι είναι πολιτικά ανύπαρκτη. Ο Ζώνη πρέπει να είμαστε ε, προδραστικοί και να είμαστε πρωταγωνιστές. Δεν έχουμε στρατιωτική εξουσία, αλλά έχουμε οικονομική εξουσία και στη Μέση Ανατολή μας θεωρούν ανύπαρκτους. Δεν έχουμε καμία σημασία στη Μέση Ανατολή, καμία. Πληρώνουμε για τους πρόσφυγες, έχουμε το πιο σημαντικό, το μεγαλύτερο εμπόριο με τη Μέση Ανατολή, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που κάνουν κουμάντο. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε επικουρική. θα συνεχίσουμε να είμαστε ένα τεράστιο στομάχι με ένα πάρα πολύ μικρό κεφάλι. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν τώρα στη μέση διαταξή που είναι το σημείο 4. Ετήσια έκθεση της ΥΠΑ Προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 130 είναι οι τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Σήμερα το συζητούμε για δεύτερη φορά. Νομίζω ότι καταφέραμε τις τελευταίες μέρες να βρούμε συμβιβαστικές τροπολογίες σχεδόν για όλα τα θέματα. Μερικές διανέμονται αυτή τη στιγμή συμβαστικές για να συμπληρωθεί. Το περισσότερο έχει συζητηθεί την περασμένη φορά συνεδρίαση των σκιωδών ε, εισηγητών και αν θυμούμε καλώς ήταν μεγάλη συνένεση. Τώρα, θα ήθελα να ξαναπώ το εξής. Θα προτείνω σε ορισμένε τροπολογίε να καταψηφιστούν, όχι επειδή τις θεωρώ λάθος επί της ουσίας, αλλά επειδή είναι υπερβολικά λεπτομερείς. Πάντα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος σε μια ετήσια έκθεση, ο καθένας να βάζει τώρα το δικό του μεράκι και αυτό που θεωρεί σημαντικό αν το κάνει αυτό ο καθένας, η έκθεση δεν έχει πια μήνυμα να εκπέμψει. Νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει από την αρχή της συζήτησης ότι ε, όσο το δυνατόν θα κρατήσουμε σε ένα σύντομο πλαίσιο αυτή την έκθεση. Αυτό δεν θα επιτύχει 100%, είμαι αρκετά ρεαλιστής για να το βλέπω, αλλά παρακαλώ να το λάβουμε υπόψη μας. Και κάποιοι από τους συντάκτες των τροπολογιών που δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβιβαστικέ, ίσως να το ξανασκεφτεί. Αν θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει την τροπολογία του, τη λεπτομερή. Γιατί για να έχει νόημα μια τέτοια έκθεση θα πρέπει να στέλνει γενικά μηνύματα και να μην είναι άθροισμα μεμονωμένων ατομικών δηλώσεων. Για μένα αυτό είναι το ζήτημα και το πρόβλημα που έχω. Αν το συζητήσετε στις πολιτικές σας ομάδες ε, στην κατάρτιση των καταλόγων ψηφοφορίας, ε, να τους το πείτε. Νομίζω έχω φτάσει στα όρια των όσων θα μπορούσε κανείς να δεχτεί. Ε, για να μην χαθεί το γενικό μήνυμα στο βωμό του μεμονωμένου και της επτομέρειας. Παρακαλώ να το λάβετε υπόψη αυτό και ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς το λόγο. Α, ήθελα να πω το ακόμα όταν θα μοιραστούν λύσεις ψηφοφορία στη συνέχεια με τις συμβαστικές κτλ. Είμαι στη διάθεσή σας και σήμερα και αύριο πριν την ψηφοφορία για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση έχετε και διμερός και ό,τι άλλο θέλετε. Και αν θέλετε να το ξαναδούμε και στους ε, σκιώδεις εισηγητές για να συμφωνήσουμε. Αλλά σας παρακαλώ να δείξετε μεγαλοθυμία να διατηρήσουμε έτσι μια γενική γραμμή, ένα ηρμό στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς το λόγο? Όχι? Καλώς. Να πάμε στο επόμενο θέμα λοιπόν. Ja, ich muss erst mal den Antrag fertig haben. Na Ost.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 Okay. So, uh, Mr. Tanok. Κύριε Τάνοκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Είχαμε μια αλλαγή προεδρίας, ήσασταν ταχύτατη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω ήδη δώσει την ομιλία μου στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής ε, για την Γενική Επισκόπηση της κατάστασης ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσεις προσχώρηση για τον Ευρωβούνιο. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν τα όσα είπα την προηγούμενη φορά. Μπορώ να πω όμως ε, σε αυτή τη φάση ότι έχουμε διαπραγματευτεί με επιτυχία με τη βοήθεια και των ε, υπαλλήλων της Επιτροπής με όλους τους κοιόδης εισηγητές από τι ε, κύριε ομάδε, 20 συμβαστικέ τροπολογίε έχουμε που νομίζουμε ότι θα μειώσουν σημαντικά ε, τον ε, όγκο των υπολείπων. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει συμφωνία και με τις υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε. 188 τροπολογίε είχαμε και νομίζουμε ότι έτσι θα συρρυκνωθεί σημαντικά ο αριθμό του. Θεωρώ ότι η έκθεση θα υπερψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία και με λίγα προβλήματα και διαφωνίε. Ο συνήθω ε, είναι καλά τα πράγματα με το Μαυροβούνιο. Σημειώνεται πρόοδο ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει ε, ένταξη. Έχουμε ανοίξει 16 κεφάλαια μαζί με τα κύρια κεφάλαια 23 24 για το σύστημα της δικαιοσύνη. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά ιδίως την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ε, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και του καθεξής. Όμως ε, η έκθεση θέλει να δώσει προσανατολισμό προς ε, την κυβέρνηση για αυτή την ανταξιακή διαδικασία και στηρίζει εν γέννη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται προβληματική έκθεση. Με τα χαρά να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων, αν θέλουν να πούν κάτι για συγκεκριμένες τροπολογίες. Εγώ έχω ήδη καθορίσει ε, τον κατάλογο των τροπολογιών που θα στηρίξω. Αν υπάρχουν διαφωνίες από συναδέλφους, μπορούν ενδεχομένως να σε επισημάνουν τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ντόλς. πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωση Μαυροβουνίου. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη προ τον κύριο Τάνοκ που αυτή η Επιτροπή πράγματι πάντα τηρεί το χρονοδιάγραμμα σε αντίθεση με άλλες ε, και έτσι έχασα την αρχή τη ομιλίας του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω αρχικά ε, για τη το, τις εργασίες του για το ψήφισμα για το Μαυροβούνιο. Από πλευρά μου εγώ ως πρόεδρος ε, της διπροσωπίας, επικεφαλής της διπροσωπίας, μπορώ να πω ότι ήταν ε, μια ιδιαίτερα παραγωγική και επικοδηματική διαδικασία και το ψήφισμα δείχνει μια σαφή και καθαρή δέσμευση ε, του Μαυροβουνίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπογραμμίζει ιδιαίτερως την σημασία της εφαρμογής Ω τομέα περαιτέρω εργασιών. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο τροπολογίες, αν μου επιτρέπετε συνάδελφοι, και οι δύο αφορούν τον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και έτσι βρισκόνται στο επίκεντρο τη ενταξιακή διαδικασία. Η πρώτη τροπολογία που θα ήθελα να επισημάνω είναι 129. Μιλάμε για ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων για τα άτομα με αναπηρία. Ένα από τα κύρια σημεία που αντιμετωπίζουν και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στο Μαυροβούνιο είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσια κτίρια, που είναι θεμελιώδη σημασία στοιχείο για να μπορούν να λειτουργούν στον δημόσιο βίο. Και πέρυσι το Δεκέμβριο, όταν ε, είχαμε ε, αντίστοιχα προβλήματα. Άτομα αναπηρία ακτιβιστέ δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο κτίριο και μάλιστα εκείνη την ημέρα που ακριβώ ε, μνημονεύαμε αυτή την ημέρα για τα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Είναι απαραίτητο ε, αυτά τα άτομα να έχουν ε, πρόσβαση ε, στα κτίρια όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις που καθορίζουν τη ζωή τους. Και δεύτερον, πολύ σύντομα, η 75 που μιλά για ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ε, διαμεσολαβητή. Ε, θα μπορούσε και αυτό να συμπεριληφθεί. Γνωρίζουμε όλοι οι ευρωβουλευτέ πόσο σημαντικό είναι ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για του Ευρωπαίου πολίτε. Όμω, ο Διαμεσολαβητή του Μαυροβουνίου αυτή τη στιγμή δεν έχει, ε, ο συνήγορο του πολίτη δεν έχει τι απαραίτητε αρμοδιότητε και πόρου. ο λαό του Μαυροβουνίου και η πολιτική και η κοινωνία των πολιτών όλοι θυμερίζονται τον ε, στόχο αυτό της ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να επιληφθούν οι τη προκλήση προκειμένου να ενταχθεί και αυτή η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα χρόνια. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κύριο Τάνοκ ε, για το εξαιρετικά αποκαθηματικό του πνεύμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Πλέγκοβιτ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ μέρου ε, του κ. Κοβάτσεκ που είναι σκιώδης συζητητής από το ΕΛΚ. Θα ήθελα να εκφράσω από την πλευρά του συγχαρητήρια στον κύριο Τάνο, όπως και στους υπόλοιπους σκιώδης συζητητές που καταφούσαν να φτάσουν σε συνένεση για σε ένα σημαντικό αριθμό συμβιβαστικών τροπολογιών ε, σε σχέση με την καλή κυβέρνηση, τα ΜΜΕ και το δικαστικό σώμα. Αυτά τα τρία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την συνολική μεταρρυθμιστική ατζέντα του Μαυροβουνίου. Τώρα έχουμε ανοίξει 16 κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις και βρίσκεται στην πρώτη θέση ε, των διαπραγματεύσεων σχέση με όλε τι χώρε ε, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κύριο Κοβάσεβιτ ε, αναφέρεται κυρίω στην εφαρμογή, γιατί στο όγκο τη νομοθεσία που υιοθετείται και πολλές φορές μέσω μιας δυναμικής διαδικασίας πρέπει να διασφαλίσουμε μια εύρωστη εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και να οικοδομήσουμε επαρκείς θεσμούς. Αυτό που χρειάζεται για την επιτυχία του Μαυροβουνίου είναι να ξεπεραστούν οι πολιτικές διενέξεις που υπάρχουν στη χώρα και στην κοινωνία και βέβαια αυτό θα βοηθήσει ε, να ε, ε, παρελθούν και οι απαραίτητες οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις πολιτικές. Επίσης αναφέρεται και στην βελτίωση του περιβάλλοντος για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το να μην υπάρχουν εξαρτήσεις επίσης ε, σε αυτό το τομέα. Αυτό είναι προϋπόθεση για μια εύρυθμη κοινωνία που θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο περιβάλλον για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε και τη συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών σε διάφορα ζητήματα. Συμπρασματικά το Μαυροβούνιο μπορεί να ενταχθεί με επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν υπάρχει πολιτική βούληση. Ευχαριστούμε κύριο Χάουιτ. Συγγνώμη, θα ήθελα να ζητήσω ε, για, από πλευρά όδου εισηγητού, μιλώ εκ μέρους του, του κυρίου Ανδουλάκη, και θα ήθελα να πω ότι τον ευχαριστούμε θερμά, τον εισηγητή, πάρα πολλά πράγματα στην έκθεση είναι, αποτελούν πολύ καλά στοιχεία και θα θέλαμε να εκφράσουμε τη στήριξή μας δίνεται σημασία στο κεφάλαιο 23 και αυτό φαίνεται ότι παράγει αποτελέσματα. Έχει ενισχυθεί η διατύπωση για το Κοινοβούλιο, για τα ε, δικαιώματα ομοφιλοφίλων, ε, φιλομεταβατικών και το καθεξής. Υπάρχει στήριξη για καλύτερη δράση εναντίον των διακρίσεων γενικότερα. Και όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετικά. Οι τροπολογίες των σοσιαλιστών ευθυγραμμίζονται με αυτή τη γραμμή. Ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες για μεταρρυθμίσεις από πλευράς Μαυροβουνίου και δίνουμε έμφαση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της ανισότητας, της φοροαποφυγής ε, και των διακρίσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, την καταπολέμηση των υψηλών επιπέδων ανεργίας, του υψηλού επίπεδου της φτώχειας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Τάνεκ στηρίζει την τροπολογία 156, τη δική μας. Θα μπορούσα να τη σχολιάσει παρακαλώ. Αυτό θα θέλαμε. Ζητούμε τη στήριξή του για να περάσει η τροπολογία 156. Και τώρα, να σας πω ότι το συζητήσαμε στην ομάδα μου, εν ώψη της ψηφοφορίας αύριο, της ψήφισης της έκθεσης και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες ευαισθησίες για το θέμα των εγκλημάτων πολέμου και σε αυτή τη χώρα και σε άλλες. Πολλή συζήτηση γίνεται πρόεδρε στην αίθουσα και δεν μπορώ να μιλήσω. Μπορείτε να ανακαλέσετε στην τάξη ε, τους κυρίους που μιλούν. Ο πρόεδρος ανακαλεί στην τάξη. Συνεχίζει ο κύριος Χάουετ. Για το θέμα λοιπόν των εγκλημάτων πολέμου και των σχετικών τροπολογιών, το σημαντικό είναι να έχουμε διατύπωση που θα στηρίζει την ανάληψη δράσης έτσι ώστε να μην υπάρχει ατιμορρησία. Ωστόσο, η διατύπωση αυτή θα πρέπει να είναι μη επιλακτική και να καλύπτει όλα τα εγκλήματα πολέμου. Ορισμένες τροπολογίες λοιπόν είναι σημαντικές υπό αυτή την έννοια. Ως προς την τροπολογία 42, ε, συμφωνούμε απολύτως με τη διατύπωση εδώ όμως το κατά πόσο αυτό πρέπει να μπει μέσα σε ψήφισμα για τη συγκεκριμένη χώρα ή με άλλο τρόπο, καλό είναι να γίνει συζήτηση, να γίνει διάλογος γι' αυτό. Το ίδιο και για το αίτημα του Μαυροβουνίου να ε, ε, γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αν είναι η διατύπωση τοποθετημένη στο σωστό σημείο και αυτό αξίζει συζήτησης. Ίσως θα πρέπει να ψηφίσουμε κατά συνείδηση για το θέμα αυτό. Και αν το καταψηφίσουμε δεν είναι ότι καταψηφίζουμε την αρχή, απλά θα καταψηφίσουμε εάν συμβεί για να πούμε ότι δεν είναι το σωστό σημείο στο κείμενο να μπει μια τέτοια διατύπωση. Σε γενικέ γραμμέ η έκθεση είναι πολύ συνενετική και μπορούμε να τη στηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Τζαμπάνσκι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για τη δουλειά του. Πράγματι, έχει λάβει υπόψη του τις επιθυμίες των πολιτικών ομάδων και το λέω αυτό διότι πιστεύω ότι το Μαυροβούνιο είναι μία από τις χώρες οι οποίες είναι και πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλωστε από πλευράς βασικών κριτηρίων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις του Μαυροβουνίου και σε ό,τι αφορά τις συμβιβαστικέ λύσεις που έχουν επιτευχθεί, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, μπορώ να στηρίξω την έκθεση του κ. Τάνοκ. Ευχαριστώ. Mr. Ευχαριστώ Ράντος. Ευχαριστώ κύριο Ράτος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Τάνοκ για την πολύ ευρία προσέγγιση που υιοθέτησε για την επίτευξη σεμιβαστικών τροπολογιών. Θα ήθελα όμως να πω ότι υπάρχει ένα θέμα διότι καλούνται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ να επιταχύνουν την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ. Και εγώ νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό όλη η ακτή της Αδριατικής να είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Όλες οι χώρες δηλαδή. Αυτό είναι προς της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Και αυτό Ενδεχομένως δεν είναι έτσι διατυπωμένο στην παράγραφο 22 της συμβιβαστικής τροπολογίας. Υπάρχει όμως μια άλλη τροπολογία που εκφράζει το ίδιο μήνυμα και γι' αυτό καλώς του ε, τους συναδέλφους να τη στηρίξουν. Καλεί τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέλη του ΝΑΤΟ να στηρίξουν την προσχώρηση του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να υποστηρίξω πλήρως ε, τη θέση που εκφράστηκε από τον σκιώδη συγητή του ΕΛΚ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Παραδοσιακά προετοιμάζει πολύ καλές εκθέσεις ε, και φυσικά τα πράγματα είναι πιο εύκολα επειδή υπάρχουν καλές επιδόσεις από το Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο ε, είναι, έχει πραγματικά ηγετική θέση στην διαδικασία προσχώρησης στην περιοχή και νομίζω ότι πρέπει να τον εθωρύνουμε να συνεχίσει την καλή δουλειά. Πιστεύω ότι πρέπει να συγχαρούμε τη χώρα για την ε, πλήρη ευθυγράμμιση με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η χώρα παίζει ένα θετικό ρόλο και έχει και καλές σχέσεις με τις όμορες χώρες. Βέβαια, υπάρχουν κάποια εκκρεμή ζητήματα, στα οποία πρέπει να προσδώσουμε προσοχή και θα πρέπει να εργαστούν και οι εταίροι μας από το Μαυροβούνιο τα θέματα αυτά και εγώ θα καταθέσω κάποιες πρωτολογίες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να ενδυναμώσουμε την ε, σαφή, το σαφή διαχωρισμό μεταξύ κράτους και κομματικής γραμμής. Δεύτερον, πρέπει να αυξηθεί η υποστήριξη του ρόλου του Κοινοβουλίου σε όλη την ευρωπαϊκή διαδικασία προσχώρησης. Και επίση έχω καταθέσει και κάποιε πρωτολογίε για την ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση, γιατί είναι ένα θέμα που εξακολουθεί να μα ανησυχεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Τάνοκ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πάσκου. Απλώς για να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, ε, κύριε Ντότ, θα χαρεί να ακούσει ότι και οι δύο τροπολογίες και την 129 και την 75 θα τις υποστηρίξω και άκουσα και τα σχόλια του κύριου Πλένκοβιτς εκ του κύριου Κόβετσεφ για το θέμα της εφαρμογής. Φυσικά αυτό είναι πολύ ζωτικό, αν και μερικές φορές είναι δύσκολο να τα μετρήσουμε αντικειμενικά αυτά τα πράγματα. Για το θέμα που έθεσε ο κύριος Χάουιτ για την τροπολογία 156, πιστεύω ότι τα νούμερα που αναφέρθηκαν δεν είναι σωστά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα ε, περισσότερο υποκειμενικό. Τώρα εγώ θα ανησυχούσα σε σχέση με τα ενεργικά μέσα της αγοράς. Ε, μάλλον είναι σοσιαλιστικός λόγος αυτός ε, και προκαλεί κάποιες ανησυχίες. Ε, μάλλον κάθε ομάδα θα ψηφίσει ανάλογα με το τι πιστεύει σε σχέση με το τι είναι ένα ενεργό μέτρο στην αγορά εργασίας και Ευρωπαίοι συντηρητικοί και δεν ίσως να μπορούσαν να υποστηρίξουν. Τώρα για τα θέματα του κ. Ράντος για το ΝΑΤΟ. Νομίζω ότι και ο Ρίτσαρτ το έθεσε ή έκανε μια αναφορά με ένα πιο σκεπτιστικό τρόπο. Φυσικά η συζήτηση αυτή προκύπτει κάθε φορά που αναφέρουμε το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Φυσικά το ΝΑΤΟ δεν σχετίζεται άμεσα στη διαδικασία προσχώρησης. Η Αλβανία, τους χάρη, ήδη είναι πλήρες, πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ αλλά η διαδικασία του ΝΑΤΟ επικαλύπτεται σε ό,τι αφορά το θέμα τα απορριθμιστικά μέτρα της ελεύθερης αγοράς που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, την ελευθερία των ΜΜΕ, καλή διακυβέρνηση, καταπολέμηση της διαφθοράς οργανωμένων κλίματος κτλ. Έτσι λοιπόν, χάρηκα που άκουσα να υποστηρίζει αυτό ο κύριο ράντο, κυρίω σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας. Τώρα, καθώ η Ρωσία προσπαθεί και πάλι να ασκήσει μόχλευση και επιρροή σε συγκεκριμένες χώρες και αυτό μάλιστα με έναν τρόπο που αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, τι κοινέ, στρατηγικέ στρατηγικές κτλ. Και μπορώ να πω το Μαυροβούνιο έχει πλήρω ευθυγραμμιστεί με την πολιτική επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία λόγω της, ε, του πολέμου με την Ουκρανία. Για την 178 ευχαρίστως ε, θα την υποστηρίξω, αν και άλλες πολιτικές ομάδες μπορούν να με την υποστηρίξουν για λόγους που ανέφερα. Και τώρα, φυσικά, ο κύριος ε, Κούκαν ο οποίος ε, είναι πραγματικά εμπειρογνώμονας ε, στην περιοχή και πολύ μεγάλος ε, διπλωμάτης. Εκτιμώ τα όσα έχει βάλει στην έκθεση και μια τροπολογία που μπορεί να θυμηθώ που αφορά το να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των πόρων του κόμματος από τους πόρους του κράτους είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστώ θα το υποστηρίξω. Αυτά πάνω κάτω νομίζω ότι κάλυψε όλα τα θέματα που τέθηκαν. Um, Ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνο. Πολύ γρήγορα αλλάζει η Προεδρία εδώ και ο κύριος Στούτσμα μου λέει ότι και ε, ο κύριος Καστάλτο και η κυρία Λούνατσεκ θέλησαν να μιλήσουν που έφτασαν αργότερα και δεν έλαβαν το λόγο. Ε, όσοι δεν ήθιστε θα τους δώσουμε το λόγο παρόλο που έχει συνοψίσει ο εισηγητής για την ε, καλή συνεργασία και το πνεύμα που διέπτει την Επιτροπή μας. Θα κάνουμε αυτή την εξαίρεση. Ποιο θα μιλήσει πρώτος, κύριος Καστάλτο; Ευχαριστώ. Εγώ δεν άργησα, απλώς δεν με είδατε. Απλώς ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον συνάδελφο Τάνοκ για το έργο του στην έκθεση αυτή. Είναι πολύ πιστική και όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή το Μαυροβούνιο είναι η χώρα που έχει προχωρήσει περισσότερο στη διαδικασία προσχώρησης και ε, είναι πολύ θετικό όταν αξιολογούμε την πρόοδο. Ήθελα να πω ότι εγώ είμαι θετικός απέναντι στη συμβιβαστική 11 σε ό,τι αφορά τα μέσα που πρέπει να δοθούν ε, στις διοκτικές αρχές, στις δικαστικές αρχές για να υλοποιήσουν καλύτερα το έργο τους και επίσης και το να έχουμε και νέα νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα είναι κάτι πολύ θετικό. Φυσικά, αν πάντα το έχουμε αποτελεσματική εφαρμογή. Τώρα, μια άλλη συμβιβαστική τροπολογία με την οποία συμφωνεί η ομάδα μου είναι η 19 για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Θεωρούμε ότι είναι θεμελιώδες να καλέσουμε το Μαυροβούνιο να αναπτύξει αηφόρο ενεργητική πολιτική και να αναπτύξει φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα η εθνική στρατηγική για την ενέργεια που θα λαμβάνει υπόψη και τη χρήση νέων πηγών ενέργειας μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα που θα εξαχθεί και σε άλλες υποψήφιες χώρες της περιοχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που δίνετε και την ευκαιρία να ξαναμιλήσω. Κανονικά στι 4 έπρεπε να αρχίσει αυτή η συζήτηση και μέχρι στι 4 και 4 είχα μιλήσει όλοι και ο εισηγητή δύο φορέ και όλοι οι άλλοι σκιώδε. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ τον εισηγητή για τι διαπραγματεύσει συμβαστικέ. Είχε πολύ μεγάλη προθυμία, έχει υιοθετήσει και δικέ μα τροπολογίε. Παρ' όλα αυτά, τέσσερις δικές μας. Θα παρακαλούσα να τι ξανασκεφτείτε για τον κατάλογο ψηφοφορίας σα και την υποστήριξη. Και ορισμένοι άλλοι ε, εδώ θα τι υπερψήφισαν. Ε, η πρώτη είναι η 42. 42. Όπως και πολλοί άλλοι εδώ εμείς επικρίνουμε τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί προεκλογικά είχε πει ότι την επόμενη πενταετία δεν θα υπάρξει νέα διεύρυνση. Όχι ότι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό, αλλά νομίζουμε ότι έστειλε λάθος μηνύματα σε χώρες υποψήφιες ε, για τη διεύρυνση ή ε, που επιθυμούν τη διεύρυνση γιατί τους αποθαρρύνει αυτό. Γιατί είναι λίγο πρόθυμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ θα μπορούσατε να το σκεφτείτε, ε, να το επαναλάβουμε γιατί εκφράζει τη θέση του Κοινοβουλίου, όχι μόνο εμάς μόνο των Πρασίνων. Ε, η 69 τροπολογία, 69, ε, για τη χρήση των δημοσίων χρημάτων και η 16 για την πρόσβαση του κοινού στις ε, πληροφορίες, στην ενημέρωση. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε εμείς και εδώ στο Κοινοβούλιο μας και σε άλλα κοινοβούλια και η τελευταία είναι 160 για την ε, προστασία της φύσης, ε, της βιοπικιλότητας. Συμφωνείτε γενικά για το περιβάλλον, αλλά ειδικά στο Μαυροβούνι. Είναι μια χώρα που έχει κατοχυρωμένο στο σύνταγμά της ε, οικολογικά ζητήματα. Οι μεγάλοι ποταμοί θέλουν ιδιαίτερη προστασία και η βιοπικιλότητα. αν το ξανασκεφτείτε ή αν το σκεφτείτε καν να υποστηρίξετε αυτές τις τέσσερις τροπολογίες μας θα σας ιδιαίτερα γνώμων Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Λούνατσεκ. Κύριε Τάνοκ, ίσως θέλετε να σχολιάσετε για το θέμα του κυρίου Καστάλτο. Δεν έρθετε σε ερωτήσεις, μάλλον τοποθέτηση έκανε για τις συμβαστικές που του άρεσαν. Δεν χρειάζεται να απαντήσω. Κάθε χρόνο αυτή τη συζήτηση έχουμε με την κυρία Λούνατσεκ. Βέβαια δικαίωμά σας είναι ε, και εξ ονόματος της ομάδας σας να προσπαθείτε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω η δική μου ομάδα, δεν ξέρω, οι άλλοι μπορεί να διαφέρουν. Κάθε βουλευτής θα ψηφίσει με βάση τη δική του άποψη και της πολιτικής του ομάδας. Σε σχέση τώρα με τη δήλωση του Γιούνκερ, μπορείτε να θεωρείτε ότι είναι λυπηρό. Εγώ θεωρώ ότι το αυτονόητο είπε ο άνθρωπος. επιταχυμένη διεύρυνση νομίζω αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Υπάρχει μια κόπωση ε, από τις διευρύνσεις και στις χώρες αυξάνεται και ο ευρωσκεπτικισμός. Ε, τουλάχιστον δική μου πολιτική ομάδα δεν θα πίεζε το Μαπροβούνι να μπει στην Ένωση την επόμενη πενταετία. Ε, παραμένω δυστυχώς αντίθετος σε αυτή την τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την άλλη που είπατε ποια ήταν 160 για το περιβάλλον και τα ποτάμια. Εδώ αναφέρεται ειδικά ενεργειακά έργα και φαίνεται ότι είστε αντίθετοι με ένα υδροελεκτρικό εργοστάσιο που σχεδιάζουν. Μπορεί να είναι θεμητές οι ανησυχίες σας για το περιβάλλον, αλλά το ενεργειακό μείγμα που έχει επιλέξει το Μαυροβούνιο είναι δική του κυρίαρχη απόφαση. Είναι για να ξέρει το κράτος, δεν θα του πούμε εμείς τι φράγματα θα φτιάξει και τι ενεργειακό μείγμα θα έχει και τι έργα θα κατασκευάσει. Εφόσον συνάδει με το κεκτημένο το κοινοτικό δεν έχουμε να του πούμε τίποτα. Έχουν αυτό αναγορηθεί σε οικολογικό κράτος. Τώρα τι μορφή παίρνει αυτό και τι σάρκα και οστά. Αυτό είναι θέμα μιας κυρίας τη χώρα να το διαμορφώσει. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Το θέμα τη διεύρυνση και το τι θα συμβεί την επόμενη πενταετία δεν είναι κάτι που ανησυχεί και ευρωματίζει μόνο το Μαυροβούνιο, αλλά όλες οι χώρες της Νότια-Ανατολικής Ευρώπης που προσπαθούν να κάνουν μεταρρυθμίσεις. Και εμείς ε, οφείλουμε να τις υποστηρίξουμε και ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο. Ε, θα ολοκληρώσουμε λοιπόν εδώ το θέμα αυτό για το Μαυροβούνιο για το 2014 και ευχαριστώ τον, ε, τον εισηγητή και τους σκιώδης. Και προχωρούμε τώρα στο επόμενο μας ε, θέμα ε, που είναι η έκθεση ε, προόδου του 2014 για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εισηγητής είναι ο κύριος Βάιγκελ. Είναι η δεύτερη φορά που συζητούμε την έκθεση αυτή. Όπως όλοι γνωρίζετε, η χώρα αυτή πρόσφατα αντιμετώπισε μια κατάσταση που αφισβητήθηκε η ίδια η πολιτική του σταθερότητα ε, λόγω κάποιων ποινικών υποθέσεων ε, και ε, παρακολουθήσεων και υποκλοπών έχει επιδεινωθεί το πολιτικό κλίμα και άρα θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να διατηρηθεί ευρωπαϊκή προοπτική και πορεία. Γι' αυτό η Επιτροπή μας απευθύνει έκκληση προς όλους τους παράγοντες και ενεχομένους για να ξέρουμε ποιες είναι οι προτεραιότητες ε, της ε, χώρας και πώς θα οδηγηθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγητής ε, είναι ο κύριος Βάγγελ, 296 είναι οι τροπολογίες, 16 συμβιβαστικές έχουν να κάνουν με ε, σημαντικά ζητήματα όπως είναι η ονομασία της Μακεδονίας, ε, λέει ο Πρόεδρος, ε, οι συνομιλίες, η σταθεροποίηση της πολιτικής σκηνής στη Μακεδονία ή η επιδείνωση της κατάστασης δεδομένων των προσφάτων εξελίξεων στην ελευθεροτυπία, στην κοινωνία των πολιτών, εξωτερική πολιτική κτλ. Εδώ και πολλά χρόνια παρά τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις και γι' αυτό οι φίλοι μας από τη Μακεδονία κάπως δυσφορούν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Βάγγελ για να μας δώσει περισσότερες υποβίδαλη. Ε, Ευχαριστώ. Ήδη είπατε όσα είχα να πω κι εγώ. Δηλαδή, οι ε, συνάδελφοι της Επιτροπής, ε, καθώς και οι σχεώδεις εισηγητές, έχουν ε, κάνει ένα πολύ σημαντικό έργο. Τα ζητήματα που αφορούν την πρώην Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι εξαιρετικά περίπλοκα, γι' αυτό και ευχαριστώ τους συναδέλφους που <clears throat> συνέβαλαν στην τροποποίηση του κειμένου, στον ολοκλήρωση του κειμένου και τη συμπλήρωσή του, γιατί τώρα είναι βελτιωμένα το κείμενο. Ευχαριστώ και όλες τις υπηρεσίες που μας ε, στήριξαν ε, κατά την επίτευξη αυτών των 16 συμβαστικών τροπολογιών που αντικατοτρίζουν στο βαθμό του δυνατού την κοινή θέση σε ένα ευρύ φάσμα κοινών ζητημάτων. Με ένα τόσο σημαντικό ρυθμό τροπολογιών είναι αδύνατον να τα ενσωματώσουμε όλα. Μάλλον στι 16 συμβαστικέ που έχουμε που είναι πολύ μειωμένε. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα. Αλλά βεβαίω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, να σχολιάσετε μπορείτε να το πείτε. Η διαδικασία αυτή τώρα ήταν πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την διαμόρφωση ενός πνεύματος συνέχειας στην ευρωπαϊκή διαδικασία διεύρυνση. Η Φύρομ είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει την πραγματεύση εδώ και πολλά χρόνια και αυτό είναι άποψη και όλων όσοι συνέβαλαν στην ε, κατάρτιση της ε, γνωμοδότησης. Ωστόσο, εξαιτία του ζητήματο ε, των διαφωνιών και αντιθέσεων με την Ελλάδα, υπάρχει αυτό το διέξοδο που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Ένα από τα κύρια ζητήματα της έκθεσης είναι η ΦΥΡΟΜ να έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Και αυτό, βεβαίως, δεν είναι κάτι το οποίο θα μας ε, αποτρέψει να επιλύσουμε αυτά τα αμοιβαία ζητήματα. Πρέπει να γίνει αυτό πριν από τη λήξη και ολοκλήρωση τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, οι συνέπειες αυτού του αδιεξόδου είναι αρνητικές. Ουσιαστικά ε, μας οδηγούν σε ένα οικονομικό τέλεμα και πολύ αρνητικό πολιτικό κλίμα στη Φύρο. Η έκθεση προόδου ε, προτείνει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και παράλληλα να καταβληθούν σημαντικέ προσπάθειε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση κάποιων παρανοήσεων και ζητημάτων προβλημάτων που ενδεχομένω ανακύψουν σε διμερεί σχέσει. Όπω γνωρίζετε, στη Φύρομ σίγουρα υπάρχουν και πολιτικέ ε, επιπλοκές, υπάρχει και κρίση εμπιστοσύνης οι βασικοί πολιτικοί φορείς ε, μποϊκοτάρουν το Κοινοβούλιο. Υπήρχαν και σημαντικές κατηγορίες και από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά ενέργειες που θα πρέπει να επιληθούν δικαστικώς και πράγματι συνέβη αυτό. Γι' αυτό και θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καλέσει τη ΦΥΡΟΜ να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και εμείς το κοινοβουλευτικό μας έργο ε, να δώσουμε την απαραίτητη έμφαση στα ζητήματα που είναι πραγματικά κομβική σημασία στην ΦΥΡΟΜ. Και αν αυτό σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να διαμεσολαβήσουμε εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να λειτουργήσει ως μεσολαβητής ή οποιοδήποτε άλλος από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να εξετάσουμε. Το αδιέξοδο λοιπόν στην διαδικασία διαπραγματεύσεων και οι αντιρρήσεις προς τη διαπραγμάτευση έχουν οδηγήσει σε προβλήματα και σε ό,τι αφορά τις ε, εθνικές σχέσεις λειτουργεί και διαμορφώνει αρνητικές δυσμενείς όρους για το ευρύτερο οικονομικό πλαίσιο και θα πρέπει λοιπόν και εμείς να κάπως ε, να μειώσουμε αυτό το φορτίο που έχει ε, επομιστεί η ΦΥΡΟΜ γιατί έχει δεχθεί σοβαρές διακρίσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ΦΥΡΟΜ. Αυτό δεν βέβαια σημαίνει ότι και οι πολιτικοί φορείς σε αυτή τη χώρα δεν συμβάλλουν στην επιδείνωση της κατάστασης. Η έκθεση πρόοδου επίσης αναφέρει κάποιες παραμορφώσεις ούτως υπήν στον ε, τομέα ε, της ε, ελευθερίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε ό,τι φορά την άσκηση πιέσεων προς τα μέσα ενημέρωσης. Μπορούμε να αναφερθούμε σε επιλεκτικές ε, δικαστικές διαδικασίες. Υπάρχουν προβλήματα σε ό,τι αφορά τις μειονότητες, τους LGBT και άλλα ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση προόδου. Καθώς ε, και μία δήλωση ότι η ΦΥΡΟΜ έχει επιτύχει πολλά σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την οικονομία, την απασχόληση αλλά και την περιφερειακή συνεργασία. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ε, προτάσεις και συστάσεις. Έχουμε λίγο χρόνο να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον συνάδελφο Πέτελε, επικεφαλής της κοινοβουλευτική Επιτροπής για τις ε, σχέσει με την ΦΥΡΟΜ και μετά συνάδελφος Βρέντε, εκ μέρου του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Μπορώ να υποστηρίξω την γνωμοδότηση του συγητή το κύριο πολιτικό σημείο θετηρίας είναι η γνωμοδότηση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η χώρα αυτή πληρεί τα κριτήρια για την έναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Χαίρομαι που έχουμε διασκεδάσει κάποιες πολιτικές φήμες και ξεκινήσαμε να προσδίδουμε δυναμική στην διαδικασία προσχώρησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι σημαντικό ότι τα κύρια θέματα έχουν, τα έχουμε βάλει σε αξιόπιστες αναλογίες, δηλαδή η έκθεση αυτή είναι ισορροπημένη και αντικατοπτρίζει το ευρωπαϊκό πνεύμα. Φυσικά υπάρχουν κάποια κρεμή θέματα που πρέπει να επιληθούν, θα πρέπει να τα εξετάσουμε στο πλαίσιο των κοινών μας συμφερόντων. Είμαι βέβαιος ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων θα μας δώσει καλύτερες δυνατότητες για να επηρεάσουμε τη διαδικασία αυτή και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποφύγουμε οποιοδήποτε διέξοδο. Είδαμε ότι οι ορισμένες προσεγγίσεις δεν εγγυώνται την πρόοδο που θέλουμε να πετύχουμε οποιαδήποτε είδους αβεβαιότητα που έχει να κάνει με τη διαδικασία προσχώρησης στη Φύρο. Αυτό δεν βοηθά στο να λυθούν οι εσωτερικές πολιτικές εντάσεις. Φυσικά έχουμε πολιτική ευθύνη με ένα κοινοβουλευτικό τρόπο να προσπαθήσουμε να υπερβούμε αυτό το status quo γιατί σίγουρα δεν θα μας επιτρέψει να έχουμε βελτιώσεις. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, γιατί η σκέδη δεν είναι εδώ και ο κύριος Πρέντα μου ζήτησε να διαβιβάσω την απόψή του. Η πολιτική μας ομάδα είναι ικανοποιημένη με την έκθεση αυτή. Είμαστε ικανοποιημένοι με τις 16 συμβιβαστικές τροπολογίες, μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Πιστεύω ότι αυτές ε, οι τροπολογίες ε, είναι ισορροπημένες και επίσης σέβονται και τις πολιτικές μας γραμμές. Δεν ήταν εύκολες οι διαπραγματεύσεις. γιατί πάντοτε ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις βουκαλικές και ελληνικές απαιτήσει. Όμως, ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν βάζουμε περαιτέρω εμπόδια στον δρόμο των διαπραγματεύσεων. Οι προτάσεις ε, του κυρίου Πρέντα και της κυρία Μέκαβελ έχουν συμπεριληφθεί σε κάποιες ε, προτάσεις μας, όπως η τροπολογία 7. Και νομίζω ότι είναι και επαρκή η διατύπωση σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Η πολιτική μας ομάδα είναι επίσης ικανοποιημένη με το γεγονός ότι έχουμε βρει καινή γλώσσα για ορισμένα θέματα που είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Ευχαριστώ κύριε Πέτερλε. Τώρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Χόλ. Ευχαριστώ. θα ήθελα να πω ότι και εμένα μου άρεσε που ήμουν ε, εισηγητής ε, τα προηγούμενα χρόνια, όμως ε, τη Κιταλή και θέλω να του ευχαριστήσω για τον τρόπο που εργάστηκε και να τον δώσω όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη. Νομίζω ότι έχουμε εδώ ένα καλό σύνολο συμβιβασμών. Χρειάστηκε περισσότερος χρόνος διαπραγμάτευση, όμω υπήρχαμε πολλά κοινά σημεία και νομίζω ότι βρήκαμε πώς να γεφυρώσουμε κάποιες διαφορές που υπήρχαν σε αυτή την Επιτροπή κυρίως αναφέρομαι στη συζήτηση που είχαμε για τη συνταγματική αλλαγή. Η ιδέα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση Νομίζω ότι είχαμε μια αρκετά σκληρή παράγραφο για την ελευθερία των μεσών μαζικής ενημέρωσης, αλλά αιτιολογείται. Και χαίρομαι και για τα θέματα των ΛΟΑΔΜ και νομίζω ότι βρήκαμε έναν τρόπο να πούμε ότι όλοι μπορούν να το υποστηρίξουν και Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κάτι τέτοιο και επίση ε, σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στην εξωτερική πολιτική και στην ΚΕΠΑ και την ευθυγράμμιση της χώρας που θέλουμε να δούμε, ε, νομίζω ότι αυτό η διατύπωση που έχουμε θα στείλει ένα μήνυμα στη ΦΥΡΟΜ. Και νομίζω ότι το έχουν ήδη λάβει οι φίλοι μας το μήνυμα αυτό, όπως ε, είπατε κύριε Πλένκοβιτς στις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Είχαμε πολύ μεγάλες ε, δυσκολίες ε, στο θέμα να αντιμετωπίσουμε το θέμα των σχέσεων μεταξύ των κομμάτων ε, στα Σκόπια και όλοι μας χρειαστήκαμε χρόνο για να σκεφτούμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να απαντήσουμε Κάποιοι θα προτιμούσαν ε, να, μην πούμε τίποτα, κάποιοι από τη Φύροπο. Όμω νομίζω ότι από εμά ε, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν υπεύθυνο ω κοινοβούλιο. Τώρα, ε, η διατύπωση που έχει βρει ο εισηγητή νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα και στα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα στη για το πόσο σημαντικός είναι ο πολιτικός διάλογος και νομίζω ότι μεταξύ του ΕΛΚ και των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών προσπαθήσαμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο από κοινού για να τα επηρεάσουμε αυτά στη χώρα και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ξέρω ότι η κυρία Μνάκοβέη ε, υπήρχαν ε, κάποιες προσπάθειες για κάποια μετακίνηση, υπήρχε όμως αντίσταση από τον κύριο Βάικλ και τον υποστηρίζουμε. Θεωρούμε ότι είναι ισορροπημένος τρόπος που τα έχετε παρουσιάσει και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι ισορροπημένη η διατύπωσή μας. Και Κάτι τελευταίο. Υπάρχει μια χωριστή παράγραφο για ε, ε, ψηφοφορία την παράγραφο 164. Έχουμε εδώ μια πρόσθετη διατύπωση που θέλαμε να δούμε. Δεν ε, μπορέσαμε να τη συμπεριλάβουμε ομόφωνα στο συμβιβασμό. Θα υπάρχει πρόσθετη ψηφοφορία και υπάρχει μια ανησυχία τη δική μας ομάδα για την ε, αλλαγή στην νομοθεσία σε σχέση με τον ορισμό του γάμου ε, και ελπίζω ότι θα μπορέσουν οι υπόλοιποι να υποστηρίξουν αυτή την πρόσθετη διατύπωση. Τώρα, για κάποια ε, θα ευαίσθητα θα ερχόμουν να ήταν καλύτερα τα πράγματα στη Φυρώμα, αλλά ίσως και εδώ καλύτερα. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η έκθεση θα μας προωθήσει για να δημιουργήσουμε κάποια κριτήρια για το πώς θα συσχετιστούμε με τη χώρα τα επόμενα πέντε έτη και φυσικά αναμένω όταν θα πάει η έκθεση στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ κύριε Χάουιτ. Ναι, φαίνεται ότι ήσασταν ο προηγούμενος εισηγητής για τη ΦΥΡΟΜ. Τώρα εκ μέρους του ECR, ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ την συντομία. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ τον νέο εισηγητή κύριο Βάγγελ, που είναι πολύ καλός ε, διάδοχος σε ό,τι αφορά τα ζητήματα και ειδικώ ε, τα ζητήματα της ευρύτερης περιφέρειας. Κατά τη γνώμη μου, παραμένει μια σημαντική πρόκληση αυτό το θέμα σε ό,τι αφορά την ε, δίκαιη διαδικασία προσχώρησης. Σε νέα χρόνια έχει το, λάβει το καθεστώ επισήμω τη υποψήφια προστατεύση χώρα. Είναι το κύριο ζήτημα αυτό με την Ελλάδα. Δεν έχουν προχωρήσει και τα πράγματα για να ανοίξουν οι διαπραγματεύσει στα επιμέρου κεφάλαια του κεκτημένου. Έχουμε 16 συμβαστικές τροπολογίες. Εγώ παρευρέθη στις διαπραγματεύσεις. Η ομάδα μου τις στηρίζει. Καλύπτουν μετά περισσότερα κύρια ζητήματα. Υπάρχουν, υπάρχει αυξανόμενος προβληματισμός για την πολιτική σταθερότητα, την πόλωση, τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, την ελευθερία του τύπου και ούτω καθεξής. Όμως η ε, η ΦΥΡΟΜ καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε ε, σε ό,τι αφορά ε, τι αντιπραγματεύσει και το γεγονό ότι δεν κινείται παρότι δηλαδή δεν υπάρχει σημαντική πρόοδο ό,τι αφορά την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε και έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα. Όπως είπα, θα υποβάλουμε και εμεί τροπολογίε, όμω η ομάδα μου και εγώ προσωπικά θεωρούμε τον ορισμό του γάμου ένα ιστορικό ζήτημα ε, του, της κάθε χώρας. Δεν έχει λόγο και αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να το θίξει ε, ως τμήμα του κεκτημένου. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Η κυρία Σακοράβα έχει τον λόγο από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ συνολικά για το ψήφισμα, γιατί την προηγούμενη φορά δεν μπόρεσα λόγω τη αλλαγή του προγράμματο. Κύριε Βάγκελ, το ψήφισμα που προτείνεται διαπιστώνει, όπω ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος, οπισθοδρόμηση στην Φύρο σε κέριου τομεί. Όπω είναι το κράτο δικαίου, της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών, τη ελευθερία τη έκφρασης και τη ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Παρά το γεγονός όμως ότι η ΦΥΡΟΜ έχει δρομήσει στους μήνες αυτούς σε όλους τους τομεί προτεραιότητα όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, στι σχέσει καλής γειτονία και στο ονοματολογικό, τόσο για εσάς όσο και για την Επιτροπή, όλα αυτά τα αρνητικά που έχουν χειροτερεύσει κατά το τελευταίο χρόνο, αθριζόμενα, συνιστούν πρόοδο της, πρόοδο της χώρας και γι' αυτό προτείνεται την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Θέτω λοιπόν ευθέω το ερώτημα, ποιον εξυπηρετεί αυτό ο θεσμικό ακροβατισμό, ποια σκοπιμότητα υπηρετεί η πλήρη περιφρόνηση τη αρχή τη αιρεσιμότητα που συνιστά βασική αρχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει. Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι η επιβράβευση τη κακή απόδοση μια υποψήφια χώρα αποτελεί ευθεία υπονόμευση των θεσμών των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως υπονομεύει την δυνατότητα προόδου και εξέλιξης της χώρας. Θέτω τα ερωτήματα αυτά, γιατί επειδή ακριβώ δεν υπάρχει απάντηση, προχωράτε σε λογικά, νοητικά άλματα που επιμένουν να συνδέσουν την αρνητική απόδοση της ΦΥΡΟΜ σε μια σειρά από κέριους τομείς με την συνεχιζόμενη καθυστέρηση της έναρξης των διαπραγματεύσεων λογικά άλματα που αποτυπώνεται εμέσως και στην συμβαστική τροπολογία 2, όπου γίνεται έκκληση προς το Συμβούλιο να ορίσει ημερομηνία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων χωρίς παραπέρα καθυστέρηση, προκειμένου να μην χαθεί το momentum, ώστε να ενισχυθούν οι κεκτημένες μεταρρυθμίσεις και διαδικασίες εκδημοκρατισμού. Κύριε συνάδελφοι, πολιτικές εκτόσεων στις βασικές αξίες και αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολιτικές δύο μέτρων και δύο σταθμών, ανάλογα με τα στρατηγικά συμφέροντα ορισμένων χωρών και συμφερόντων που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το δημοκρατικό ιδεώδες, ούτε με τις δημοκρατικές αρχές, είναι αυτές που υπονομεύουν την αξιοπιστία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διεύρυνση. Κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά, ώστε να γίνει κατανοητό από όλους, Πώ το ονοματολογικό δεν αποτελεί γενικά και αφηρημένα ένα διμερέ ζήτημα μεταξύ τη Ελλάδα και τη Φύρων, όπω θέλουν ορισμένοι εδώ μέσα να παρουσιάζουν και όπω αποτυπώνεται για παράδειγμα στι συμβαστικέ τροπολογίε 2 και 4, αλλά ένα διεθνέ, ανοιχτό ζήτημα που ο μόνο δρόμο για την επίλυσή του είναι η συνέχιση διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται υπό την ηγίδα του ΟΗΕ. Με πράξει και δηλώσει που επηρεάζουν αρνητικά τι σχέσει καλή γειτονία και οι οποίε βρίσκονται σε έξαρση συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών επίλυσης των νοματολογικού και να σας θυμίσω την φωτογράφηση του Αντιπροέδρου της Βουλής και τέος Υπουργού Εξωτερικών κ. Μιλοσόφσκη στην κορυφή του Ολύμπου, στη χώρα μου δηλαδή, κρατώντας παλιά σημαία της χώρας που φέρνει τον ήλιο της Βεργίνας, το μόνο που καταφέρνουν είναι να υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την περιφερειακή συνεργασία, τα οποία είναι και τα βασικά προαπαιτούμενα της ενταξιακή διαδικασίας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η διατήρηση καλών σχέσεων γειτονία, καθώ και η εξέβρεση αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα του ονόματο ή την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, παραμένει αναγκαία για την ενταξιακή διαδικασία τη χώρα. Η επιβράδευση λοιπόν τέτοιων πρακτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, υποδαβλίζει και την εθνικιστική φρενίτιδα που επικρατεί στη χώρα, αλλά και συντηρεί την δυσμενή κατάσταση της χώρας που περιγράφει το ψήφισμα. Επιτρέπει δηλαδή στην πολιτική ελίτ της Φύρομ να επενδύει στην επινόηση της παράδοσης, να αντιστρατεύεται τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ένωμης τάξης και να αγνοεί την έλλειψη προόδου στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σακοράφα. Και τώρα... able uh, be... Ζητώ συγγνώμη, ο κύριος ε, δεν ε, ήμουν παρόν ε, για να ακούσω τον εισηγητή. Ήμουν σε άλλη συνεδρίαση για συμβιβαστικέ τροπολογίες. Πρέπει να πω ότι η συνεδρίαση των σχεδόν εισηγητών ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και παραγωγική για τις συμβαστικέ τροπολογίες και θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το τελικό κείμενο που έχει συμπεριλάβει τις συμβαστικές τροπολογίες. Κοιτάξτε, θέλω να πω το εξής δεν αφορά ε, ε, το τμήμα του ψηφίσματος ε, ή ε, τις συμβαστικές τροπολογίες αλλά και το γεγονός και μόνο ότι είναι ασταθής η κατάσταση στη Μακεδονία μπορεί να οδηγήσει στην αναβολή της συζήτησης και του ψηφίσματος. Όπως έχουν σήμερα τα πράγματα το συμβαστικό κείμενο είναι κάτι το οποίο θεωρούμε θετικό, λογικό και θα μπορούσαμε να δεχτούμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μέσεριτς. Και τώρα Ευχαριστώ και για τη συντομία σας. Θα παρακαλούσα δύο λεπτά ο καθένας για να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι και να συνοψίσει πριν τις πέντε ο εισηγητής. Ο κύριος Καστάλτο. Ευχαριστώ. Σύντομα. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά για να μπορέσει να καταλήξει και σε ένα καλό συμβιβασμό προκειμένου και πάλι να ε, αναφερθούμε στο εγγενές πρόβλημα που είναι το θέμα της ονομασίας ε, της φύρων. Σε σχέση τώρα με τη συμβιβαστική τέσσερα. Εγώ προσωπικά θα την υπερψηφίσω. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να φτάσουμε στο άνοιγμα των διαπραγματεύσεων και μάλιστα να προσπαθήσουμε να λυθεί αυτό το διμερές ζήτημα το συντομότερο για να μην είναι τον ιωστό εμπόδιο και η νοιαστή πρόφαση για να παραμείνουμε στο τέλμα και στην παράλυση. Φυσικά είναι πολύπλοκη κατάσταση, να μην ξεχνάμε και τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά και το υποκοτάζ ε, των κοινοβουλευτικών εργασιών ε, και επίσης ε, τα όσα συνέβησαν με τις αποκαλύψεις για τις υποκλοπές Επίσης θα ήθελα να εκφράσω και την εκτίμησή μου σε ό,τι αφορά τις συμβαστικές 13 και 14 σε σχέση με την ελευθερία του τύπου. Σίγουρα θα πρέπει να γίνουν βήματα προς τα μπρος και για το σημείο 14 σε ό,τι αφορά την ισχυρή ανάγκη να υπάρχει ανεκτικότητα προς την κοινότητα των Ρωμά και των ΛΟΑΔΕΤΗ. σε ευχαριστώ ε, και το συνάδελφο που είναι ανοιχτό στον εδικτή και τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τις υπόλοιπες ομάδες. Ευχαριστώ το συνάδελφο. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Πιτίδιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχάς θα ήθελα να σας παρακαλέσω Ε, καταρχάς θα ήθελα να σας παρακαλέσω ότι εφόσον ομιλείτε με το θεσμικό σας ρόλο του Προέδρου της Επιτροπής να αναφέρεστε στη, στην ΦΥΡΟΜ με το όνομα το οποίο διεθνώς μέχρι στιγμής ε, είναι αποδεκτό ως ΦΥΡΟΜ και όχι ως Μακεδονία ένα όνομα το οποίο όπως γνωρίζετε πολύ καλά ε, θίγει και προσβάλλει την Ελλάδα και με δύο λόγια θα σας το πω αμέσως γιατί. Πριν πω αυτό θα ήθελα να παρατηρήσω ότι το, η μη συμφωνία για την ονομασία της Φύρων χρησιμοποιείται ως πρόσχημα και όχι ως πραγματικό γεγονός της μη πρόοδου των ενταξιακών σχέσεων της χώρας αυτής. Γνωρίζετε πολύ καλά και αναφερθήκατε όλοι σε αυτό ότι η χώρα αυτή δεν πληρεί τα κριτήρια της Κοπενχάγης και κατά συνέπεια ε, νομίζω ότι είναι μεγάλος βαθμός υποκρισίας να λέμε ότι εμποδίζει η Ελλάδα την ένταξη της χώρας αυτής. Η χρησιμοποίηση του ονόματος Μακεδονία δεν είναι μόνο προσβολή της ιστορίας. Εκφράζει και επεκτατικές τάσεις της φύρων κατά της Ελλάδος. Λέγεται επισήμως ότι αυτή είναι ένας ξεχωριστός λαός, ο μακεδονικός λαός, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, ένα τμήμα του οποίου, το νότιο τμήμα, είναι υπόδουλο στην Ελλάδα και πρέπει να απελευθερωθεί. Αυτό λοιπόν δείχνει επεκτατικέ τάσει, και αν πραγματικά θέλετε να λυθεί το πρόβλημα και το θέμα του ονόματος μπορείτε να ασκήσετε πιέσει προς την πλευρά τη ΦΥΡΟΜ. Συνεπώς το θέμα αυτό δεν είναι διμερές, είναι διεθνές και θέλω να πιστεύω ότι αν η χώρα η δική σα αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα δεν θα δεχόταν μια συμβιβαστική λύση ούτε θα δεχόταν να υποχωρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια και όλα τα υπόλοιπα είναι υποκρισία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Πιτίδη, η ε, Κροατία αναγνωρίζει τη Μακεδονία ως δημοκρατία της Μακεδονίας και ως Ευρωβουλευτής θα την ε, ε, αποκαλώ όπως την αναγνωρίζει και αποκαλεί η χώρα μου. Παρακαλώ. Τη δική μου φωνή με τις διαπιστώσεις οι οποίες έχουν γίνει από την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια της Συνεργασίας στην Ευρώπη αλλά και από την Κοινή Διακοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Φύρων. Και αυτές οι διαπιστώσεις λένε κάτι απλό ότι η χώρα έχει οπισθοδρομήσει τους, τους τελευταίους 12 μήνες σε όλους τους τομείς προτεραιότητας που έχουμε βάλει. Και αυτοί είναι τα πολιτικά κριτήρια, οι σχέσεις καλή γειτονία, το θέμα του ονόματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνει οπισθοδρόμηση κυρίως στους τομείς της ελευθερίας έκφρασης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία της Ευρώπης διαπιστώνει αύξηση της πολιτικοποίησης των κρατικών θεσμών, του κυβερνητικού ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και στο πλαίσιο της διαδικασίας των εκλογών. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Ζάεφ, αφού έχασε τις εκλογές, δεν έχει επιστρέψει ακόμα στα έδρανα του Κοινοβουλίου και μάλιστα πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να σχηματίσει σκιώδη κυβέρνηση και σκιώδες κοινοβούλιο. Στις σχέσεις τώρα καλής γειτονίας. Η χώρα των Σκοπίων, η Φύρομ, δείχνει τάσεις αλυτρωτισμού. Σας τα είπαν και άλλοι συνάδελφοι για μνημεία στο Γευγελί, στο Γαζί, για Μεγάλη Μακεδονία, προκλητικές ενέργειες σε γειτονικέ χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Βουλγαρία. Κάτω από αυτές τις συνθήκε. Η ΦΥΡΟΜ δεν είναι έτοιμη για ένταξη στι ευρωπαϊκέ οικονομικέ κοινότητε και για ένταξη ενταξιακή διαπραγμάτευση για τη χώρα αυτή. Όσο αφορά τι τροπολογίε, ακούστηκαν πάρα πολλά, Έχει γίνει, έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα. Κάποιε από αυτέ τι τροπολογίε, τι κοινέ τροπολογίε, θα τι υπερψηφίσουμε. Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο εισηγητή την τροπολογία νούμερο 5 να διαγράψει με δικιά του πρωτοβουλία την ε, λέξη Μακεδόνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κεφαλογιάννη. Το λόγο τώρα έχει. Από το Σιέρα συνάδελφος Τζαμπάσκι. Благодаря ви, господин председател. колеги, Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. έχουν υποθεί πολλά για την έκθεση αυτή, έχουν γίνει πολλά και βλέπω σε κάποιες συμβαστικές ε, προτάσεις και δικές μας τροπολογίες. Στην 8 και στην 11 συμβιβαστική συμπεριλάβατε και τις θέσεις της ομάδας μας. Για να ε, πω όμως ότι εμείς κάναμε προτάσεις, αλλά όχι για θέματα ιστορικά που ανάγονται στο παρελθόν. Εμείς μιλήσαμε ακριβώς για τη σημερινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Πρόκειται για διάφορα μίση, για διάφορα... Ε, ε πώς να το πω, διάφορες καταστάσεις που αποκλείουν ε, από ολόκληρα τμήματα του πληθυσμού τη χρήση της μετρικής τους γλώσσας κτλ. Αυτά θα έπρεπε να είχαν ε, εκφραστεί στο κείμενο, γιατί αν τα παραγνωρίζουμε ή τα παρακάμπτουμε δεν λύνουμε κανένα πρόβλημα. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους συναδέλφους και τον εισηγητή ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη συμβαστική 4 που γίνεται λόγος για τις διμερείς σχέσεις να κάνουμε χωριστή αναφορά σε ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο. Αυτό το, το είχα προτείνει στην τροπολογία 147 και θεωρώ ότι θα ήταν σκοπιμότερο και προτιμότερο για όλους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Εδώ ολοκληρώνεται ε, ο κατάλογος με τις εξής συναδέλφους, ε, Πετήρ, ε, Σπυράκη, Κούκαν και ο τελευταίος ο εισηγητής και κλείνω τον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι μέλος της Επιτροπή Αντιπροσωπείας για τι σχέσει ε, με τη Μακεδονία. Θερίζω τις ε, τροπολογίες που μας καλούν να προσδιορίσουμε την ημερομηνία των διαπραγματεύσεων, γιατί η Μακεδονία πραγματικά το δικαιούται. Το ψήφισμα επίσης ε, αναφέρει ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, τι έχουμε εντοπίσει και σίγουρα θα πρέπει να επιληθούν. συνεργαζόμαστε και με τους συναδέλφους από τις διεθνείς ε, αποστολές και γι' αυτό έχω καταρτήσει κάποιες τροπολογίες. Θα ήθελα να επιδοκιμάσω την ε, Μακεδονία γιατί είναι από τις ε, χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις προβλέπεται ανάπτυξη 3,8% σε ό,τι αφορά τις υποψήφιες προς τα χώρες. Κάτι το οποίο αναφέρεται είναι και οι προσπάθειες των μακεδονικών αρχών για τη στήριξη των αρχών σε ό,τι αφορά την προστασία της οικογένειας, του γάμου και της ζωής. Εξαιτίας αυτής της ε, διμερούς διαφωνίας ε, με την Ελλάδα για την ονομασία, η Μακεδονία περιμένει την έναρξη των διαπραγματευτικών διαδικασιών εδώ χρόνια. Και αυτό ε, διακινδυνεύει τη μεθοδολογία τη όλη αυτή τη υπόθεση θέτει σε κίνδυνο και υπονομεύει το, την ευρωπαϊκή πορεία της Μακεδονίας. Γι' αυτό θα θέλαμε να καλέσουμε τους πάντες να επιλέξουν την ε, προσέγγιση των βέλθων πρακτικών, όπως έγινε και με τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία και επιγόντως να βρεθεί λύση, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Μακεδονία και τα διμερεί ζητήματα να επιληθούν με βάση και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σπυράκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα το οποίο βλέπουμε και τοποθετούμε ως μέλος της Επιτροπής των Σχέσεων της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει σοβαρές και θεμελιώδεις αντιφάσεις. Καταγράφει και μάλιστα πολύ αναλυτικά μια σειρά παραβιάσεις, μια σειρά γκρίζες ζώνες σε πολύ βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι χώρες που ξεκινούν τις συνταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων ή των άλλων εθνοτήτων, γιατί θέλω να θυμίσω ακριβώς την πληθυσμιακή αναλογία των Αλβανών με τους ε, ε σλαβόφωνους που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, το σεβασμό των ελευθεριών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, τις σχέσεις κράτους κυβερνώντος κόμματος, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και αυτά είναι μόνο κάποια. Ποιο θα είναι ο μοχλός πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ώρα που θα δώσουμε ημερομηνία έναρξης διαπραγματεύσεων με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ώστε να έχουμε να κάνουμε με ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος, με ένα κράτος στο οποίο η δημοκρατία λειτουργεί. Δεν δίδεται απάντηση σε αυτό το ψήφισμα. Αντιθέτως, αποδίδεται μόνο στη διαφορά με την Ελλάδα, ο λόγο για τον οποίο, ενώ εδώ και 9 χρόνια η πρώην Ιγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία έχει λάβει καθεστώ υποψήφια χώρα δεν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσει. Οι λόγοι είναι πολλοί, είναι ουσιοδέστεροι και σε καμία περίπτωση δεν αφορούν τη διαφορά με την Ελλάδα. Θέλω όμω να θυμίσω εδώ ότι η Ελλάδα από το 2008 και μέχρι σήμερα και με τη νέα κυβέρνηση κρατά μια σταθερή στάση κάνοντας το μισό του δρόμου του συμβιβασμού. Έχει ήδη προτείνει μια σύνθετη ονομασία μία ονομασία έναντι όλων, έργα όμνες, προς την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και περιμένει απάντηση που ποτέ δεν ήλθε. Το τελευταίο είναι ότι επίσης θα ήθελα να θυμίσω και προς τον εισηγητή ότι η επίσημη ονομασία είναι πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ΦΥΡΟΜ, ως τέτοια υπογράφει η χώρα αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση την συμφωνία για να λάβει καθεστώς υποψήφιας χώρας. Ως εκ τούτου τουλάχιστον ας σεβαστούμε τα, τα υπάρχοντα, τα κεκτημένα, τα γραμμένα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Ορισμένε παρατηρήσει. Πρώτον, σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση στη χώρα ε, που έχει κάνει μία δραματική μεταβολή τις τελευταίες εβδομάδες και δεύτερον ότι αφορά το μέλλον. Εγώ παρακολουθώ την εξέλιξη της χώρας εδώ και πολλά χρόνια μαζί με άλλους συναδέλφους και στηρίζουμε τις ευρωπαϊκές της φιλοδοξίες. Με προβληματίζει ιδιαίτερα επομένως ε, με προβληματίζουν ε, οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, δυστυχώς, ε, το πολιτικό τέλμα σε αυτή την κατάσταση έχει προχωρήσει σε ε, πολιτικές διαφωνίες, σε σημαντικές συμμαχίες στο πολιτικό βίο της χώρας σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό της σύστημα και υπονομεύουμε και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική σκηνή διαφαίνεται και αποτυχία των ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών στο πολιτικό σύστημα και θα πρέπει λοιπόν να διαρευνηθούν καταλήλως από ανεξάρτητους φορείς αυτά τα δεδομένα. Όμως, σε ό,τι αφορά την... και η αντιπολίτευση θα πρέπει ε, να δράσει υπεύθυνα, όμως θα ήθελα να τους παρακαλέσω να απόσχουν από τυχόν ε, ακραία μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα την σημερινή συζήτηση προ του αγαπημένου και αγαπητούς μάλλον ε, και διακεκριμένου Έλληνε συναδέλφου, λένε ότι η χώρα δεν πληρεί τα κριτήρια τη Κοπεχάγη. Θα ήθελα να του υπενθυμίσω με κάθε ταπεινότητα ότι αυτό το ψήφισμα έχει προετοιμαστεί βάσει τη έκθεση προόδου που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφέρει ότι η χώρα πληρεί τα κριτήρια της Κομεχάγης και συστήνει την έναρξη ε, των διαπραγματευτικών διαδικασιών. Εδώ στο Κοινοβούλιο απλώς στηρίζουμε αυτή τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, Έντουαρτ. Πριν δώσουμε το λόγο και ε, πάλι στον εισηγητή, τον κύριο Βάγκελ, να δώσουμε το λόγο σε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Πόρτιου, αν κατάλαβα καλά, θα λάβει το χώρο, Το λόγο σου νόμι, είναι Μεγάλη πρόκληση αυτός ο φάκελος για τον Επίτροπο Χάν και ελπίζουμε στο τέλος της πενταετού θητείας να έχουν σημειωθεί σημαντικές επιτυχίες ό,τι αφορά την, το φάκελο τη Μακεδονίας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα γνωρίζετε ότι ο Επίτροπος Χάν έκανε την πρώτη επίσκεψη στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας την περασμένη Τρίτη και εξέφρασε τι σοβαρέ ανησυχίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, καλώντας όλα τα πολιτικά μέρη, τους παράγοντες να μπουν σε έναν επικοδομητικό διάλογο μέσα στο Κοινοβούλιο με ε, έμφαση στις στρατηγικές προτεραιότητες για τη χώρα και τους πολίτες. Και ε, μάλιστα προσέφερε την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας υπόψη την πολύ επιτυχημένη αποστολή της Επιτροπής του Κοινοβουλίου σας στην Αλβανία, εάν τα εμπλεκόμενα μέρη στη χώρα θεωρούν αυτό ότι είναι χρήσιμο για να εγκαθιδρυθεί ο πολιτικός διάλογος μέσα στο Κοινοβούλιο και περιμένει αντιδράσεις από τα κόμματα και τις πολιτικές ομάδες της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το θέμα αυτό και θα σας στηρεί ενήμερους για την απάντησή τους. Εν ώψη λοιπόν της κρίσης αυτής, ο Επίτροπος Χάν υπενθύμησε σε όλους τους συνομιλητέ ότι το κράτος δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η ελευθερία των μίντια του τύπου είναι στην καρδιά της ε, προενταξιακή διαδικασία. και εξέφρασε τι ε, βαθιές του ανησυχίε σε σχέση με, τις, ε, με τους ισχυρισμούς για την παρακολούθηση χιλιάδων πολιτών και ζητά αυτά να διερευνηθούν επισταμένω και ενδελεχώ και θα πρέπει οι έρευνες να γίνουν με πλήρη αμεροληψία, με διαφάνεια, με διαχωρισμό εξουσιών, με ανεξαρτησία του δικαστικού ε, κλάδου, της δικαιοσύνης. Παρόλες αυτές τις δυσκολίες θα ήθελα να ολοκληρώσω τη σύντομη παρέμβασή μου επαναλαμβάνοντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι σημαντικό η χώρα να προχωρήσει στην ευρωπαϊκή της πορεία. Επιτρέψτε μου κυρία Σακοράφα να σας πω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαμηλώσουμε τα σημεία αναφοράς και θα ε, επαναλαμβάνουμε την έκτη χρονιά συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ότι δηλαδή η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ικανοποιεί παρκώς τα κριτήρια για την έναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων. Χωρίς σαφή και αξιόπιστη προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κίνδυνος ουσιαστικής οπισθοχώρησης και οπισθοδρόμησης. Και ενδεχομένως αυτό εξηγεί όλα αυτά που έχουμε δει ή εν μέρει αυτό που έχουμε δει τους τελευταίους 12 μήνες. Θα πρέπει εμείς να ε, ασκήσουμε πίεση ακριβώ για να προχωρήσει η χώρα προς τα εμπρός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος η ηγητής μας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω όλους όσοι έχουν συμβάλει ε, σε αυτή τη συζήτηση η οποία έγινε με τις καλύτερες προθέσεις και για σωστό σκοπό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι απήχαν από, τις, ε, την υιοθέτηση μιας ε, λεκτικής υπερβολής αν θέλετε έτσι ώστε να έχουμε μία ε, σωστή συζήτηση στα κοινοβουλευτικά πλαίσια. Ξέρετε, ε, τα άσπρα μαλλιά που έχω στο κεφάλι μου ενδεχομένω μου δίνει το δικαίωμα να εκφράσω και επιθυμίες. Ότι δηλαδή όλες οι γειτονικές χώρες να ε, ζουν εν ειρήνη μέσα σε αμοιβαίο σεβασμό. Και είμαι βέβαιος μάλιστα ότι μια σταθερή Μακεδονία είναι μια ανοιχτή Μακεδονία, μια Μακεδονία η οποία θα είναι ανοιχτή στα συμφέροντα της Ελλάδας και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή στιγμή να δηλώσουμε τις προσδοκίες μας. Προσδοκίες για αλληλεγγύη έναντι της Μακεδονίας, όπως άλλωστε έχουμε δείξει και αλληλεγγύη και σε άλλες χώρες που παίρνουν δύσκολες στιγμές. Έχουμε εκφράσει και πολύ αλληλεγγύη ε, προς την Ελλάδα και σωστά και καλώς. Και με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Διακεκριμένοι συνάδελφοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον και να οικοδομούμε την Ευρώπη επί τη βάση της πολιτικής καλής γειτονίας και ε, αμοιβαίας κατανόησης. Και αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους ε, λόγους για τους οποίους ασκούμε κριτική σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, ασκούμε κριτική στις ε, διαστάσεις που εντοπίσαμε στη Μακεδονία που δεν, πληρούν, που δεν συνάδουν πλήρως με το κράτος ε, δικαίου π.χ. μεταξύ άλλων και νομίζω ότι η έκθεση και η κάθε έκθεση αυτά ακριβώς αποσκοπεί να βελτιώσει και να διορθώσει και για να το κάνει βασίζομαι στη στήριξή σας. Ε, υπάρχουν οι προτάσεις που έχετε υποβάλει με τη μορφή τροπολογιών. Στο βαθμό που είναι εφικτό αυτό θα προσπαθήσω ε, να ε, βελτιώσω αυτό το κείμενο. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση σήμερα δείχνει ότι η έκθεση θα τύχει αρκετή στήριξη. ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος και εγώ ευχαριστώ. Βεβαίως και στηρίζω την επικοδοματική σας προσέγγιση ως προς τη Μακεδονία και τη λύση δηλαδή του να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις και μετά να επιληθεί το θέμα της ονομασίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση. Νομίζω ότι το επίπεδο ματέωσης ε, το οποίο βιώνει ε, αυτός ο λαός αυτή τη στιγμή είναι κάτι που καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι εδώ. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε τώρα το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ε, ε, ενωσιακή ενταξιακή διαδικασία για το κοσφοπέδιο, έχουμε έκθεση από την κυρία Λούνατσεκ, η οποία είναι εδώ, η συγγήτριά μας. Το 2014 ήταν δύσκολη χρονιά γιατί υπήρξε πολιτικό τέλμα μετά τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές του Ιουνίου, κάτι το οποίο είχε αποτέλεσμα σε επίπτωση σε όλες τις διαδικασίες τις συνταματικές. Από τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο του 2014 έχει αρχίσει το νομοθετικό έργο και στις 9 Φεβρουαρίου ξαναξεκίνησε ο διάλογος υψηλού επίπεδου Πρίστινας Βελιγραδίου. Υπήρξε συμφωνία για το δικαστικό σώμα, για τη δικαιοσύνη, ωστόσο παραμένουν πολλά να γίνουν. Αυτό το λέει και η έκθεση και οι 212 τροπολογίες που υποβλήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής μας. Έχουμε 15 στις συμβιβαστικές ε, τροπολογίες που ε, έχουν τυχεί συμφωνίες μεταξύ εισηγήτριας και σκιωδών εισηγητών. Να δώσω το λόγο στην κυρία Λούνατσεκ για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές για την εξαιρετικά καλή τους προετοιμασία και μάλιστα να ευχαριστήσω τους καινούριους σκιώδεις εισηγητές τους οποίους δεν γνώρισα, όπως ο κύριος Παντσέρη ε, χάρηκα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Νομίζω ότι βρήκαμε ένα καλό τρόπο να μπούμε σε, να περιλάβουμε επαρκείς και αρκετές συμβιβαστικές λύσεις ε, τις οποίες πρότειναν πολλοί συνάδελφοι από όλες τις πολιτικές ομάδες, από όλο το πολιτικό φάσμα γιατί η βούλησή μας ήταν να δείξουμε ότι πραγματικά θέλουμε και μπορούμε να συνεργαστούμε. Ξέρω και γνωρίζω ή μάλλον πριν πω αυτό, θα ήθελα να πω κάτι άλλο που έχει να κάνει περισσότερο με τις μεταφράσεις. Κατά τη διάρκεια της δουλειάς μας εκεί είδαμε δύο σημεία όπου η μετάφραση ήταν εσφαλμένη σε σχέση με την πρωτότυπη εκδοχή του κειμένου στα αγγλικά. Η πρώτη έχει να κάνει με την πρώτη παράγραφο, όπου το πρωτότυπο κείμενο λέει ότι καλωσορίζει το γεγονός ότι έχει τελειώσει το εξάμεινο πολιτικό τέλμα και το καθεξής, το εξάμεινο τέλμα και εν περιπτώσει έχει συγκροτηθεί το κοινοβούλιο σε σώμα και στα γαλλικά λέει καλωσορίζουμε τη συγκρότηση του Κοινοβουλίου και τον ορισμό αν θέλετε της νέας κυβέρνησης που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα για να μην πω ότι είναι και τελείως διαφορετικό γιατί εμείς λέμε ότι καλωσορίζουμε όχι το ότι υπάρχει ναι, κυβέρνηση εμείς καλωσορίζουμε ότι άρθηκε το αδιέξοδο, το τέλμα και μετά στην τροπολογία 51 του Γιάννης Νέλσον από την ΚΟΕΣ σε γενικές γραμμές και δεν ξέρω αν το πρωτότυπο ήταν στα σουηδικά, στα αγγλικά ε, λέει ότι παρόλο που τονίζει την ανάγκη να βρεθεί λύση και ούτω καθεξής, ε, και δεν θα πρέπει να λέει παρόλο, although, θα έπρεπε να λέει also, επίσης. Επομένως, ζητώ από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, το δει το θέμα με αυτές τις δύο λάθος μεταφράσεις, γιατί δεν ερμηνεύεται σωστά το νόημα. Αυτά λοιπόν για τη μορφή Α έρθω τώρα στο περιεχόμενο. Έλεγα λοιπόν ότι εκτιμώ ιδιαίτερω για το γεγονό ότι είχα πολύ καλή συνεργασία με του σκιώδει εισηγητές και θέλω να το πω για, τη συγκεκριμένη, για το Κόσοβο, για το Κοσφοπέδιο, διότι έχουμε μέλη στην Επιτροπή μα που δεν στηρίζουν την ε, θέση που έχει κατά πλειοψηφία υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν, το οποίο έχει ταχθεί υπέρ τη ανεξαρτησία του Κοσφοπεδίου ότι είναι δημοκρατία και ανεξάρτητο κράτο. Βεβαίως πάρα πολλές τροπολογίες δεχτήκαμε από μέλη που δεν υιοθετούν αυτή τη θέση και που ε, ζητούν να μην μιλούμε για κυβέρνηση, για κράτος, για χώρα και πάντοτε να περιλαμβάνουμε το ψήφισμα 1244 ε, των Ηνωμένων Εθνών και όλες αυτές τις τροπολογίες όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να τις περιλάβω και στον κατάλογο ψηφοφοριών η πρόταση είναι αρνητική. Υπάρχει πρόταση καταψήφισης τους και αυτό ε, δεν είναι κάτι που μπορώ να δεχτώ, δηλαδή δεν μπορώ να βρω συμβαστική λύση ε, ως προς την πρόταση αυτή. Όχι μόνο διότι είναι η δική μου θέση αυτή, αλλά διότι αυτό έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τότε που ανέλαβα ε, το θέμα αυτό, από το 2010. Ζητούμε λοιπόν από τους πέντε που δεν αναγνωρίζουν να αναγνωρίσουν και το καθεξής. Όλα αυτά θα έχουμε ψήφιση για όλα αυτά τα θέματα αύριο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Τώρα, μπορέσαμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις ως προς την πρόοδο, την οποία σημειώνουμε, που έχει σημειώσει το πέδιο την τελευταία χρονιά για ορισμένα ζητήματα και επικρίνουμε κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει λόγω του εξάμεινου ε, τέλματος ή ε, αδιεξόδου. Και καλωσορίζουμε το γεγονός ότι ξαναξεκίνησε ο διάλογος στις 9 Φεβρουαρίου, ε, με ομαλό τρόπο, από ό,τι φαίνεται έχει γίνει μια κάποια δουλειά καλή βλέπουμε την κατάσταση στο κοσμοπηδίο και λέμε ότι χρειάζεται βελτίωση εκεί, αλλά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει. Εκφράζουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι η διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα είναι διαδεδομένα, η κατάσταση σε σχέση με τα δικαιώματα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει με τη Συμφωνία ε, Σύνδεσης Σταθεροποίησης και προβάλλουμε το εξής επιχείρημα, ότι δημιουργούνται προβλήματα για τους πολίτες του Κοσφοπεδίου, με ε, τους πέντε που δεν αναγνωρίζουν, όχι μόνο πολιτικά, αλλά σε θέματα πολιτισμού, σε θέματα αθλημάτων. Π.χ. αν σας αρέσει ο διαγωνισμός της Eurovision, δεν αρέσει σε όλους, αλλά σε πολλούς αρέσει και οι νέοι θέλουν να συμμετάσχουν. Και οι καλλιτέχνες του Κοσφοπεδίου δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό της ε, Eurovision, γιατί το Κοσφοπέδιο δεν το αναγνωρίζει η EBU. Ή στον τομέα των αθλημάτων, η FIFA πολύ πρόσφατα επέτρεψε η ομάδα του Κοσμοπεδίου Υποδοσφαιρική να παίξει φιλικά και όχι επίσημα ε, παιχνίδια, αγώνες με άλλα. Νιώθουν λοιπόν αποκλεισμένοι οι πολίτες του Κοσμοπεδίου και είναι και η μόνη χώρα στην περιφέρεια, στην περιοχή όπου οι πολίτες συνεχίζουν να μην μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα για τρεις μήνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητούμε λοιπόν απελευθέρωση των θεωρήσεων Ζητούμε από το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση του Κοσφοπεδίου να προχωρήσουν τα πέντε ε, νομοθετήματα, νομοθετικά πακέτα που ε, παραμένουν και ζητούμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να προχωρήσουν προς τα εμπρός και να διασφαλίσουν ότι θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πολίτες του Κοσφοπεδίου. Εάν υπήρχε αυτή η απελευθέρωση από την υποχρέωση θεώρηση, δεν θα είχαν φύγει τόσοι πολλοί Κοσοβάροι από τη χώρα ε, του τους τελευταίους μήνες. Αν δεν υπήρχαν θεωρήσεις θα μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιστρέψουν, ε, όπως κάνουν άλλοι πολίτες της ε, περιοχής. Δεν είχαμε μαζική μετανάστευση από τις γειτονικές χώρες, κάτι που φοβόντουσαν ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αλλά δεν είχαμε από τις γειτονικέ χώρες μαζική μετανάστευση όταν ε, ήραμε την υποχρέωση για θεώρηση, για βίζα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ισχυρισμοί ε, διαφθοράς μέσα στη Ulex. Το αναφέρουμε. Αναφέρουμε ότι η Ulex έχει κάνει σημαντική δουλειά στο κοσφοπέδιο, αλλά αναφέρουμε και το στραβό εντό εισαγωγικών. Και ελπίζουμε ότι θα διευκρινιστούν θα ε, διαλευκανθούν αυτές οι, αυτοί οι ισχυρισμοί, οι κατηγορίες και θα μπορέσει η Γιούλεξ να συνεχίσει το έργο της. Τώρα, ως προς την λάθρο μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση ε, το τελευταίο ένα με δύο μήνες από πλευράς πολιτών κοσφοπεδίου που περνάνε αμέσα από τη Σερβία για να ζητήσουν άσυλο στην Ουγγαρία ή στη Γερμανία και ούτω καθεξής. Έχω ένα στοιχείο που θέλω να υποβάλω αύριο στο συνάδελφο κύριο Μακάλιστερ, γιατί θέλω να μπει ως τροπολογία και στην έκθεση για το Κοσμοπέδιο και στην έκθεση για τη Σοερβία. Μόλις τελειώσω και μόλις κλείσω το μικρόφωνο κύριε Μακάλιστερ θα έρθω να σας βρω για να σας παρουσιάσω αυτή την προφορική τροπολογία που θέλω να σας προτείνω. Θέλω να καλέσουμε όλες τις αρχές να ενισχύσουν τη συνεργασία για να εξαρθρώσουν τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης λαθρεμπόρων, δουλεμπόρων που ε, διοχετεύουν ε, τους πολίτες ε, μέσα από το κοσμοπέδιο διαμέσου της Σερβίας προς τις χώρες της Ευρώπης. Τώρα, για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, σίγουρα βλέπουμε ε, πρόοδο ως προς τα δικαιώματα ορισμένων ε, εθνοτικών μειονοτήτων, όπως είναι ε, ο σερβικής προέλευσης καταγωγής πληθυσμός του κόσυφου πεδίου. Σημειώνουμε ότι παραμένουν τα προβλήματα με τους ασκάλι, με τους Ρωμά, μεταξύ άλλων και πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες. Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει γίνει για τα δικαιώματα λεσφιών, ομοφιλοφίλων, φιλομεταβατικών κτλ. με το πρώτο Gay Pride που έγινε πέρσι. Για τα δικαιώματα των γυναικών εκφράζουμε τη θλίψη μας για το γεγονός ότι μεταξύ των 21 νέων υπουργών η νέα κυβέρνηση δεν έχει ούτε μία γυναίκα. Και κάτι που δεν είναι στην έκθεση θέλω να σας πω. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο στο μέλλον κάποια στιγμή θα θέσει θέμα ποσοστώσεων για ε, ε, να υπάρχουν γυναίκες στην κυβέρνηση. Και ε, η τελευταία μου παρατήρηση είναι η εξής. Ορισμένες από τις τροπολογίες σας ε, δεν είναι και πολύ κατανοητές σε μένα και γι' αυτό θα σας έρθω σε επικοινωνία μαζί σας για να το επιβεβαιώσω. Π.χ. το θέμα με τη Γιούλεξ, με, τη, με τους ισχυρισμούς για διαφθορά. Ε, ε, η τροπολογία 114 ή 141 λέει η ομιλήτρια αναφέρει κάποια προβλήματα αλλά ε, δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με το CPCC. Ε, ελπίζω λοιπόν να έχουμε ε, καλή ψηφοφορία αύριο και ελπίζω και να συνεργαστούμε ομαλά στο μέλλον. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούνατσεκ και φυσικά ανυπομονούμε να δούμε τον διάλογο υψηλού επίπεδου καθώς ο και το εξωτερικό τη Σερβία είναι από το δύο κράτος μέλος. Όχι. Αυστρία, συγγνώμη. Έχουμε δύο χώρες που τη δίνει μια κοινή γλώσσα. Βλέπω ότι ο κύριος Πιτσούλα δεν είναι εδώ. Επομένως, ως ε, πρόεδρος της Επιτροπής για τη Σχέση με το Κρατοπέδιο δεν θα μιλήσει. Θα δώσω το λόγο στο σκιώδη συγγητή από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριο Αντακτούσον. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την κυρία Λούνεφεκ. Σα ευχαριστώ για την έκθεσή σα. είναι πολύ καλή. Και μιλά για περαιτέρω ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και αναφέρεται και στις κύριε προκλήσει που έχει το Πρωθυπουπέδιο για το μέλλον του. Όλα αυτά είναι σαφέστατα στην έκθεσή σας. Καλωσορίζω τις διάφορες προτάσεις που έγιναν, κυρίως για ένα καλύτερο κλίμα για τις επιχειρήσεις, το καλωσορίζω αυτό. Επίσης, τη σημασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας θα πρέπει να λειτουργούν κατάλληλα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια για τα εκτιμάτα αγορά, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κοσυφοπεδίου. Χρειαζόμαστε δικαιοσύνη, σεβασμό του νόμου και καλύτερη χρήση της γης. Ένα άλλο θετικό σημείο που αναφέρεται είναι η αναφορά στην ε, εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Αυτό είναι στις Τροπολογίε και είναι κάτι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που υπάρχει εκεί για τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και σύνδεση. Είναι πολύ μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για το κοσοπέδιο και φυσικά πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία της χώρας. Και πάλι το κείμενο είναι σαφέστατο και το καλωσορίζω. Τέλο. Η έκθεση αναφέρεται και σε ένα άλλο θέμα και με πολύ σωστό τρόπο σε σχέση με τη Γιούλεξ και την έρευνα με τους ισχυρισμούς, για τους ισχυρισμούς διαφθοράς. Εγώ μάλιστα στην αρχή του έτους ήμουν στην Πρίστινα και παρατήρησα ότι συνέβαινε τοπικά και ήταν σαφές για μένα ότι είναι υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ότι ο εμπειρογνώμονας που θα ορίσει η κυρία Μογκερίνη θα προβεί σε μια αμερόληπτη έκθεση. Φυσικά αυτό είναι ένα θέμα εμπιστοσύνη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αφορά μόνο το κοσυφοπαίδιο, αλλά αφορά και τη δική μας φήμη και όλες οι χώρες μας και όλοι μας οι πολίτες ε, θα σχηματίσουν άποψη για τα Βαλκάνια από το θέμα αυτό. Πρέπει να είναι πλήρε λοιπόν η έρευνα, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα μάλλα την ευκαιρία αυτή, πρέπει να ξέρουμε τι έκανε ποιο, τι πήγε λάθο και ποιο έχει την ευθύνη. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Λούνετσεκ για την εξωτερική συνεργασία και την εξωτερική έκθεση. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αντάκτουσον. Τώρα να δώσω το λόγο στον αγαπητό συνάδελφο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια. Κύριο Παντσέρη. Οι συμβαστικές τροπολογίες ε, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό απαντούν ε, στα αιτήματα που είχαμε θέσει κι εμείς και θεωρώ ότι είναι ισορροπημένη η έκθεση συμπερασματικά. Κυρίως σε κάποια ουσιαστικά σημεία που θεωρώ πολύ σημαντικά. Όπως το να προχωρήσουμε ταχαίως, να προχωρήσει ταχαίως το στην οδό των μεταρρυθμίσεων, το ότι επιμείνεται στο ενισχυθεί το κράτος δικαίου, το δικαστικό σύστημα, την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς και το ότι υπογραμμίζεται ένα θέμα ζωτικό για τη χώρα αυτή, την ανεξαρτησία ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την αποτελεσματικότητα των δικαστών και των εισαγγελέων. Και βεβαίως φυσικά και σε ό,τι αφορά το θέμα της Ιούλεξ σχετικά με τις κατηγορίες διαφθοράς. Θεωρώ ότι το αίτημα να υπάρχει πλήρης διαφάνεια είναι ένα δίκαιο αίτημα από την πλευρά του Κοινοβουλίου και πολύ σωστά αναφέρεται στην έκθεση. Τέλος, όπως και η κυρία Λούνατσεκ και εγώ είμαι αρνητικός επί όλων των τροπολογιών που και πάλι προτείνουν ένα τέλμα, δηλαδή στο να μην γνωριστεί η χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παντσέρη. Συνάδελφος Νταμπάσκη από το ECR. Ευχαριστώ. Είμαι σκοτής εισηγητής και δεν μπορώ παρά και εγώ να συμφωνήσω με τα καλά λόγια που υπόθηκαν για την κυρία Λούνατσεκ και για τις τροπολογίες που προτάθηκαν. φυσικά έχουν ληφθεί υπόψη στις τροπολογίες όλα όσα προτείναμε. Έτσι λοιπόν την ευχαριστούμε πολύ για το έργο της. Φυσικά το κοσμοπέδιο πρέπει να καταβάλει ακόμα πολλές προσπάθειες. Υπάρχουν ε, και επαρκώς οτιολογημένες κριτικές από την πλευρά των συναδέλφων και εκφράζεται πολύ καλά η κατάσταση που υπάρχει επί τόπου. Και πάλι θέλω να συγχαρώ την κυρία Λούνατσεκ για να την ευχαριστήσω. Ευχαριστούμε. Τώρα, κυρία Βάλτμαντς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια στην κυρία Λούραντσα και η εκθεσή της είναι καλή και ισόρροπη. Δείχνει και τα θετικά και κάποια αρνητικά. Ε, τα περισσότερα θέματα ήταν στην αρχική διατύπωση, αλλά δεν θα ήμασταν πολιτικοί αν δεν θέλαμε να βάλουμε και το δικό μας στίγμα. Ε, ε, βλέπουμε ότι είναι 212 οι τροπολογίες και μεταξύ αυτών έχουμε κάνει και εμείς φιλελεύθεροι και να τονίσω τα εξής έτσι διπλωματικά να πω ότι οι περισσότερες ανησυχίες μας έχουν καλυφθεί από τις συμβαστικές. Ε, αυτό που παραμένει ε, ως θέμα τριβής για το Κωσυφοπαίδειο, είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στον πληθυσμό εκεί, ότι θέλουμε το κράτος τους να είναι βιώσιμο πολιτικά και οικονομικά στην περιοχή και μελλοντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπό την έννοια αυτή έχουμε κάνει μια τροπολογία στην αρχή του ψηφίσματος που δεν αναφέρεται ε, στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά λέει ξεκάθαρα το ίδιο πράγμα. Δεύτερον, θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους ερετούς ε, της σερβικής μειονότητας ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους δημόσια και πολιτικά. Τρίτον, ε, έκκληση στις πολιτικές αρχές να δείξουν πλήρη υποστήριξη για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δικαστών και εισαγγελέων. Τέταρτον, ε, έκκληση για ε, σε βάθος και ευρεία έρευνα των γράφων για τις αιτιάσεις διαφθοράς, τη Γιούλεξ, πράγμα που δεν είχαμε δει. Και επίσης καλούμε τις αρχές στην Πρίστινα ε, να αντιμετωπίσουν ε, τις εγκληματικές δραστηριότητες στη διακίνηση ανθρώπων με τη βοήθεια ε, των Ευρωπαίων στην Πρίστινα. Τέλος, θα σας πω με χαρά ότι η Άλτε θα υπερψηφίσει το ψήφισμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ πολύ. κύριος Καστάλτο. Καστάλτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Λούνιτσεκ για την εξαιρετική δουλειά τη στην έκθεση αυτή και κυρίως για τις συμβαστικές τροπολογίες τις οποίες κατέληξε που νομίζω ότι ε, όλα τα θέματα που τέθηκαν από διάφορες ομάδες και σε ό,τι αφορά το θέμα που μας ενδιαφέρει, σε ό,τι αφορά τη διακίνηση όπλων ε, και το ότι πρέπει να ισχυθεί συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών με τις αρχές του πεδίου. Υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό δεδομένου και της γεωπολιτικής κατάστασης. Και μεταξύ άλλων Συμφωνώ με τις ανησυχίες ε, που τέθηκαν για τη συμβαστική 10 από άλλους συναδέλφους ε, σε ό,τι αφορά την αποστολή Ιουλέξ. Ε, όχι μόνο γιατί είναι η πιο μεγάλη και δερματική αποστολή που έχει υλοποιηθεί μέχρι τώρα από την Ένωση, γιατί πραγματικά μας κοστίζει την αξιοπιστία μας σε σχέση με τις υποψήφιες χώρες. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες και εις βάθος για να διαφωτίσουμε τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης αυτής και φυσικά θα υποστηρίξουμε την έκθεση. Γιατί θεωρώ ότι έχει υλοποιηθεί με, την, με μια πολύ ισορροπημένη και διπλωματική προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σοπράτ. Merci. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά την κυρία Λόνατσα και την έκθεσή τη και για τη δουλειά τη, ακόμα και αν δεν συμφωνώ καθόλου με τα συμπεράσματα. Θέλω να θυμίσω τρία στοιχεία που θεωρώ σημαντικά για να αντιταχθώ σε αυτή τη λογική ένταξη στο Κόσοβο. Πέντε είναι τα κράτη-μέλη που δεν είναι ευκαταφρόνητο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι κατά της ανεξαρτησίας. Κάπως παράδοξο δεν είναι να μιλάς για ένταξη όταν δεν συμφωνείς για την ανεξαρτησία της χώρας. Ε, επίσης, Υπάρχει και μια ε, λογική εθνοκάθαρσης. Θυμάμαι, ε, θυμίζω 99 με 2004 ε, από 235.000 που διώχθηκαν από διάφορε μειονότητες επέστρεψαν μόνο 12.000. Αυτά δεν τα λέει η έκθεση. Και το τρίτο είναι το εγκληματολογικό στοιχείο. Οι πάντε γνωρίζουν ότι το κοσυφοπέδιο είναι αιστεία διεθνούς εγκλήματο. Ε, δηλαδή εμπόριο ναρκωτικών, διακίνηση ανθρώπων και θε να βάλεις μια τέτοια χώρα στην Ευρώπη είναι, ε, σημαίνει να θα ενταθεί η διεθνή εγκληματικότητα που αγγίζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε αντίθετοι με τη λογική τη έκθεση, ολόκληρη, ακόμα και αν καλωσορίζω τη σοβαρή δουλειά τη κυρία Λούναζε, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με τα συμπεράσματα, το αντίθετο μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω το εξή. Αυτή τη βδομάδα πήγα στη Μητροβίτσα και στην Πρίστινα δύο μέρες και ένα από τα βασικά θέματα εκεί ήταν η μασική ε, αποδημία προ τη Γαλλία, την ε, Αυστρία ή τη Γερμανία. Και στις πολιτικές συζητήσεις που είχα διαπίστωσα ότι είναι σαφή τα αίτια. Η φτώχεια, η ανεργία, ε, η ακρίβεια που αυξάνεται όλο και περισσότερο και μια ε, απεσιοδοξία, μια έλλειψη ελπίδας και γενικότερη ζωφερή κατάσταση. Ε, πολλοί κόσοβάροι όμως που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη ε, για το άσυλο πέφτουν θύματα ε, σε κάποιους διακινητές που θέλουν να βγάλουν λεφτά και ε, τους παραπλανούν μέσω διαδικτύου και τα λοιπά. Ε, και τους λένε ότι θα κάνουν αίτηση άσυλου χωρίς να έχουν την παραμικρή δυνατότητα να πάρουν ε, άσυλο. Φεύγουν από τη χώρα, πουλάνε τα σπίτια τους, ε, όλο τους το βιός και μετά όταν αναγκάζονται να επιστρέψουν είναι απελπισμένοι. Καλωσορίζω το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι όσοι θέλουν να επαναπατριστούν θα ενσωματωθούν το συντομότερο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιταχύνει τις διαδικασίες. Αλλά σημασία έχει ο κόσμος να τα ξέρει αυτά πριν φύγει. Ο δρόμος του ασύλου είναι αδιέξοδο κατά κανόνα και θα πρέπει να τονίσω αυτό που είπε και η κυρία Λούνατσεκ. Τελικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Κόσοβο ε, ε, πρέπει να έχει μια οικονομική ε, προοπτική να προσελκύσει ξένους επενδυτές που χρειάζονται ασφάλεια ε, και σταθερότητα και η πηγή όλων των κακών και των δεινών είναι η διαφθορά. Ευχόμαστε σε αυτή τη μάχη καλή επιτυχία στην κυβέρνηση στην Πρίστινα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μακάλιστε. Πραγματικά ε, είναι πολύ οξύ αυτό το πρόβλημα των τελευταίων εβδομάδων, πολύ σωστά το αναφέρατε, και η οικονομική κατάσταση και γενικότερη η προοπτική και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών του Κωσόβου. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον επικεφαλής ε, της Αντιπροσωπείας για σχέση με το Κόσοβο, τον κύριο Πίτσουλα που μόλις έφτασε και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για να ολοκληρώσει η συνάδελφος από την Αυστρία λοιπόν η κυρία Λούνατσε. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση, ιδίω δεδομένου και το ότι το έγγραφο αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίσει ε, τη δυναμική των τελευταίων μηνών. Εδώ αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στη μετανάστευση που επιβαρύνει και επιδρώνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απαντήσει καταλήλως ε, και πολύ ορθώ ε, σε αυτή την κατάσταση μέσω τη έκθεση της κυρίας Λούνατσεκ. Η μετανάστευση ε, βρέθηκε στο πρώτο σέλιδο του ευρωπαϊκού τύπου και μπορεί να αποτελεί και αποτέλεσμα της ανεπαρκούς και καθυστερημένης απάντησης από τις αρχές του κοσμοπεδίου. Από την άλλη όμως είναι και απόρρια της έλλειψη προοπτικών και της απεσιοδοξία που αισθάνονται όχι μόνο οι νέοι ε, του κοσμοπεδίου αλλά και άλλοι. Ιδίω όμως οι νέοι δεν βλέπουν μέλλον, δεν βλέπουν προοπτική στο κοσμοπέδιο. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επίση διαδραμάτισαν ένα ρόλο με την αντίδρασή του και σε ό,τι αφορά την πολιτική διεύρυνση, αναφέρθηκε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ενδείξεις ότι θα σταματήσει η διαδικασία διεύρυνσης, ιδίω σε αυτή την περιφέρεια που το έχει τη διεύρυνση τόσο πολύ, διεύρυνση τόσο πολύ ανάγκη. Εν γέννη όμως χαιρετίζουμε την έκθεση και σας διαβεβαιώνω ότι στην ε, ομάδα μου θα προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε στην προφορική διαδικασία για την ε, βελτίωση τη κατάσταση σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Επόμενο συνάδελφος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγγνώμη, ε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για το περιεχόμενο τη έκθεση, αλλά γενικότερα και για την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το 25 τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε και ότι θα έχουμε τη στήριξή σας και μέσα στα επόμενα χρόνια. Επί τη ευκαιρία να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση για ένα πολύ σημαντικό θέμα που βρισκόμαστε ότι αφορά τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και σύνδεση που θα αποτελέσει ιστορικό βήμα στις σχέσεις μας με τη Σερβία. Συγγνώμη, διαφωνώ. Μιλήσω με το κοσμοπέδιο. Η αρχική, μάλλον ε, μονογραφήθηκε η συμφωνία στις 25 Ιουλίου. Ε, η συμφωνία αυτή είναι εμπεριστατωμένη, ολοκληρωμένη και εύρωστη, καλύπτει όλες τις κύριες ε, θεματικές ενότητες που καλύπτονται και από τις υπόλοιπες τέτοιες συμφωνίες στην περιφέρεια. Μετά τον Ιούλιο έχουμε περάσει σε φάση νομικής επαλήθευσης και μετάφρασης ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα αλβανικά και στα σερβικά. Θα ολοκληρωθεί στα τέλη Μαρτίου αυτή η διαδικασία και ελπίζουμε να έχουμε την έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή τον Απρίλιο και να υποβληθεί στο Συμβούλιο τα τέλη Απριλίου. Επισημαίνω ότι το Κοινοβούλιο έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτή τη διαδικασία βάσει του άρθρου 218 της Συνθήκης προβλέπεται σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και όταν θα υπάρξει σύμφωνη γνώμη του έχει εγκριθεί μάλλον η συμφωνία από το Συμβούλιο και υπογραφή μεταφέρεται, διαβιβάζεται στο Κοινοβούλιο για την σύμφωνη γνώμη. Αν ε, θέλουμε να ληφθεί, να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία ε, το 2016, θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού, γιατί θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Και να κινηθείτε κι εσείς γρήγορα από πλευρά σας. Ε, να υπογραμμίσω εδώ ότι η συμφωνία αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ε, απαιτεί κύρωση από τα κράτη-μέλη, ούτε ενδιάμεση συμφωνία. Ουσιαστικά από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και μετά, από τη σύναψη της συμφωνίας και μετά, τίθεται σε ισχύ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αποφασιστικό βήμα στην πορεία του κοσμοπεδίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μόρτζιου. Κατανοούμε και έχουμε πλήρη επίγνωση της ε, σημασίας των συμβατικών σχέσεων και του γεγονότος ότι θα υιοθετηθεί και θα εφαρμοστεί από την στιγμή της ε, σύναψης της συμφωνίας. Κυρία Λούνατσεκ, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να διορθώσω κάτι που είπα στην πρώτη μου παρέμβαση. Ξέρω ότι υπάρχουν δύο γυναίκες υπουργοί του Κοσμοπεδίου, παρόλα αυτά δεν τις ανέφερα και γι' αυτό θα ήθελα να το διορθώσω αυτό. Το Κοσμοπέδιο έχει δύο γυναίκες υπουργούς για την ε, Υπουργό ε, Εμπορίου και Βιομηχανία και Υπουργό Αρμόδια και ζητήματα σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο όμω από του 21 είναι ιδιαίτερα μικρό ο αριθμό, αλλά επισήμω να διορθώσω αυτό που είπα προηγουμένω, ότι δεν υπάρχουν δηλαδή γυναίκε υπουργοί στην κυβέρνηση του Κοσμοπεδίου. Υπάρχουν δύο. Τώρα, για τι παρατηρήσει των συναδέλφων μου, σα ευχαριστώ όλου και τους εσκιώδεις εισηγητές ε, που στηρίζουν την έκθεση αλλά στηρίζουν και την πορεία του κοσμοπεδίου προς την ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ελπίζω να έχω και τη στήριξη σας στην ψηφοφορία αύριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν ε, για αυτή σας τη στάση. Προς ε, τον κύριο Μακάλιστερ να πω σαφέστατα αναφέρατε αυτό που ήθελα να φέρω και εγώ με αυτή την προφορική τροπολογία. Μιλάμε και για τα δίκτυα διακίνησης ε, ανθρώπων που δημιουργούν έτσι φήμες ότι ναι θα λάβετε το καθεστώς ε, ασύλου στην Αυστρία, στη Γερμανία και αλλού και αυτό δεν ισχύει. Είναι σαφές λοιπόν. Είναι σαφή η θέση μας από την ε, έκθεση. Για τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σας ευχαριστούμε για τις εργασίες σας επί της συμφωνίας ελπίζουμε να τεθεί σε ισχύ το στομότερο δυνατόν. Τώρα να πέρασω στα γαλλικά για να απαντήσω στον κύριο Σουφάτ, γιατί γνωρίζετε ότι δεν συμφωνούμε και δεν συμμερίζομαι την άποψή σας, όμως ήθελα να πω τρία πράγματα για τα όσα είπατε. Πρώτον, είπατε ότι είστε αντίθετος στην λογική της ε, ολοκλήρωσης ε, Λυπάμαι που εσεί, η πολιτική σα ομάδα, το κόμμα σα μάλλον και άλλοι στο Κοινοβούλιο δεν συμμερίζονται την ε, άποψη ότι η ολοκλήρωση και η προσχώρηση όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων είναι ένα ε, έργο ειρήνης, γιατί υπήρχαν πόλεμοι σε αυτή την περιφέρεια, υπήρχε πόλεμος που δεν θέλουμε να ξαναδούμε. Ούτε εγώ, ούτε και η μεγάλη πλειονότητα ε, του Κοινοβουλίου. Για μας λοιπόν είναι μια διαδικασία ειρηνευτική. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνει. Δεύτερον, μιλήσατε για εθνοκάθαρση κάποιων ε, Αλβανών έναντι Σέρβων. Ναι, υπήρξαν και εγκλήματα από των Αλβανών έναντι των ε, Σέρβων. Αλλά επειδή οι Αλβανοί αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα, βασικά αποφάσισαν να πολεμήσουν πριν ε, ε, πρώτα χωρίς όπλα και μετά πολέμησαν με όπλα ε, εξαιτία του καθεστώτος Μιλόσεβιτς που προχώρησε σε εθνοκαθάρσεις για πολλά χρόνια. Γι' αυτό και η διεθνής, το Διεθνές Δικαστήριο τον Ιούλιο 2010 απεφάνθη σαφώς ότι η δήλωση ανεξαρτησίας του Κοσμοπεδίου δεν αντίκειτο στο διεθνές ε, δίκαιο. Και τρίτον, μίλησατε για το κοσμοπέδιο ως εστία εγκληματικότητας. Ναι, πράγματι υπάρχει εγκληματικότητα και οργανωμένο έγκλημα και στο κοσμοπέδιο. Όμως, σε όλες τις χώρες της περιφέρειας υπάρχει αυτό, αλλά και στις δικές μας χώρες. Υπάρχουν εγκληματικά δίκτυα και στις χώρες μας. Να μιλήσω μόνο για τη δική μου. Δεν θα μιλήσω καν για τη Γαλλία. Για τη δική μου, για την Αυστρία. Την Τετάρτη ξεκινά μια μεγάλη δίκη κατόπιν, ή μάλλον διερεύνηση και στο δικό μας κοινοβούλιο ε, για εγκληματικά δίκτυα που συνδέονταν με τράπεζες και ούτω καθεξής. Γι' αυτό αναφέρω και στην έκθεσή μου ότι υπάρχουν επικρίσεις. Δεν έκαναν αρκετά τα τελευταία χρόνια για να καταπολεμήσουν αυτή την εγκληματικότητα. Όμως αυτό δεν αφορά μόνο το κοσμοπέδιο. Υπάρχουν αυτές οι προσπάθειε που έχουν καταβληθεί και από πλευρά Κοσμοπεδίου και από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Thank you very much, Madam Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λούνατσεκ. ολοκληρώνεται έτσι τη συζήτηση για την ε, έκθεσή σα, έκθεση πρόοδου για το Κοσμοπέδιο 2014. Και ε, ε, προχωρούμε στο επόμενο σημείο, υπαριθμόν 8, έκθεση πρόοδου 2014 για τη Σερβία. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η Σερβία άρχισε διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο του 2014 και η διαδικασία screening ελέγχου ε, διεξήχθη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο δεν έχουν ανοίξει μέχρι τώρα κεφάλαια. Στις 9 Φεβρουαρίου ο διάλογος Βελγραδίου Πρίστινα σε υψηλό επίπεδο επαναλήφθη και οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν για τα δικαστικά θέματα. Επίσης έχει γίνει πρόοδος την τελευταία ε, χρονιά, αλλά παραμένουν πολλά να γίνουν, ιδιαίτερα για την ελευθερία της έκφρασης και του τύπου, ενίσχυση της δικαιοσύνης. Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις, αλλά θα πρέπει τώρα να υλοποιηθούν, όπως επίσης και οι συμφωνίες με τη Φρίστινα. Ε, το Μάιο του 2014 πλήγει από πλημμύρες η Σερβία, που επέδρασαν ε, ακόμα πιο αρνητικά στην οικονομία. Ο συνάδελφος Μακάλιστερ έχει κάνει την έκθεση, 222 τροπολογίες των συναδέλφων και μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές συναδέλφους του κατάφεραν ε, τις 222 να τις κάνουν 22 συμβιβαστικές που έχετε στα χέρια σας. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μακάλιστερ για να παρουσιάσει την έκθεσή του. Είναι η δεύτερη φορά που τη συζητούμε. Παρακαλώ, έχει το λόγο. David. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, λέει στα κροατικά ο, ο ε, εγώ επισκέφθηκα τη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο την περασμένη εβδομάδα και μεταξύ άλλων συναντήθηκα με τον πρόεδρο Μίκολιτ στο Βελιγράδι, τον πρωθυπουργό Βούτσης και τον υπουργό εξωτερικών Ντάτσης και εκπροσώπους ε, των κομμάτων της αντιπολίτευσης αλλά και από την κοινωνία των πολιτών. Πολλά από όσα άκουσα και παρατήρησα με έκαναν να βεβαιωθώ ότι είμαστε σε σωστό δρόμο με το ψήφισμά μας. Όπως μόλις είπε ο, ο Πλένκοβιτς, 222 ήταν οι τροπολογίες που είχαν κατατεθεί. Δηλαδή κέρδισε σε δύο το Κόσοβο κατά 10 τροπολογίες. Αλλά ε, καμία τύχη απέναντι στον Τάνοκ, ούτε και το Βάιγκελ με την έκθεση για τη Μακεδονία που ήταν περίπου 300 οι τροπολογίες. Βασικό το θέμα ήταν ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και πολλές ακόμα ε, τροπολογίες είχαν να κάνουν με εξωτερική πολιτική, εξομάλυνση των σχέσεων με τον Κόσοβο, ελευθερία του τύπου στη Σερβία και διεθνείς σχέσεις στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές στο Στρασβούργο πριν από δύο εβδομάδες, πολύ επικοδομητική και γόνιμη συμφωνήσαμε να παραμείνει το ψήφισμα όσο γίνεται πιο ευσύνοπτο και ακριβές. Επειδή είναι μεγάλη η ποικιλία των διαφόρων τροπολογιών, αποφασίσαμε να μην βάλουμε διμερεί θέματα ή συμφωνίες και να μην αναφερθούμε σε ειδικές περιπτώσεις. Τελικά συμφωνήσαμε σε 21 συμβιβαστικές, τις οποίες λάβατε πριν από λίγες ώρες. Ήταν σημαντικό για μας να τονίσουμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει πρώτα είναι τα βασικά, τα ουσιώδη θέματα, ιδιαίτερα κράτος δικαίου, οικονομική διακυβέρνηση, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και εξομάλυση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας. Αυτό αντανακλάται λοιπόν και στις ίδιες τις συμβαστικές τροπολογίες. Τονίζουμε ότι είναι ζωτική σημασία στη σχέση καλής γειτονίας και πόσο σημαντική είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με το Κόσοβο. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική της Σερβίας, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Υποστηρίζουμε τις ανεξάρτητες αρχές όπως είναι ο συνήγορος του πολίτη. Τονίζουμε και πάλι ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του τύπου είναι θεμελιώδη χαρακτηριστικά μιας δημοκρατίας. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων θα πρέπει να προαχθούν, να ε, προστατεύονται και να υλοποιούνται σε όλα τα επίπεδα της σερβικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα λάβαμε υπόψη μας ότι η Σερβία έχει εγκρίνει σημαντικούς νόμους για την πτώχευση, για τις ιδιωτικοποιήσεις, ε, για την ε, δικαιοσύνη και για τους ε, καταγγέλλοντες, whistleblowers, τα στρεβλά. Ε, όλα αυτά είναι θετικά και θα ήθελα να εθαρρύνω και την κυβέρνηση και τη Βουλή της χώρας αλλά κυρίως την κοινωνία των πολιτών να παραμείνουν στην ευρωπαϊκή τους πορεία και στον ευρωπαϊκό δρόμο. Όπως είπα στην πρώτη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μας, πιστεύω ότι το 2015 θα πρέπει να είναι το έτος ε, που θα ανοίξουν τα πρώτα κεφάλαια, ιδιαίτερα αφού για λόγους τεχνικούς το screening ε, θα ολοκληρωθεί τον άλλο μήνα κανονικά. Θέλω να ευχαριστήσω τους και τους ηγητές για την γόνιμη συνεργασία και πάλι πιστεύω ότι ε, καταλήξαμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τη γραμματεία ε, της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Με χαρά θα λάβω υπόψη μου όλα τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. David, που ήσουν τόσο σύντομο. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Edward Κούκαν, ο οποίο ε, είναι επικεφαλή τη αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου με τη Σερβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, σύντομα. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον εισηγητή που προετοίμασε ένα καλό κείμενο. Είναι ισορροπημένο και πλήρε και νομίζω ότι αντικατοπτρίζει αντικειμενικά την πρόοδο της Σερβίας νομίζω ότι θα πρέπει να σκοπεύσουμε στο να έχουμε μια ρελιστική έκθεση για τη Σερβία, υπογραμμίζοντας τα κύρια επιτεύγματα και πιέζοντας για το να ξεκινήσουν τα πρώτα διαπραγματευτικά κεφάλαια. Ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή που συμπεριέλαβε την τροπολογία για το να ανοίξουν τα διαπραγματικά κεφάλαια στις συμβαστικές τροπολογίες. Επίσης πιστεύω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε την σημασία των τροπολογιών που αφορούν την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και του κράτους δικαίου. Θα πρέπει πολύ προσεκτικά να εξετάσουμε το πώς αναπτύσσονται αυτοί οι τομείς. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στις τροπολογίες που αφορούν την εξαρτησία του γραφείου του συνήγορου του πολίτη, γιατί έχουν ε, υπάρξει κάποιες αμφισβητήσεις τελευταία. Στις άλλες εκθέσεις που συζητήθηκαν σήμερα είδα πολλές τροπολογίες που να αφορούν διμερεί ζητήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο σόφρονες με αυτές τις τροπολογίες γιατί αντιμετωπίζουν κυρίως θέματα μειονοτήτων που είναι πάντοτε πάρα πολύ ευαίσθητα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο γενική διατύπωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Έντουαρτ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Φαγιόν που είναι σκιώδη, εισηγήτρια. Ευχαριστώ, θα μιλήσω σλοβενικά, λέει κυρία Φαγιόν. Καταρχήν, συγχαρητήρια στον εισηγητή για την καλή του δουλειά. Νομίζω ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες και αυτό αποδεικνύει περαιτέρω ότι η πολιτική της διεύρυνσης είναι πολύ σημαντική για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες που κατατέθησαν από τους συναδέλφους μου κυρίως αφορούσαν το θέμα των μεταρρυθμίσεων και της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων αφορούσαν ε, την ε, διαδικασία της εξομάλυνσης ε, των σχέσεων με το Κωσυφοπέδιο. Πολλοί εξέφρασαν ανησυχίες για την ελευθερία των μέσων μαζικής και επικεντρωθήκαμε στην προστασία των μειονοτήτων και των ευπαθών ομάδων. Επίσης, ε, ζητάμε να καταπολεμηθεί το οργανωμένο εγκλήμα και διαφθορά. Υπάρχει και μια προφορική τροπολογία προς την κατεύθυνση αυτή, σχετικά με την ελλειψή διαφάνειας ε, για, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στο γραφείο του Συνήγορου του Πολίτη. Εμείς κάνουμε την εξή έκκληση. διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις ε, για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι διαφανής και καλούμε την κυβέρνηση στο Βελγράδι να συμπεριλάβει και την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες, το κοινό σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει οι πολίτες να είναι ενημερωμένοι, να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Επιπλέον η Σερβία θα πρέπει να συνεργαστεί με τα όμορα κράτη της ε, προκειμένου να ε, αναπτύξει τις ε, συνορικές περιοχές. Αυτό είναι σημαντικό για τη συνοριακή συνεργασία. Επίσης υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία ε, που έχει να κάνει με τα θύματα πολέμου. Έχει κάνει μεγάλη πρόοδο η Σερβία, είναι σοβαρός εταίρος, έχει προευρωπαϊκή στάση και θέλω να αναφερθώ και στο ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος για την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Βελιγραδίου. Οι εκπρόσωποι της νέας κυβέρνησης ήταν εκεί αυτή τη φορά και το ίδιο και η κυρία Μογκερίνη. Υπήρξε συμφωνία για το δικαστικό σύστημα και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει την περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεων. Όπως ξέρετε, απευθύνουμε έκκληση να ξεκινήσουν το συντομότερο διαπραγματεύσει και σε πολύ σημαντικά κεφάλαια όπω το 23 και το 24. Και μπορώ να αναφέρω ότι η κυβέρνηση της Σερβίας επισκέφθηκε τη Σλοβενία την περασμένη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργό Μπούτσιτς ήταν εκεί. Και όπως είπαν και οι δύο εταίροι, η Σλοβενία είναι πάρα πολύ σημαντικό εταίρο για τη Σερβία και ένα συνδεσμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ο πιο στενό σύμμαχο τη Σερβία στη Σλοβενία. Τι ήθελα να ευχηθώ ότι καλύτερο στη Σερβία, στο δρόμο προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι η σημερινή έκθεση θα πρέπει να σα δώσει τα κίνητρα για να πράξουμε όλες ένα απαραίτητο για κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ Τάνια. Τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ ο είναι εισηγητής ε, από το ECR. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ το μόνιμο εισηγητή David McAllister για την ιδιαίτερα επιμελή και πλήρη έκθεσή του σε ένα φάκελο γεμάτο προκλήσεις ε, με πολλές διαφορετικές πτυχές. Φυσικά είναι ο κύριος περιφερειακός παίκτη της Σερβίας ε, και πρέπει να πω ότι κάποιος που είναι φίλος της Σερβίας για πολλά χρόνια ε, η πρόσφατη θέση που έχει πάρει για ορισμένα θέματα εξωτερική ε, πολιτική, όπω ε, παραδείγματο χάρη να διαφωνήσει με την επιβολική Ρώσων από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη Ρωσία, είναι ένα θέμα που μα ανησυχεί, όπω και άλλα θέματα, όπω τα δικαιώματα των μειονοτήτων και η ανάγκη για διαφάνεια και για δίκες διαδικασίες για το τι έγινε κατά την περίοδο του πολέμου δικές αποζημιώσεις για το τι έγινε στην περίοδο του πολέμου. Επίση, άλλε χώρε, τα Δυτικά Βαλκάνια, όπω και το Μευροβούνιο, για το οποίο είμαι ε, συγητή, έχουν ε, παρομοιά θέματα. Σίγουρα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και το να υπάρχει, να δημιουργήσουμε και ένα καλό κλίμα για τι επιχειρήσει και να συνεχιστεί και ο διάλογο με την Πρίστινα. Θα δράξω την ευκαιρία και πάλι για να θέσω ένα θέμα που μου έθεσαν πολλές επιχειρήσεις στη Σερβία. Το αμφιλεγόμενο ζήτημα του άρθρου 234 του ποινικού κώδικα και την πιθανή κατάχρησή του για πολιτικούς σκοπούς. Σε ό,τι αφορά ε, την ε, ε, χρήση ιδιωτικής ιδιοκτησίας ε, από το δημόσιο με καταχρηστικό τρόπο. Εξακολουθεί να παραμένει πρόβλημα αυτό και στο να υπάρχει ένα ελεύθερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Σερβία. Όμως ε, παρόλα αυτά εμείς θα υποστηρίξουμε τις 21 συμβαστικές τροπολογίες και το συνολικό πνεύμα της έκθεσης και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μακάλιστερ για την εξαιρετική δουλειά του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευεβάγγελα από τους Φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μου ικανοποίηση για την δουλειά που έχει γίνει με τον κύριο Μακάλιστερ. Ήταν μεγάλη χαρά να συνεργαστώ με τον κύριο Μακάλιστερ, τον εισηγητή και να μπορέσουμε να καταρτήσουμε μια σύντομη και αποτελεσματική έκθεση. Διαπραγματευθήκαμε και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες πολύ ολοκληρωμένες και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό ε, είναι ένας τρόπος που εκφράζει τη μαεστρία της γερμανικής διπλωματίας. Η Σερβία σίγουρα έχει ευρωπαϊκή πορεία, αταλάντευτη. Και η τρέχουσα, η σημερινή κυβέρνηση έχει διαλέξει να δώσει σημασία στην οικοδόμηση ε, της, ε, ενός χώρου που θα την προσεγγίσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα αναγνωρίζουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε υψηλότερο, υψηλότερο πολιτικό επίπεδο αξίζει να αναφερθούμε στην προσπάθεια που γίνεται για τη συμφιλίωση με τις γειτονικές χώρες ή περιοχές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι υπ' αυτή την έννοια είναι σημαντικό και το είπαμε αυτό, είναι σημαντικό να τονίσουμε την προστιθέμενη αξία της στροφής προς την Ευρώπη της Βοηβοντίνας. Και είπαμε ότι αυτός ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός πρέπει να στηριχθεί και ότι η αυτονομία της Βοηβοντίνας θα πρέπει να διευρυνθεί. και να έρθουν τα εμπόδια. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη Σερβία, στη Προεδρία ε, του ΟΑΣΕ. Θα είναι πολύ σημαντικό για τη σερβική διπλωματία να διαδραματίσει επικοδομητικό ρόλο και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ως πολιτική ομάδα θα υποστηρίξουμε όλες τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Συγχαίρω τον εισηγητή για την σύνταξη αυτών των συμβιβαστικών τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούνατσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι εισηγήτρια για το κοσφοπέδιο. Ωστόσο, ο σκιώδης εισηγητής της, για τους πράσινους μου ζήτησε να το αντικαταστήσω και γι' αυτό τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος της πολιτικής ομάδας μου και όχι ως εισηγήτρια για την έκθεση για το κοσυφοπαίδιο. Παρόλα αυτά θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ντέιβιτ Μακάλιστερ για την πολύ καλή συνεργασία. Ε, αυτά μου ζητήθηκε να σας μεταφέρω κύριε Μακάλιστερ. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, οι συμβιβαστικές τροπολογίες είναι πολύ καλές και ε, θα τύχουν στήριξη ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι συμβαστικές τροπολογίες που ε, επιβραβεύουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Σερβίας. Σας ευχαριστώ γιατί περιλάβατε πολλές από τις δικές μας τροπολογίες των πρασίνων. Θα ήθελα να σταθώ σε κάποια σημεία που περιλαμβάνονται στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες και τα οποία βρίσκω εξαιρετικά σημαντικά. Η Τάνια Φαγιόν το ε, ανέφερε προηγουμένως η σημασία της ανεξαρτησίας των μέσων επικοινωνίας στη Σερβία του τύπου. Είδαμε ότι είχαμε επιθέσεις στο δίκτυο ανεξάρτητης δημοκρατίας των Βαλκανίων μεταξύ άλλων ε, ερευνητικής δημοσιογραφίας και πρέπει να υπάρξει πρόοδος ως προς αυτό και γίνεται αναφορά. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Μακάλιστερ διότι έχετε συμπεριλάβει μια τροπολογία ε, την οποία έχω συντάξει εγώ. 11. Ε, υπαριθμών 11. Καλούμε τις σερβικές αρχές να ανοίξουν τα αρχεία του Ιουκοσλαβικού στρατού για να υπάρξει αλήθεια για τα περασμένα γεγονότα και να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Και έρχομαι τώρα στη συμβιβαστική τροπολογία 12. Θα ήθελα να πω ότι βεβαίως η Σερβία προοδεύει στα ζητήματα των δικαιωμάτων ε, λεσβιών, ομοφιλοφίλων, φιλομεταβατικών κτλ. Και έγινε πορεία ειρηνική, χωρίς προβλήματα και αυτό αξίζει σχολιασμού στην έκθεση. Και τέλος, να εκφράσω την εκτίμησή μου για το γεγονός ότι ο εισηγητής συμπεριέλαβε επίσης το ότι ζητείται από τις σερβικές αρχές και την κυβέρνηση να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ε, προσέγγισης της νομοθεσίας τους με τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο είναι προαπαιτούμενο για να πετύχουμε τους στόχους του 2020. Ε, βεβαίως η ομάδα των Πρασίνων στηρίζει πλήρως τη σχετική συμβιβαστική ε, τροπολογία. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη επιτυχία στην ψηφοφορία αύριο. Ευχαριστώ κύριο Καστάλτο παρακαλώ. Ευχαριστώ εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μακάλιστερ που έκανε εξαιρετική δουλειά. Και μπορώ να πω ότι ήταν και ιδιαίτερα συμπεριληπτική. Έλαβε υπόψη τι παρατηρήσει που παρουσιάστηκαν από διάφορε ομάδε και διαφορέ από τι δικέ μου τροπολογίε. Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη η έκθεση και αντικατοπτρίζει και τι πρόοδους αλλά και τα κενά που πρέπει να καλυφθούν ε, ακόμη στο μακρύ δρόμο που περιμένει τη Σερβία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια είναι πολύ σημαντικό να επεγραμμίσουμε τη διαδικασία εξομάλυνσης σχέσεων με το κοσυφοπαίδιο το διάλογο με την Πρίστινα που θα πρέπει να αντικοποιηθεί για να υπερβληθούν τα εμπόδια που ακόμη χωρίζουν τις δύο χώρες. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και μια εξαιρετική σχέση συνεργασίας μεταξύ των εισηγητών Λούνα και Μακάλιστερ για τους δύο φακέλους, όπως και η καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος και της διαφθοράς. Θέλω να υπογραμμίσω στους συμβιβασμούς 8 και 9 εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά μου για το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται μια καταδίκαση της Σερβίας που δεν έχει ευθεγρυμιστεί με τη θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για το θέμα της Ρωσίας. Η κριτική μου δεν έχει να κάνει με το την λανθασμένη μία ευθυγράμμιση, γιατί κατανοούμε το πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια συνεκτική πολιτική μεταξύ της Ένωσης ε, και των υποψηφίων χωρών. Όμως εγώ θα ήθελα να εκφράσω κάποιες επιφυλάξεις για την επιλογή της πολιτικής επιβολής κυρώσεων. Όμως, εδώ θα πρέπει να δούμε τη Σερβία ως ένα σημείο επαφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία γιατί υπάρχουν ε, συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών και επίσης είναι καλό και που ο ΑΣΕ, με συγχωρείτε, προσπαθεί να διαμεσολαβήσει για την επίλυση της κρίσης. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Μαριάννα Πετήρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Άλιστερ εργάστηκε με μεγάλο ενθουσιασμό για την έκθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά λείπει κάτι σημαντικό από την έκθεση και εμεί θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό εμπόδιο. στον δρόμο της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά είναι τα άστρα 2 και 3. Σε ό,τι αφορά την δικαιοδοσία που έχουν οι κυβερνητικέ αρχέ στο να δικάσουν εγκληματίε πολέμου. Εγώ νομίζω ότι το να καταργηθούν αυτά τα δύο άρθρα θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι ενταξικές διαπραγματεύσεις στα, στα κεφάλαια 23 και 24. Γιατί με αυτό το νόμο για πέντε χρόνια έχουν εκδιώξει και δικάσει τον κύριο Μάριτς και το αποτέλεσμα είναι ότι έχει υπάρξει παραβίαση πολλών συμφωνιών μεταξύ Σερβίας και Κροατίας. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η Σερβία δικαιούται να μηνύσει τους δικούς σου πολίτες. Αυτό αποτελεί προηγούμενο που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και εγώ νομίζω ότι κανένας ε, δεν θα επέτρεπε στους πολίτες του να υποστεί μια τέτοια μεταχείριση. Είναι λοιπόν απαράδεκτο να το κάνει αυτό η Κροατία. Δεν μπορούμε να δεκτούμε ανάμειξη της Σερβίας στα εσωτερικά της Κροατίας. Επομένως, εγώ έχω μαζί με την ομάδα μου καταθέσει μια τροπολογία που απαιτεί την κατάργηση των άρθρων αυτού του νόμου που δίνει τη δυνατότητα στην βία να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία. Εμείς θα πρέπει ως βουλευτές να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου και γι' αυτό σας καλώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μας που ζητούν τη διαγραφή των άρθρων 2 και 3 αυτής της συγκεκριμένης νομοθεσίας της Σερβίας. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πίτσουλα. Ευχαριστώ. Καταρχήν ε, θα ήθελα να επενέσω την πολύ σοβαρή δουλειά του κυρίου Μακάλιστερ. Έπρεπε να καταγράψει την πρόοδο ή την μη πρόοδο της Σερβίας ε, στην έκθεση κατάφερε να το αποτυπώσει. Όπως είπα και πριν λίγες εβδομάδες, η πρόεδρος της Σερβίας την ευρωπαϊκή πορεία της είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται για μια χώρα η οποία έχει μια συγκεκριμένη ευθύνη για τη ε, ποιότητα των σχέσεων των κρατών στα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης, η Σερβία μπορεί να είναι ενεργή και μπορεί να βελτιώσει πολλά εσωτερικά σημεία της εσωτερικής της δομής για να συνεισφέρει στην περιφερειακή σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Τα Δυτικά Βαλκάνια είναι μια περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη πολιτική δυναμική και πρέπει να πούμε ότι είναι προφανές ότι ενέχονται και αρκετοί κίνδυνοι, πολιτικοί, οικονομικοί κίνδυνοι ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, αυτό το βλέπουμε στην πράξη όταν πρόκειται για μειονότητες. Η πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση θα συνείσφερε σε καλύτερη συνεννόηση της Σερβίας με τους γειτονές της. Θα ήθελα επίσης να πω ότι οποιαδήποτε χώρα που έχει ευρωπαϊκές φιλοδοξίες θα πρέπει να σέβεται όχι μόνο το κεκτημένο αλλά και την ε, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ε, αν ανοίξει το κεφάλαιο 21 θα στείλει το σωστό μήνυμα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει κάποιες προκλήσεις στα Βαλκάνια. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη συνολική πρόοδο που έχει κάνει η Σερβία. Ευχαριστώ, επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που συνεγάρισαν τον εισηγητή κύριο Μακάλιστερ. Η έκθεση είναι ιδιαίτερα ρεαλιστική και ισορροπημένη. Χαίρομαι που επέλεξε μία σύντομη και σαφή έκθεση και επέμενε στα αρχές τους ό,τι αφορά τα διμέρη ζητήματα. Είναι ρεαλιστική λοιπόν η έκθεση, μπορώ να την αποδεχθώ, δεν θέλω να επισέλθω τις λεπτομέρειες, θα ήθελα μόνο να προσθέσω κάποιες γενικές παρατηρήσεις έχουμε το εξή πρόβλημα. Κάποιες φορές λέμε ναι στα διμερεί ζητήματα, κάποιες φορές όχι. Πριν από μερικά λεπτά μόνο, συζητήσαμε ένα θέμα όπου εξετάσαμε τα διμερεί ζητήματα, ενώ σε αυτή την έκθεση δεν θα μιλήσουμε για διμερεί ζητήματα. Καλό λοιπόν είναι να έχουμε τα ίδια κριτήρια για όλες τις περιπτώσεις. Και συμφωνώ εδώ με τον κύριο Μακάλιστερ. Το δεύτερο σχόλιο μου αφορά το θέμα της ε, συμφιλίωσης. Η έκθεση υπογραμμίζει το θέμα της συμφιλίωσης μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Θα ήθελα το θέμα της συμφιλίωσης να λάβει μεγαλύτερε διαστάσει στην ευρύτερη περιφέρεια. Ναι, διαφέρουν τα ζητήματα, αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό, μπορούμε, μπορεί να έχουμε και ανεπιθύμητε ε, επιπτώσει. Θα ήθελα λοιπόν να σα πω ότι διάβασα την ε, πρόταση των κρατών συναδέλφων σε ό,τι αφορά την ε, τροπολογία 58. Διάβασα την τροπολογία με αυτό το πνεύμα. Κάποιοι Κροάτες συνάδελφοί μας ε, αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα ως διμερές. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό απολύτως. Νομίζω ότι είναι και αυτό ένα θέμα ε, για το οποίο απαιτείται συμφιλίωση. Ωστόσο, να συγχαρώ τη Σερβία για τα επιτεύγματά τους και για την παραμονή τους ε, στην ευρωπαϊκή πορεία. Ευχαριστώ, Σόιτσα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο Μακάλιστερ για την ε, εξαιρετική του προσπάθεια. Είναι σύντομο και περιεκτικό το κείμενο της έκθεσής του. Σκοπίμως ε, επέλεξε αυτή την προσέγγιση και πέτυχε το στόχο του. Όπως γνωρίζετε η κρατική αντιπροσωπεία έχει υποβάλει ε, τροπολογίες. Ευχαριστούμε όσους τις αποδέχτηκαν, όμως ε, ακόμα υπάρχει λόγος ε, συζήτησης για όσους δεν τις έχουν αποδεχθεί. Η συνάδελφος Πετήρ επεσήμανε τις τροπολογίες 102 και 98. Νομίζω ότι πρέπει να τις συζητήσουμε περαιτέρω, τους ώστε να γίνουν περαιτέρω κατανοητές. Δεν συμφωνούμε με τη θέση που έχει λάβει η Σερβία απέναντι στο ε, στα εγκλήματα πολέμου στην ε, περιοχή αυτή κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90. Πρέπει να τα συζητήσουμε περαιτέρω αυτά τα θέματα. Ε, πρόκειται για τα άρθρα 2 και 3 και θεωρούμε ότι ο διάλογος είναι μια καλή βάση για όλα τα ζητήματα και επομένως θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος και για αυτό το ζήτημα. Παρεμπιπτόντως θα ήθελα να αναφέρω ότι κατά την ορκομοσία του νέου Προέδρου ήταν και ο Πρωθυπουργός Βούτιτς ε, παρόν, ένα πολύ καλό βήμα. Ε, προανήγγειλε επίσκεψη πρόεδρος ε, τον Μάιο στη Σερβία, η πρόεδρος Κροατίας και δεν θέλουμε να διαμορφωθεί η εντύπωση ότι η κρατική αντιπροσωπεία είναι και η Κροατία πιο συγκεκριμένα είναι υποδεέστερο κράτο. Δεν υπάρχει διακρισή και διαχωρισμό των κρατών μελών ανάλογα με το αν είναι στη Σέγγεν ή όχι και ούτω καθεξής. Αυτό ισχύει και εδώ στην περίπτωση κρατία. Επομένω, θέλουμε να έχουμε το βλέμμα στραμμένο προ το μέλλον και σε σχέση με τη Σερβία, ε, ώστε το σύνολο τη ε, νοτιοευρωπαϊκή νότι Ανατολικής Ευρώπης να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το διμερές ε, ζήτημα, κάποια έχουν συμπεριληφθεί στις ε, τροπολογίες, επαναλαμβάνουμε ε, την ανάγκη επίλυσης όλων των υποθέσεων αγνοουμένων, να τοποιηθούν όλοι οι αγνοούμενοι το ίδιο ισχύει και με τα πολιτιστικά αγαθά. Άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα είναι τα σύνορα στον ποταμό Δούναβη. Και θέλουμε οι εκπρόσωποι, ε, ή μάλλον η κροατική μειονότητα, να εκπροσωπείται και στην Εθνοσυνέλευση της Σερβίας. Να επαναλάβω κάτι ακόμα. Δεν θέλω να πιστέψει κάποιος ότι οι Κροάτες Ευρωβουλευτές ασκούν πιέσεις για να παρεμποδίσουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Θέλουμε να βοηθήσουμε τη Σερβία στη διαδικασία αυτή, να τους ε, προσφέρουμε ένα χέρι βοηθείας και ε, είμαι πεπισμένη, κύριε Μακάλιστερ, ότι και εσύ τον ίδιο ρόλο θέλετε να δραματίσετε και αυτό θα βρούμε μια καλή λύση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπω έγινε και με τα προβλήματα μεταξύ Κροατία και Σλοβενία. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει Βελέντερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Ντέιβιτ Μακάλιστερ για την εξαιρετική του αυτή έκθεση φέτος για τη Σερβία. Ο συζητής επέδειξε πραγματικά αξιοθαύμαστη ε, προθυμία και ανοιχτό πνεύμα στη διαχείριση των τροπολογιών. Έχει μια θετική ε, στάση ε, και για τις δικές μας τροπολογίες και τον ευχαριστώ εξ ονόματος της Ουγγρικής Αντιπροσωπείας διότι ήταν μεγάλο ζήτημα για μας αυτό και πολύ σημαντικό. Αυτό που έχει σημασία για μένα είναι το εξή. Όπως είπε και ο ίδιο ο εισηγητή προηγουμένω, η έκθεση αυτή πρέπει να είναι ισόρροπη και ε, έτσι τη βρίσκω κι εγώ. Το έχει καταφέρει. Από τη μια δίνει έμφαση στην ευρωπαϊκή προσήλωση της Σερβίας και στην ευρωπαϊκή της πορεία και προοπτική. Και αυτό το δείχνουν και τα θετικά σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορούν να δώσουν ε, περισσότερη όθηση, ενέργεια και δύναμη στην κυβέρνηση της Σερβίας να προχωρήσει σε αυτό το δρόμο. Το άλλο πολύ σημαντικό για μένα προσωπικά και για τους Ούγγρους ήταν τα δικαιώματα των μειονοτήτων που θα πρέπει να έχουν τη θέση που τους αναλογεί σε αυτή την έκθεση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά σε θέσεις εθνικά συμβούλια και τη σωστή και δίκαιη εκπροσώπηση των μειονοτήτων στη δημόσια διοίκηση και σε άλλους φορείς του δημοσίου. Αυτά είναι βασικά στοιχεία, τα αναφέρει η έκθεση και ευχαριστώ τον εισηγητή γι' αυτό. Που έλαβε υπόψη του τις δικές μας τροπολογίες σχετικά. Και τέλος, η έκθεση αυτή ε, είναι μια πραγματική δοκιμή για να δούμε και απόδειξη μάλιστα ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, σύμμαχοι και τέρι και παραστάτες στο πλευρό της Σερβίας προς την πόρια της αυτή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντέλη. Θα ήθελα να δώσω ε, το λόγο στον εαυτό μου. Αλλά πριν το κάνω αυτό, ε, θέλω να ακούσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα παρακαλούσα τον εκπρόσωπό της να ε, απαντήσει στα όσα είπαν κάποιοι συνάδελφοι και ρώτησαν. Αν μπορείτε δηλαδή να μας διευκρινίσετε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ε, την ε, παγκόσμια καθολική ποινική ε, δικαιοδοσία που υπάρχει στην ένωμη τάξη διαφόρων κρατών μελών. Και η Σερβία έχει δώσει στον εαυτό της αυτή τη δυνατότητα να καλύπτει όλο το έδαφος της πρώην Ιουγκοσλαβίας ε, δεν ξέρω αν μπορεί και ελπίζω να μπορέσει να απαντήσει με σαφήνεια σε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που σας ρώτησαν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αρχίσω με μερικά σχόλια για την έκθεση χωρίς να επαναλάβω τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη συζήτηση. Ευχαριστήσαμε πάρα πολύ τον εισηγητή και τονίσαμε ότι συμφωνούμε με τη γενική του εκτίμηση και την ε, εκτίμηση της Επιτροπής σας για την έκθεση. Για να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα ε, στην όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Τον άλλο μήνα τελειώνει το screening. Τώρα το συζητάει το Συμβούλιο της εκθέσεις για το κεφάλαιο 5 δημόσιες συμβάσεις, 20 ε, βιομηχανία και επιχειρήσεις και 26 παιδεία και εκπαίδευση. Αυτό που χρειάζεται τώρα η Σερβία είναι να έχει αποτελέσματα σε βασικούς τομείς, το κράτος δικαίου και περαιτέρω εξομάλυνση των σχέσεών της με το Κόσοβο. Η επανάληψη του διαλόγου Σερβίας-Κοσυφοπεδίου στις 9 Φεβρουαρίου με διαμεσολάβηση και διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ κρίσιμο και θετικό στοιχείο και θα βοηθήσει η συμφωνία για την δικαιοσύνη και το δικαστικό σύστημα στο Κόσοβο. Τώρα θα πρέπει και οι δύο πλευρές να υλοποιήσουν τη συμφωνία αυτή και αυτή τη στιγμή γίνει και η πρώτη αξιολόγηση. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 35, το οποίο ασχολείται με τη διαδικασία ακριβώς εξομάλυνσης στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι καλωσορίζουμε πάρα πολύ την έκκληση της έκθεσης για να ανοίξουν νωρίς τα κεφάλαια. Και το άρθρο, το κεφάλαιο 32 είναι έτοιμο να ανοίξει και ειλικρινά είναι και προς το δικό μας το συμφέρον αυτό. Γιατί αν ανοίξει αυτό που έχει να κάνει με τον ε, χρηματοοικονομικό έλεγχο θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, και θα δείξει ότι η Σερβία μπορεί σωστά και με ασφάλεια να διαχειρίζεται κοινοτικά κονδύλια. Σε άλλους τομείς συνεχίζεται εντατική δουλειά στη Σερβία, κεφάλαια 23 ε, κράτος δικαίου και 24 προγράμματα δράσης. Πολύ σημαντικά και αυτά τα κεφάλαια, ενδεχομένως να ανοίξουν στα τέλη του 2015. Σε σχέση με αυτό που μόλις είπατε, Πρόεδρε, έχει σημασία να μην προσθέτουμε απαιτήσει ή προαπαιτούμενα που δεν προβλέπει το κοινοτικό κεκτημένο ή διαπραγματεύσεις για την ένταξη. Και έρχομαι στην ερώτησή σας συγκεκριμένα. Πρώτον, υποστηρίζουμε την ιδέα ότι τα διμερεί ζητήματα θα πρέπει να λύνονται διμερώς να μην έχουν ε, αρνητικές επιπτώσεις στην ε, προενταξιακή διαδικασία. Το σωστό πλαίσιο είναι το διμερές. Αυτό το έχουμε κάνει και σε προηγούμενες διευρύνσεις. Ε, Γνωρίζουμε πλήρως ότι υπάρχει διαφορετική ε, χρειά στο θέμα της εξομάλυνσης σχέσεων με το Κόσοβο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παράδοση και την μεταγωγή ε, κλιματιών πολέμου, ε, το ρώτησαν και άλλοι συνάδελφοί σας, η Σερβία έχει ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων στο κεφάλαιο 23 και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βεβαιωθεί ότι οι συστάσεις αυτές εφαρμόζονται σωστά. Θα ήθελα να σας απαντήσω ειλικρινέστατα και σαφέστατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής το να συνδέσουμε τώρα το άνοιγμα του κεφαλαίου 23 ε, με την υποχρέωση της ε, βίας να τροποποιήσει νόμο που κατά τα άλλα είναι παρόμοιος με εκείνους που ισχύουν σε πολλά κράτη-μέλη. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Στο Βέλγιο υπάρχει αυτό, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κατοχώρηση, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει κοινοτικό και εκτιμένο. Αν το κάνουμε αυτό θα δημιουργηθεί προηγούμενο που θεωρούμε ε, εμείς αρνητικό και επιβαρυντικό. Αν μου επιτρέπετε, η νέα διατύπωση στην συμβαστική τροπολογία 12 ε, δίνει μια διέξοδο γιατί τονίζει πόσο σημαντική είναι η περιφερειακή συμφιλίωση και οτιδήποτε μπορεί να συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή συνιστά θετικό βήμα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούμε σήμερα να ζητούμε τροποποίηση του νόμου και μάλιστα να είναι αυτό απόλυτο προαπαιτούμενο πριν ανοίξει το κεφάλαιο 23. Ένα τελευταίο ε, και ε, υπάρχει πλήρης υποστήριξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Επιτρόπου Χάν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ελευθερία των μέσων επικοινωνίας. Είναι διαπραγμάτευτο αυτό θεμελιώδες δικαίωμα και ε, το θέτουμε και ε, στις συμφωνίες που έχουμε με άλλες χώρες εταίρους μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στον εισηγητή, πρέπει να παραδεχτώ ότι ανέμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι καλύτερο δουλειά στο σπίτι. Τώρα τώρα να μας αφέρετε κάποια πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την ε, ιονή δικαιοδοσία που έχει επεκτείνει η Σερβία στις ε, χώρες της πρώην Ιουκοσλαβικής ε, της πρώην Ιουκοσλαβίας ε, είναι ε, σημαντικό θέμα και θα σας ζητούσα να μην μπερδεύετε τώρα ε, να μην μπερδεύετε πράγματα που είναι άσχετα μεταξύ τους. Αυτό δεν θα έπρεπε να το κάνετε και θα ήθελα να μελετήσετε λίγο καλύτερα ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτού του νόμου ποιες είναι οι αρχές της ασφάλειας δικαίου στο διεθνές δίκαιο και στο ποινικό δίκαιο και τι σημαίνει εμπλοκή ε, το εσωτερικό δίκαιο στην δικαιοδοσία των άλλων κρατών. Δεν είμαι ικανοποιημένο ε, με την απάντησή σα, γιατί φαίνεται ότι η Κομισιόν δεν έχει μελετήσει επαρκώ αυτό το φάκελο και δεν το καταλαβαίνει. Και δεν είναι θέμα διμερών σχέσεων, είναι θέμα διεθνού δικαίου, καλών σχέσεων γειτονία που σχετίζεται με τι αξίε του κοινοτικού κεκτημένου. Και εγώ σκοπεύω να συνεχίσουμε τις συζητήσεις για αυτό το πολύ λεπτό και συγκεκριμένο θέμα που δυστυχώ ε, αφορά μόνο τη Σλοβενία και την Κροατία και όχι άλλε χώρε, αλλά αν θίγονταν ε, ίσω θα ήταν πιο ενεργητικέ σήμερα. Τώρα, θα ήθελα τώρα να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Άλιστερ και το συγχαίρω για αυτή την έκθεση που είναι δείγμα πολύ ποιοτική δουλειά και είμαι πολύ ικανοποιημένο με του συμβιβασμού που κατόρθωσε να παρουσιάσει, εμφανίζει μια σειρά ιδεών που είχαν διάφοροι συνάδελφοι. Έχετε το λόγο, David. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας και τη συνεισφορά σας. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Καθώς τέθηκαν συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις, δεν είμαι πολύ σύντομος. Εγώ προσπάθησα να καλύψω όσο δυνατόν περισσότερες τροπολογίες και προσπάθησα να διατηρήσω το ψήφισμα όσο το δυνατόν πιο συνοπτικό και συγκεκριμένο, γιατί ήθελα να είναι βενάγνωστο για τους ενδιαφερόμενους. Ίσως ε, στην έκθεση του χρόνου να έχουμε περισσότερη δυνατότητα για λεπτομέρειες και από το Μάρτιο η Κομισιόν θα ξεκινήσει το δικό της έργο για την έκθεση πρόοδου 2015 σε σχέση με τις τροπολογίες 98 και 102 που κατέθεσαν οι Κροάτες συνάδελφοι. Όλοι σημειώνουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές νομικές απόψεις για το θέμα αυτό και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη στο μέλλον. Θα ήθελα να κλείσω με την εξής ευχή. Το 2015 να είναι αποφασιστική χρονιά για το μακρύ δρόμο της Σερβίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι πιστεύω ότι θα είναι καλό μήνυμα να ανοίξουμε το πρώτο κεφάλαιο ή τα πρώτα κεφάλαια μιλώντας για τα κεφάλαια 23 και 24 αυτά είναι θεμελιώδη αλλά ξέρουμε όλοι ότι και το άρθρο 35 θα πρέπει να το δούμε στην αρχή της διαδικασίας και ε, μπορώ να πω ότι έγινε και ένα σημαντικό βήμα προς το στην κατεύθυνση στις 9 Φεβρουαρίου όταν έλαβε χορό ο πρώτος διάλογος ψηλοπιπέδου με την κυρία Μογκερίνη, την και την κυρία Μπούτσης εδώ στις Βρυξέλλες. Τώρα, αν, πώς, πότε θα πρέπει να ανοιχθούν τα κεφάλαια ή όχι, αυτό εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Νομίζω όμως ότι αυτή η έκθεση θα δώσει καλά επιχειρήματα στα κράτη-μέλη για να σημειώσουν πρόοδο και να βοηθήσουν τη Σερβία να ακολουθήσει την πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ. Και εδώ ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το σημείο 8 της σημερινής ημερησίας διάταξης και μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 9 το οποίο είναι οι συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Έρχεται ο κύριος Μπρόκ. Δεν είναι εδώ ο πρόεδρος. Θα συνεχίσω λοιπόν εγώ τη συζήτηση. Κάνουμε τώρα στην εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, της ΕΚΤΑ για τη διατλαντική τερική σχέση εμπορίου και επενδύσεων. Δεν ε, θα υπερβάλλω αν πω ότι η TTIP είναι η ε, η εξέλιξη που είχε τη μεγαλύτερη όθηση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, η δυνατότητα τη συμφωνία να θέσει ε, παγκόσμια πρώτα και κανόνε, ε, είναι σημαντική και για τι δύο μερέ. Ταυτόχρονα, οι διαπραγματεύσει ε, έχουν τύχη αυξημένου ελέγχου από το κοινή γνώμη και υπήρξαν φωνέ για την έλλειψη διαφάνεια, ε, ακόμη και για εμά ω μέλη του Διεθνού Κοινοβουλίου και γενικέ ανησυχίε για ότι ε, διακυβεύεται η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και, τις, ε, και τα πρότυπα ασφαλείας. Εδώ εμείς θέλουμε όμως να δώσουμε μια σκοπιά εξωτερικών σχέσεων στην έκθεση ίντα, στις διαπραγματεύσεις εμπορίου. Υπάρχει ο κίνδυνος στις λεπτομερείς συζητήσεις για κανόνες και διαδικασίες ε, να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Αυτή η συμφωνία θέλει να μειώσει το κόστος ε, για ένα μικρό ποσοστό κάπου και απλούστευση των προτύπων κάπου αλλού. Συνεισφέρει στο μέλλον της διατηλετικής σχέσης και της ενδυνάμωσης της συμμαχία μας με το πιο σημαντικό μας διεθνή εταίρο είναι η ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση που ε, θα πρέπει να επιστήσουμε στους συναδέλφους της ΙΝΤΑ. Και χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Μιλανμόν, ο οποίος εκπώνησε την γνωμοδότηση για την ΑΦΕΤ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και το κείμενο είναι σύντομο, έπρεπε να είναι σύντομο άλλωστε και νομίζω ότι είναι και αρκετά ξεκάθαρο. Συμφωνώ με αυτό που είπατε. Θέλησα να δώσω έμφαση, άλλωστε δεν μπορούσα να κάνω και αλλιώς, στις πτυχές που έχουν να κάνουν με την αρμοδιότητα τη δική μας, της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Αυτή η συμφωνία είναι πολύ ευρεία, περιλαμβάνει πολλές διαστάσεις και εγώ θέλησα να εστιάσω κυρίως στα θέματα που άπτονται της αρμοδιότητός μας. Υπογραμμίζουμε ότι η ΕΠΑ είναι ο πιο σημαντικός στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζουμε ότι αυτή η συμφωνία δεν έχει διαστάσεις που έχουν να κάνουν μόνο με το εμπόριο και τις ε, επενδύσεις. Θα ενισχύσει η συμφωνία αυτή την διατλαντική σχέση σε μια χρονική στιγμή λεπτή, ευαίσθητη, σημαντική. Διότι η ΕΠΑ αυτή τη στιγμή ε, προχωρούν στον επαναπροσανατολισμό τους προς την Ανατολή, προς την Ασία. Επομένως ε, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον κόσμο στις γεωγραφικές περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού και νομίζω ότι είναι σημαντικό σε Ευρώπη να συνάψουμε μια συμφωνία τόσο φιλόδοξη όσο είναι η διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και παιδίσεων. γιατί η ΕΠΑ είναι βασικός μας εταίρος. Από εκεί και πέρα. Δεν είναι μόνο διμερείς, ε, διμερεί τα σκέλη που μας ενδιαφέρουν. Είμαστε το 1 τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου. Το εμπόριο ε, από τη μία και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι το 1 τρίτο των παγκοσμίων εμπορικών συναλλαγών και αυτό είναι σημαντικό. Πέρα από αυτό όμως Ό,τι συμφωνήσουμε εμείς με την Αμερική θα έχει επιπτώσει σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ε, αυτή τη διάσταση γιατί ξεπερνά τα αμυγός διμερή όρια. Με αυτή τη συμφωνία ε, ατενίζουμε το ενδεχόμενο ενός οικονομικού χώρου ε, πιο ευρύ, πιο ευρέως χώρου αν θέλετε οι έχουν την ναύτα, είχαν την άφτα με τον Καναδά, το Μεξικό, με διάφορες άλλες χώρες και εμείς έχουμε με την Λατινική Αμερική, έχουμε πρόσφατα μια συμφωνία με τον ε, Καναδά, εδώ και 12 χρόνια προσπαθούμε να έχουμε συμφωνία με το Μεξικό και έχουμε συμφωνία με την Κολομβία, με το Περού και έχουμε και μια παλιά συμφωνία με τη Χιλή που θέλουμε να αναβαθμίσουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι με αυτή τη συμφωνία, την TTIP, μπορούμε να ε, ολοκληρώσουμε ένα τεράστιο οικονομικό χώρο και αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία παρόλο που η πρόοδος έγκυται στο Καναδά προς το παρόν. Από εκεί και πέρα, από πλευράς θεμάτων ενέργειας. Είναι σημαντικό. Η ενέργεια είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Το έχουμε συζητήσει επανελειμμένως στην Επιτροπή μας. Έχουμε συντάξει εκθέσεις για την ενέργεια και το σκέλος της που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική και γι' αυτό θέλω να τονίσω αυτό το θέμα σε αυτή την ε, έκθεση ή σε αυτή την γνωμοδότηση. Ίσως ε, θα πρέπει να μην υπάρξουν πλέον άδειε για, την εξαγωγή, ε, για τις εξαγωγές αερίου ή Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικέ πηγές. Ίσως θα πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί που υπάρχουν σήμερα για τις ε, εξαγωγές πετρελαίου, εάν τελικά προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα προβλέπεται συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κανονιστικών και ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ. Στενή συνεργασία σε τακτά χρονικά διαστήματα, πολύ σωστά πλαισιωμένη. Κάτι που πρέπει να κάνουμε ε, στο πλαίσιο του διατλαντικού νόμα παρασκευαστικού και νομοθετικού διαλόγου είναι να ε, ε, ενισχύσουμε αυτό το είδος διαλόγου του περί της νομοθεσίας. Δηλαδή οι επιτροπές που μπορούν και που έχουν αρμοδιότητα να προτείνουν νομοθεσία, η αντίστοιχη τον είπα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλό θα είναι να συσφίξουν τις σχέσεις τους. Είναι μια σχέση που ήδη υπάρχει, αλλά θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να ενισχυθεί έτσι περαιτέρω. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, Εάν τελικά ολοκληρώσουμε, φτιάξουμε αυτό το τεράστιο ολοκληρωμένο οικονομικό χώρο μεταξύ ΙΠΑ και ΕΕ, ίσως θα μπορούσαμε στη συνέχεια να εξετάσουμε μια διατλαντική ε, πολιτική ε, σχέση. Ε, το ενδεχόμενο μια τέτοιας ε, πολιτική συμφωνίας από τη στιγμή που ο οικονομικός χώρος γίνεται όλο και πιο ολοκληρωμένος, θα μπορούσαμε στη συνέχεια να έχουμε μια πολιτική συμφωνία πολύ πιο φιλόδοξη, κάτι το οποίο δεν υπάρχει βέβαια σήμερα. Και η η έκθεση αναφέρεται σε κάτι που είπε ο κ. Πλένκοβιτς προλίγου, το θέμα της διαφάνειας είναι κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως. Το τελευταίο 1,5 χρόνο πάρα πολλοί θεώρησαν ότι η διαφάνεια δεν είναι επαρκή, στο επίπεδο διαφάνειας δεν είναι επαρκές, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει βήματα προς τα εμπρός και έχουμε περισσότερη διαφάνεια για τα έγγραφα, για τη διαπραγματευτική εντολή, έχουμε περισσότερες γνώσεις για τους διαπραγματευτές και ούτω καθεξής και έτσι ε, εμείς ε, συγχαίρουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και κρίνουμε θετικά αυτή την αύξηση του επίπεδου διαφάνειας που έχει επιτευχθεί το τελευταίο 1,5 χρόνο. Τέλος, Κάτι που μου τράβηξε την προσοχή είναι το εξή. Η έκθεση του κυρίου Λάγκε στην ΙΤΑ θα ε, βασιστεί σε 14-15 γνωμοδοτήσεις. Σχεδόν όλες, όλες οι κοινοβουλευτικέ επιτροπές θα εκφράσουν γνωμοδότηση για την έκθεση της Ίτα. Και γι' αυτό εγώ θέλησα στη δικιά μας γνωμοδότηση, έκθεση αν θέλετε συμβουλευτική, να ασχοληθώ με ε, τις διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής. Άλλωστε πολλοί συνάδελφοι στις άλλες επιτροπές έχουν αγγίξει τα λοιπά ζητήματα. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι προσπάθησα να περιοριστώ. Δεν είχα και πολύ χώρο και να το ήθελα να επεκταθώ δεν θα μπορούσα. Αλλά επιθυμούσα κιόλας να ε, περιοριστώ ε, στα θέματα της αρμοδιότητάς μας γιατί η δική μας θα είναι μία από τις 14 που ε, θα υποβληθούν στον κύριο Λάγκε τον επικεφαλής από πλευράς Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΙΝΤΑ. Αυτό προσπάθησα λοιπόν να κάνω σε αυτό το προσχέδιο και με μεγάλη χαρά θα ακούσω τις υποδείξεις σας οι οποίες σίγουρα θα εμπλουτίσουν το κείμενό μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιλανμόν. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ζήλ Παγνιών από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ισχυώδης ηγετής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Σεγητά, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τον εισηγητή, κύριο Μιλάν Μον, ε, για το έργο του στο προσχέδιο ψηφίσματος μάλλον. Μια τέτοια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και ΕΠΑ είναι πολύ σημαντική σε τη φορά ε, τη γεωπολιτική πτυχή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να διαμορφώσουμε ε, το πολιτικό και τεχνικό σκέλος ε, του μεγαλύτερου εμπορικού χώρου στην Ευρώπη. Γι' αυτό και ασχολήθηκε η δική μας Επιτροπή. Όπως ανέφερε η συγητής, και εγώ πιστεύω πρέπει να στοχεύσουμε στην πτυχή που αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις της TTIP, για να μην αναλωθούμε σε διάφορα ζητήματα που δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Πρέπει να πάμε σε βάθος. Εάν επιθυμούμε, μπορούμε να το τροποποιήσουμε σε βάθος αυτή την ε, συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να επικεντρωθούμε στο δικό μας πεδίο εφαρμογής της Επιτροπής ΑΦΕΤ. Και αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου για αυτό το ψήφισμα. Πρώτον, απλήρης απουσία του ISDS, ε, του Μηχανισμού Επίλυσης Διαφορών είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι μία από τις κόκκινες γραμμές μου αυτός ο αποκλεισμός του ISDS. Ε, γιατί μια τέτοια κόκκινα γραμμή θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στο δικό μας ψήφισμα. Παράλληλα θα ήθελα να πω ότι δεν είμαι το αισιόδοξο συζητητή εισηγητής σε ό,τι αφορά τον θετικό αντίκτυπο του TTIP. Η Επιτροπή προβλέπει ε, αύξηση του ΑΕΠ, ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 0,5%. Ε, Εναλλακτικέ προβλέψεις, μάλιστα, ε, μιλούν ακόμα και για συρρήκνωση του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υποτιμήσουμε ούτε να υπερτιμήσουμε την συμβολή αυτής της συμφωνίας του TTIP στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μετά, για τα όσα αναφέρθηκαν για τη διαφάνεια, συμφωνώ. Όμως, το ίδιο Ρέιλι, τον ε, Γενάρη του 2015, η ίδια Μεσολαβήτρια λοιπόν ανέφερε ότι είναι απαραίτητα να βελτιώσουμε περαιτέρω την πρόσβαση του ε, Εβραίου κοινού στα κείμενα διαπραγμάτευση και να βελτιώσουμε τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τι ε, συναντήσει των υπαλλήλων τη Κομισιόν και των λόμπι. Πράγματι πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός εμπιστευτικότητας ε, στις διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ, ωστόσο η ε, αμερικανική ε, έλλειψη προθυμίας, προθυμία μάλλον, να μας να δημοσιεύσει τα κείμενα και τις λεπτομέρειες διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση σε αυτά τα κείμενα που θα πρέπει να, πρέπει να αιτιολογούνται και να τεκμηριώνονται επιμελώς για τις τροπολογίες που θα υποβάλω ε, εκ μέρους ε, της ε, ομάδας μου. Αυτά είχα να πω. Θα συνεργαστώ με τον εισηγητή για να βρούμε συμβασμούς αν αυτό είναι δυνατόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε. Συνάδελφε, τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Charles Tannock, σκιώδης εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Πλέκοβιτς. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον φίλο και συνάδελφο Μιλάν Μον για την εξαιρετική αυτή σύντομη και περιεκτική έκθεση μουσική σταθιά του ΙΣΙΑ, e των Ευρωπαίων Συνδετικών Μεταρρυθμιστών, οτιδήποτε ε, μιλάει για το TTIP με τέτοιο τόνο. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό πολιτικό και βορικό μέσο για την ομάδα μου. Ε, διαφωνώ με τους ε, Γάλλους τους που μίλησαν προηγουμένως. Από μεθοδολογική σκοπιά, εύρωστες μελέτες αναφέρουν ότι η αύξηση του ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου κατά συνέπεια του TTIP μπορεί να ε, ισούται και με τις Δικέ μας οικονομικέ εισφορέ ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, είμαι εξαιρετικά αισιόδοξο ότι θα βοηθήσει ε, πάρα πολύ την ευρωπαϊκή οικονομία σε μια περίοδο ε, στασιμότητας και στην Ευρωζώνη πιο συγκεκριμένα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πιστεύω ε, αυτή την όθηση και να στραφούμε περισσότερο σε αυτή την αναπτυσσόμενη ευρωατλαντική αγορά γιατί η ΕΠΑ έχουν στραφεί προς τα εκεί με όλες τους τις δυνάμεις ε, και θα είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για την επόμενη δεκαετία. Πρέπει και εμείς λοιπόν να επιμείνουμε. Αυτό ισχύει και για την ε, ε, πλευρά του ειρηνικού, με συνεργασίες των ΗΠΑ, με Μεξικό, Ιαπωνία και Ασία. Η δική μας συνεργασία με αυτές τις χώρες θα ήταν ένα πραγματικό όνειρο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τέτοιες εναλλακτικέ ε, έννοιες που έχουν ε, πολλοί ευρωσκεπικιστές ε, στη χώρα μου να λάβει ένα τέλος. Γιατί υπάρχει υπεποίθηση στη χώρα μου ότι αν αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο με, κάποιον τρόπο θα επανέλθουμε στην κοινοπολιτεία μαζί με τη ΣΥΠΑ. Νομίζω ότι το TTIP θα είναι κάτι το οποίο θα ενισχύσει ε, αυτή μου την πεποίθηση. Απορρίπτω και την ε, τρομοκρατία, την τρομολαγνία και όλα όσα αναφέρθηκαν για τον ISDS και πώς ε, παραβιάζει την κυριαρχία μας, υπονομεύει τις εθνικές μας υπηρεσίες και το καθεξής. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχουν ήδη συμφωνίες μηχανισμού επιλύσης διαφορών σε πολλές ευρωπαϊκές συμφωνίες εμπορίου και είναι απλώς ζήτημα κοινή λογικής και κράτους δικαίου. Ε, για την ε, διαμεσολάβηση και διευθέτηση, επίλυση διαφορών ε, όταν υπάρχουν διαφορές. Είμαι υπέρ λοιπόν του ISDS στο TTIP και συμφωνώ με τον Μιλάν Μον και πάλι ότι ίσως χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό κείμενο γεωπολιτικής επικέντρωσης, όπως είδαμε και στην περίπτωση του Καναδά πρόσφατα η ΙΠΑ είναι ο στενότερος μας εταίρος και η μεγαλύτερη και πιο σημαντική δημοκρατία στον κόσμο από πλευράς οικονομίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Τσάρλ. Η κυρία Σχάκη από την Άλτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μιγιάν Μον. Εξαιρετική γνωμοδότηση το σχέδιο αυτό επειδή καθημερινά ασχολούμαι με την TTIP, γιατί είμαι και μέλος στην Επιτροπή ΙΝΤΑ, ε, σας ευγνωμονώ που επικεντρωθήκατε σε ένα θέμα που συχνά λησμονείται ε, στη συζήτηση που είναι το γενικότερο παγκόσμιο και γεωπολιτικό πλαίσιο. Φαίνεται από τη γνωμοδότησή σας ότι αν θέλουμε να δούμε μια μετατόπιση ε, στην προμήθεια της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν μετριέται σε ευρώ έχει τεράστιο αντίκτυπο αν δεν είμαστε πια τόσο εξαρτημένοι από χώρες όπως είναι η Ρωσία ή η Σαουδική Αραβία. Ένα άλλο σημαντικό σημείο και θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτό είναι ότι και εμείς και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε ε, ήδη συμφωνίες ε, με τρίτες χώρες ε, που αν ευδοκιμήσει η συμφωνία TTIP όπως ελπίζω θα επηρεαστούν. Ας πούμε χώρες όπως η Τουρκία και το Μεξικό καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν για να μας πούν τις σκέψεις τους γιατί τους αφορά η συμφωνία επειδή έχουμε τελωνιακή ένωση. Επίσης, ε, πολυμερείς ε, σχέσεις ε, εμπορικές και συμφωνίες είναι θετικές και δεν θέλω να θεωρηθεί εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια αλλά είναι κάτι το θετικό και να συνδυαστεί με βάση το εμπόριο που θα βασίζεται πάντα σε κανόνες αυτό θα είναι υποφελές παγκοσμίω. Θα ήθελα να σταματήσω εδώ και να πω ότι δεσμεύομαι να συνεργαστώ με τον εισηγητή ε, έτσι ώστε η γνωμοδότησή του να επικεντρωθεί σε αυτό το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό στοιχείο. Υπάρχουν, όπω είπατε, και άλλε επιτροπέ που ασχολούνται με τα δικά του θέματα και γνωμοδοτούν και δεν χρειάζεται, πιστεύω, να συζητήσουμε το ISDS, το σύστημα επίλυση διαφορών, στα πλαίσια τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Και τώρα θέλω στο λόγο στον συνάδελφο Μέλανσο. Μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ε, ευχαριστώ, κύριε Σιγητά, για τον ενθουσιασμό της πρότασής σας, γιατί μου επιτρέπει να ε, ορίσω τις αντιφάσεις μας. Λυπάμαι που η Επιτροπή ε, ε, που θα ήταν η καλύτερη για να αποφανθεί δεν μίλησε, δεν είπε λέξη για τον τρόπο με τον οποίο κατασκοπεύουν οι ΗΠΑ τις πρεσβείες μας και τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφού ε, μιλήσαμε για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή, ένα εκατομμύριο 269.000 ε, πολίτες ε, υπέγραψαν σχέδιο Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας που ε, έκανε στην άκρη χωρίς να εξετάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και επίσης για εκείνους που εκφράστηκαν αρνητικά για το Δικαστήριο επίλυση Διαφορών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό το απόφησε θεωρώντας ότι δεν είχαν πλήρη ε, πληροφόρηση. Ε, όλα αυτά και ιδιαίτερα τα δικαστήρια επίλυσης διαφορών είναι ζήτημα δικό μας, της δικής μας Επιτροπής, γιατί εδώ πραγματικά ε, αλλάζουν τα γεωστρατηγικά δεδομένα γιατί βάζουν σε δεύτερη μοίρα τα κράτη και σε πρώτη μοίρα ιδιωτικά συμφέροντα, επενδυτές και εταιρείες. Ε, δηλαδή πρόκειται για πλήρη ανατροπή της Διεθνούς Ένωμης Τάξης, γιατί μέχρι τώρα τα διαιτητικά δικαστήρια ε, ε, έκαναν τη διαιτησία μεταξύ των διαφόρων εθνικών δικαστηρίων. Εδώ πρόκειται για διαφορές μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Το έγγραφο έχει μια διάσταση, θέλει να είναι γεωπολιτική και βιάζεται για να μην έρθουμε εκ των υστέρων οι Ηνωμένε Πολιτείε λέτε θα στραφούν προ τον ειρηνικό. Μα αυτό δεν είναι πάρα πολύ ε, νυφάλαιο σκέψη ή οξυδερκέ. Έτσι κι αλλιώ θα υπάρξει μια δια ειρηνική συμφωνία στον ειρηνικό ωκεανό. Εμεί έχουμε μια διατλαντική συμφωνία για να μπορέσουμε στη συνέχεια αυτό λέτε να το κάνουμε εθνικό, παγκόσμιο κανόνα. Δεν πρόκειται περί αυτού. Μέσω ε, αυτού θέλουν να επιβάλλουν αυτό που δεν κατάφεραν να περάσουν από τον ΠΟΕ ε, που έσπασε τα μούτρα του, για να το πω έτσι, ε, ε, μπροστά σε ένα παγκόσμιο κανονισμό διεθνούς εμπορίου, που σήμερα έχει γίνει ταύτα. Μετά, όταν αποκαλείται μέγα στρατηγικό εταίρο στις ΗΠΑ, Πολιτείες, εμπορικά δεν διαφωνώ, αλλά κανονικά αν τους αποκαλείται έτσι θα έπρεπε να ανησυχούμε γιατί ε, είναι ε, φθήνουσα υπερδύναμη και το νόμισμά τους κινδυνεύει τα μάλα αυτή τη στιγμή. Ε, είναι σε παρακμή. Κανονικά θα έπρεπε να ψάξουμε νέους εταίρους, νέους συμμάχους με την Κίνα γιατί όχι και με τη Ρωσία. Αλλά ξέρετε ότι αυτό το δρόμο δεν το παίρνουν. Και θα ανοίξουμε τώρα μια αγορά που φέρνει τις βιομηχανίες μας σε ευθεία μορφή ανταγωνισμού, αυτό για ποιο, πώς θεωρείτε ότι είναι ε, πρόοδος. Αυτός ο ανταγωνισμός θα είναι και κούρσα εις βάρος των ασθενεστέρων και δεν ε, είναι τα προϊόντα πάντα της δέουσας ε, περιβαλλοντικής ή άλλης ποιότητας. Και πολύ εφάνταστο το βρίσκω αυτό που λέτε, ότι αν πούμε σε μια μεγάλη διατλαντική αγορά θα πάρει μεγάλη φόρα και ορμή ευρωπαϊκή οικονομία ε, τελειώνω. Το, θερμόμετρο, ε, το χρονόμετρό μου δεν είναι εξίσου ακριβές με το δικό σας, Πρόεδρε. Ε, πάντως αναγνωρίζω και χαίρομαι για την ελληνική κυβέρνηση που είπε ότι θα βάλει βέτο στην ε, υπογραφή αυτής της συμφωνίας που θεωρώ κακή όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά γενικότερα για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε και τώρα ο κύριος Μέσεριτς, κατόπιν κύριος Καστάλτο, κύριος Πρέντο, κύριος Βαλτσίτης. Και στο τέλος ο κύριος Μιλανμόν. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να με μακρηγορήσετε. Γιατί διερμηνία θα έχουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Παρακαλώ κύριος Μέσεριτς, ευχαριστώ. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω και τον συγγετή για την γνωμοδότηση αυτή που πραγματικά είναι ιδιαίτερα εύστοχη και σύντομη. Είναι σημαντικό αυτή η Επιτροπή με επικεντρωθεί στα παγκόσμια αποτελέσματα και ιδίω ε, στις γεωπολιτικέ συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι οι πράσινοι δεν είναι και τόσο ενθουσιώδει για το όλο εγχείρημα. όπω πρέπει το σχάρι φίλοι μας ε, στο ECR, ότι φαίνεται να ακούγεται τόσο ευχάριστο για το ECR. Υπάρχουν ε, πολιτικέ στην οικονομία που ουσιαστικά δεν υποστηρίζουν τόσο τα καθολικά ωφέλη του ελεύθερου Διαφωνούμε γι' αυτό. Τώρα, αυτό που θα ήθελα να επαναλάβω σε σχέση και μας είπε ο της συνάδελφος είναι ότι αν και σημερινές διευθυντή της Κομιτιών σε σχέση με την ε, διαφάνεια των διαπραγματεύσεων πηγαίνουν κάποια βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά καλούν για, μεγαλύτερη διαφάνεια. Εγώ προέρχομαι από ένα κράτος μέλος, ε, το οποίο σήμερα δεν ε, μπορώ να πω είναι και το παράδειγμα της πολιτικής διαφάνειας σε κρατικό επίπεδο. Η πρόσβαση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις αυτές, ακόμη και στο δικό μου κράτος μέλος, ε, θα ήταν αμφίβολο. Αναφέρομαι λοιπόν στην ποιότητα αυτής της διαφάνειας αν ε, και αυτό ίσως να μην ε, είναι τόσο σημαντικό για αυτή την Επιτροπή, δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι όχι μόνο ο ελάχιστος κοινός παρονομαστής ε, στα πρότυπα ασφάλειας και σε όλα τα θέματα ρυθμιστικής ε, συνεργασίας ε, διακυβεύεται, αλλά εδώ μιλάμε για μείωση των προτύπων ε, σε, των προτύπων σε πολλούς τομείς οικονομίας και αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλω να υπενθυμίσω ότι οι ευρωπαϊκές συνθήκες τονίζουν την συμπεριλαμβάνουν την αρχή της πρόληψης, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Για την νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Κύριος Καστάλντο. <laughs> για λιγότερο. Πρόεδρε, όπως μου δείτε το χρόνο θα μιλήσω. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Καταλαβαίνω τις απαιτήσει του για ένα σύντομο κείμενο και εκτιμώ της προπαθίας του. Όμως μιλάμε για μια θεμελιώδη συμφωνία εδώ που ίσως να μην έχει προηγούμενο στην ιστορία των διμερών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ δυστυχώς ε, για νιωστή φορά θα πρέπει να εκφράσω πολύ μεγάλες αμφιβολίες και κριτικές γιατί εμείς την TTP τη θεωρούμε ότι εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα και μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές και όχι τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το κοκαλιά της χώρας μου αλλά και πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έλεγε ο συγητής ότι υπάρχει φιλοδοξία να δοθεί και μια πολιτική διάσταση. Όμως ακριβώς γι' αυτό κατά την απόψή μου πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να δούμε και το θέμα αυτό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις προβληματικές που τέθηκαν στο παρελθόν, όπως ε, παραδείγματος χάρη τα βασανιστήρια από το CIA, e, αλλά αναφέρομαι και στο θέμα της θανατικής ποινής. Όπως ε, ξέρετε, το απορρίπτουν αυτό τα κρατήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δυστυχώς ε, εφαρμόζονται ακόμη σε διάφορες πολιτείες ε, στην Αμερική σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές πηγές. Ε, παρά την διαφοροποίηση στις ε, πηγές, εμείς δεν πιστεύουμε ότι το σχιστολιθικό αέριο θα μπορούσε να αποτελεί μια καλή εναλλακτική λαμβάνοντας υπόψη και την τιμή αλλά και την ε, προβληματική σε περιβαλλοντικό επίπεδο, τις συνέπειες από την εξορυξή του δηλαδή στο περιβάλλον. Επίσης, θα θέλαμε να αναφέρεται και η ρήτρα ESDS, επίλυση διαφορών κράτους επενδυτή και η επιπτώση του όχι μόνο σε νομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο θα αντικατοπτρίζονταν ε, αναπόφευκτα και στις ε, σχέσεις ισχύω μεταξύ κρατών και μεγάλων ομάδων συμφερόντων. Και τέλος, θα θέλαμε αυτή η Κομισιόν να εξέφραζε την αναγκαιότητα ε, να μην μειώνουμε τα πρότυπα προστασίας του καταναλωτή και προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν στα κράτη-μέλη μας. Και κλείνω για τη διαφάνεια Σίγουρα εγώ θα ανέπτυσα το σημείο 6 και θα ζητούσα να ληφθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις στο θέμα της διαφάνειας και να μπορεί να συμμετάσχει και η κοινωνία των πολιτών και οι πολίτες. Είναι μια συμφωνία που θα έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή τους. Ε, δεν είναι δυνατόν να μην έχουν το δικαίωμα να σχηματίσουν μια άποψη πριν να υιοθετηθεί και πριν να είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Καστάλντο, ο κύριος Πρέντα. Ναι, πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Θέλω να υπερασπίσω ξενόματο ε, του ΕΛ και το όραμα που παρουσίασε ε, τη σκεπτικό του κυρίου Μιλανμόν. Ε, αυτές οι διαπραγματεύσεις θα έχουν θετικό αντίκτυπο και κατόπιν, σε αντίθεση με ό,τι είπαν οι συνάδελφοι, οι Σοσιαλιστή συνάδελφος και ο Κομμουνιστή συνάδελφος, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει διαφάνεια και δεν πρέπει να μπερδεύουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, με ένα τηλεοπτικό διάλογο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο εδώ και θα πρέπει να δεκτούμε τα όρια αυτά. Και νομίζω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε εδώ σε αυτή τη γνωμοδότηση στην πτυχή που έχει να κάνει με τις εξωτερικές υποθέσεις ε, και όχι να αναφερθούμε και σε θέματα που άπτονται των άλλων επιτροπών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρέντα. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδους εισηγητές για την κατάρτιση αυτού του εξαιρετικά δύσκολου εγγράφου. Στη σημερινή κατάσταση βλέπουμε μία μετατόπιση δυνάμεων και πρέπει υπό αυτό το φως να εξετάσουμε αυτή την εμπορική ε, διαπραγμάτευση και συμφωνία. Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και πολιτικά. Και για τη χώρα μου, αλλά και για πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ε, θα είναι εξαιρετικά ωφέλιμη αυτή η συμφωνία, γιατί θα προαγάγει περαιτέρω την ασφάλεια και θα αποσοβήσει τον κίνδυνο πολέμου. Δεν μπορούμε να ζούμε τη ζωή μας και να ελπίζουμε μόνο ότι αυτό θα συνεχιστεί για πάντα. Αντιμετωπίζουμε επιθέσεις από τα έξω και αν συνεχιστεί αυτό θα αλλάξουν τα πάντα. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι στο μέλλον αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ένας τρόπος να προχωρήσουμε και σε πολιτική συμφωνία κατανοούμε τις πολιτικές δυσκολίες, το, μέγε, το μέγεθος αυτής της ε, διαπραγμάτευσης. Ελπίζω όμως ε, σε μερικά χρόνια να καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη συμφωνία και να βελτιώσουμε και τις σχέσεις μας με μία από τις μεγαλύτερες αγορές ε, του κόσμου. Ευχαριστώ. Εν συντομία να δώσουμε το λόγο από τον, στον συνάδελφο της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, που ζήτησε το λόγο. Για δύο λεπτά μόνο, αν μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εν συντομία, να πούμε ότι ε, χαιρετίζουμε την ευκαιρία που μας δίνεται ε, να συμμετάσχουμε κι εμείς σε αυτή τη διαδικασία. Συμφωνούμε ότι δεν είναι μόνο μία απλή ε, συμφωνία ελεύθερου εμπορίου η TTIP. Είναι μια πραγματική ευκαιρία ε, για οικονομική και πολιτική μόχλευση κατά ε, αυτό το παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό που συνεχώς αλλάζει. Είναι μια πολύ ισχυρή στρατηγική συμφωνία που μπορούμε, μπορεί να ενισχύσει τις ε, σχέσεις μας με τις ΗΠΑ μαζί και με άλλους πολιτικούς και θεσμικούς εταίρους ενώ παράλληλα βέβαια θα ε, διασφαλίζουμε και το σεβασμό των ευρωπαϊκών προτύπων και αξιών. Η σύνδεση ε, με το ευρύτερο θεματολόγιο, πολυμερές θεματολόγιο, ε, είναι κάτι το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Τέλος, ε, κατά πόσο θα συμβάλλει στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι θα υπάρξει τέτοιο όφελος θα πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείριση αυτού του οικονομικού αντικτύπου και πολιτικού αντικτύπου και με τι άλλε τέτοιε χώρε όπω το Μεξικό, η Τουρκία, η ΕΦΤΑ, αλλά και με αναπτυσσόμενε ε, χώρε θα υπάρξει σημαντικό αντίκτυπο και προκειμένου να επιτύχουν οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να γίνουν με ένα πνεύμα συνεργασία. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι ε, αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν ως στόχο να αντιταχθούμε σε κάποιον συγκεκριμένο εταίρο. Για την ενέργεια συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και γι' αυτό παρεμβαίνω, όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά και για τους ε, εμπορικούς κανόνες. Όχι μόνο για τις εξαγωγές δηλαδή, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τους κανόνες ε, στο εμπόριο ενέργειας, γιατί αυτό θα επηρεάσει και την ασφάλεια. Ευχαριστώ που ήσασταν ε, τόσο σύντομο. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Μιλάν Μόν για να κλείσει η συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε για να δούμε αν μπορώ να πατήσω σύντομα στις παρατηρήσεις που έγιναν και σας ευχαριστώ για όλες. Ε, σύντομα, ελπίζω να μπορέσω να πω και σε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ κύριε Παρνιό, γιατί και εσείς επικεντρώνεστε στις εξωτερικές πτυχές. Και εσείς λέω ασχολείστε με τις πτυχές που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική. Ε, λέτε ότι απουσιάζει αναφορά στη ρήτρα ISDS για την επίλυση διαφορών. Η ίδια η έκθεση του κ. Λάγκη αφαιρώνει πάνω από τέσσερι παραγράφους αυτό. Το δεύτερο, οι ξένες επενδύσεις και επιχειρήσεις δεν είναι δική μας αρμοδιότητα της ΑΦΕΤ, αλλά είναι της ΣΥΝΤΑ. Και επιπλέον και η ΕΚΟΝ, η Οικονομική Επιτροπή, έχει αφαιρώσει πάνω από μία παράγραφο στην προστασία των επενδύσεων και στο ISDS. Ε, και απαντώ και στον κύριο Μελανσόν. Ε, θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται η διευθέτηση. Ε, η διατησία είναι το περασμένο αιώνα. Ήταν μια διατησία μεταξύ κρατών και αυτό θα ήτανε δικό μας θέμα. Η διαμεσολάβηση, η ε, δικαιοδοσία, τα, τα διεθνή δικαστήρια. Αυτό είναι κλασική ε, περίπτωση διαφορών μεταξύ κρατών. Εδώ πρόκειται για μια διαφορά μεταξύ κράτους και επενδυτή. Αυτό είναι το ISDS. Και εγώ υποστηρίζω κύριε Μελανσόν, δεν ξέρω, δεν το συμμερίζετε δικαίωμά σας. Δεν είναι τόσο θέμα διεθνού δικαίου αυτό ε, ε, και, αλλά τη ΣΥΝΤΑ, γιατί έχουμε κατανομή αρμοδιοτήτων. Εδώ δεν πρόκειται λοιπόν για συμφέροντα διακρατικά. Ε, διεθνούς δημοσίου δικαίου, αλλά είναι ο τρόπος επίλυσης διαφορών μεταξύ εταιριών. Και θέλω να πω και στον κύριο Μελανσόν και ίσως και στον κύριο Πάρνιο μπορεί να τον ενδιαφέρει. Από το 1960, 50 χρόνια τώρα, έχουμε μηχανισμούς. Δεν αλλάζουμε τίποτα, κάνουμε καμιά επανάσταση διεθνώς το 2015 ξαφνικά. 3.000 τόσες είναι οι συμφωνίες παγκοσμίω για την προστασία επενδύσεων και πολλές έχουν τέτοιους μηχανισμούς και στις ευρωπαϊκές χώρες παρακαλώ μεταξύ μας και με άλλες χώρες τρίτες. Και έχουν εκεί μηχανισμούς επίλυσης διαφοράς, πολλές συμφωνίες. Από το 2008 μέχρι το 2012, από τις 200 τόσες ε, διενέξεις που υπήρχαν μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων, 100 τόσες ε, αφορούν ευρωπαϊκές εταιρείες. Σιγά την επανάσταση. Πολλές λοιπόν ευρωπαϊκές εταιρείες είναι που προσφεύγουν. Αυτό το θέμα του ISDS θα πρέπει λίγο να ε, το αποδραματοποιήσουμε. Και να πω και στον κύριο Παρνιό. Ε, Αναφέρομαι σε αυτό, γιατί φαίνεται ότι είναι συναντήληψη διαφόρων πτέρυγων. Ε, θα πρέπει να αφαιρέσουμε λίγο τη συναισθηματική φόρτιση και να το δούμε γενικότερα, πιο ε, ισορροπημένη. Και είναι πολύ ισορροπημένη επίσης και η εντολή που έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αν είμαι εγώ αισιόδοξο για το μέλλον ε, της ε, οικονομίας. Εσείς λέτε, λέτε είστε απεσιόδοξο, κύριε Παρνιό. Υπάρχουν πολλές ε, μελέτες. Εγώ θεωρώ ότι ο πλούτος παράγεται από το εμπόριο. Και δεν είμαστε οικονομίες ε, για την επιβίωση σε μικρή ε, κλίμακα. Ε, είμαστε ανοιχτέ οικονομίε διεθνεί και δεν θα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Θα ανοίξουν λέτε οικονομίες. Μα είναι αρκετά ανοιχτέ. Εγώ δεν έχω αυτή την αρνητική αντίληψη και την απεσιόδοξη για το αποτέλεσμα. Είναι ένα κύριο που έχει γράψει για αυτά που λέγεται Καπάλτο, μια διατριβή έχει κάνει, με πάρα πολύ αρνητική αντίληψη, αλλά η συντριπτική πλειονότητα των μελετών και των ε, ε, διατριβών ε, είναι διθυραμβικές. Ε, για τη διαφάνεια έχουν γίνει πολλά προγράμματα. Ήταν σοσιαλιστής ο προηγούμενος πρόεδρος της ΣΥΝΤΑ πέρσι τον Απρίλιο και είπε στην Ισπανική τηλεόραση ότι ήταν τρομερά διαφανής η συζήτηση και διαπραγμάτευση. Δεν τα λέω αυτά εγώ, ο κύριος Μορέιρα το έλεγε και η Επιτροπή Γιούγκερ και ο Γιούγκερ ο ίδιος έχει κάνει περισσότερα βήματα για τη διαφάνεια. Και υπάρχει και κόσμος που δεν θεωρεί ότι είναι τόσο σκοταδιστικά όλα αυτά. Ε, θέλω να ευχαριστήσω ε, τον επόμενο συνάδελφο. Συμφωνώ. Αν προχωρήσει τι TTIP ε, κύριε Τάνοκ, είναι εγγύηση για να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, ε, πρόεδρε μην ανησυχείτε, τρέχω τρέχω. Για την κυρία Σχάκε, θέλω να την ευχαριστήσω, αλλά έχει φύγει. Ε, κύριε Μέλανσόν μου, το θέμα της κατασκοπίας. Κοιτάξτε, ε, αυτό και η προστασία των δεδομένων έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, Ελευθεριών. Ξέρω ότι σε αυτό το θέμα έχουμε περάσει δύσκολους καιρούς πέρσι. Ξέρω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν καταλάβει το σφάλμα τους, βελτιώνονται. Ξέρετε ότι ο κύριος Ομπάμα τις προάλλες ε, ε ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να προστατεύσει νομικά ε, και τους Ευρωπαίους πολίτες και θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα να προσφεύγουμε στα Αμερικανικά δικαστήρια. Ε, εντάξει, υπήρξε η υπόσχεση ότι θα σταματήσουν να κατασκοπεύουν τους εταίρους και τους φίλους και τις χώρες μας και επίσης νομίζω ότι προχωράει η συμφωνία για την προστασία δεδομένων. Αυτά είναι θέματα της ΛΥΜΠΕ όπως γνωρίζετε. Αλλά συμφωνώ ότι δοκιμάστηκαν οι σχέσεις μας πέρσι με τις Ηνωμένες Πολιτείες Ε, ε, ξέρετε ότι ο, ο βασικός ε, διαπραγματευτής και όλοι είπαν ότι η προστασία των δεδομένων είναι εκτός TTIP, θα είναι σε άλλη συμφωνία. Γι' αυτό δεν θέλησα εγώ να μπω σε χωράφια ξένα. Ο έχει μπλοκαριστεί, βεβαίως. Τι να κάνουμε, έτσι έχει ζωή. Ε, ε, υπάρχουν περιφερειακοί παράγοντες που ε, διαπραγματεύονται. Λέτε ότι είναι σε παρακμή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Διαφωνώ. Και επίση διαφωνώ για αυτά που λέτε για τον ανταγωνισμό. Γιατί τα βλέπετε τόσο μαύρα. Ο ανταγωνισμό δείχνει και τι τιμέ για του ε, καταναλωτέ. Και στον κύριο Μέσεριτ θέλω να το ευχαριστήσω για τα λόγια του. Θέλω να πω ότι και αυτό είναι λιγότερο αισιόδοξο. Δεν θέλουμε να ρίξουμε πρότυπα και προδιαγραφέ σε καμία περίπτωση. Ποια είναι η γραμμή, να δούμε ποια πρότυπα είναι περιτά, υπερβολικά, επικαλύψεις για να κατεργηθούν. Για γραφειοκρατία μιλάμε. Και απαντώ και στον κύριο Καστάλτο. Δεν είναι για τις πολυεθνικές αυτό. Οι μικρομεσαίες θα ωφεληθούν. Γιατί σε αυτή την τεράστια ζούγκλα της γραφειοκρατίας και των αδειών που χρειάζεται για να μπουν στην αγορά των ΗΠΑ, χάνουν τα λεφτά τους σε ενδιάμεσους δικηγόρους και άλλους. Για τις μικρομεσαίες είναι ευεργετικό. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα διαφωνούμε. Το είπατε κι εσείς ότι έχουν τη θανατική ποινή. Και η Νότια Κορέα τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε κάνει συμφωνία με τη Νότια Κορέα. Η Ιαπωνία, η Ινδία. Διαφωνούμε. Αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά στην εξωτερική πολιτική, αλλά δεν είναι το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής ούτε της εμπορικής. Για το ISDS απάντησα. Α, κατά τα άλλα. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ωφεληθούν, γιατί υπάρχουν αμερικανικά δικαστήρια που δεν αναγνωρίζουν διεθνή δικαιοδοσία. Διαφάνεια. Είπα και προηγουμένως ε, τι φρονώ. Προχωρούμε. Κάνουμε πρόοδους. Ευχαριστώ τον κύριο Πρέντα για τη ε, καλά του λόγια. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Θα διαβάσω με μεγάλο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις και τροπολογίες σας. Και ε, κάνω και μια έκκληση. Λίγο να πειθαρχηθούμε. Μια αυτοσυγκράτηση. Δεν μπορώ να κάνω παράλληλη έκθεση ε, απέναντι στην ίντα και του κυρίου Λάγκη. Εμείς νομοδοτούμε. Ας νομοδοτήσουμε ε, βάσει των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Εξωτερικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κύριε Σιγητά, ευχαριστώ όλους σας. Διακοπή της συνεδρίασης. Ραντεβού αύριο στις 9 για τις ψηφοφορίες. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς για την υπέρβαση ωραρίου.